Dear colleagues, Αγαπητοί συνάδελφοι, μπορούμε μάλλον να ξεκινήσουμε. Έχουμε καθυστερήσει λιγάκι. Α ξεκινήσουμε με το σημείο 1 τη ημερήσια διάταξη, την έγκριση τη ημερήσια διάταξη. Πολλέ ομάδε ζήτησαν να αναβληθεί η ψηφοφορία για τα σημεία 20, 20, 21 και 22 ε, θα τα αναβάλουμε για 5η-14 Ιανουαρίου και διατηρείται η ψηφοφορία Ολομέλειας ε, για τη μικρή Ολομέλεια του Ιανουαρίου. 25 ε, Ιανουαρίου είναι η προθεσμία. Αν δεν υπάρχει αντίρρηση μπορούμε να υιοθετήσουμε τι σχέδιο μερίστη διαθέξεις με αυτή την αλλαγή. Δεν υπάρχει ένσταση, μπορούμε να συνεχίσουμε. Σημείο 2. Ανακοινώσει του Προέδρου. Στη συνάντηση έμβη του Ιανουαρίου η απογευματινή συνεδρίαση 5η 14 Ιανουαρίου ακυρώνεται και μια έκτακτη συνεδρίαση θα λάβει χώρα στο Στρασβούργο την 5η 21 Ιανουαρίου από τις 9 μέχρι τις 11.30 ώστε για να, να ψηφίσουμε μεταξύ άλλων ε, κάποιες επίπουσες ε, γνωμοδοτήσεις. Σήμερα έχουμε γερμηνία σε 21 γλώσσες και όπως συνήθω. Ε, τα έγγραφα υπάρχουν διαθέσιμα μέσω της εφαρμογής e-meeting και μεταδίδεται σε άμεση μετάδοση η συνεδρίαση επίσης και μπορούμε τώρα να περάσουμε στο επόμενο σημείο ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Επίτροπο Καρμένου Βέλα. Τον ευχαριστούμε που βρίσκεται εδώ. Επίτροπος Αρμόδιος για το περιβάλλον, την θαλάσσια πολιτική και την αλληλεία. Σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για πρώτη φορά την κυκλική οικονομία και τα σχετικά μέτρα. Και όπως συνήθως ξεκινάμε με την παρουσίαση του Επιτρόπου για 10 λεπτά, κάπου εκεί, και θα συνεχίσουμε με μια συζήτηση με τις πολιτικές ομάδες για αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα. Κύριε Επιτρόπε, ευχαριστώ πολύ Τζοβάνι, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί ευρωβουλευτές, καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία που μου δίνετε να παρουσιάσω το νέα μέτρο της Επιτροπής για την Κυκλική Οικονομία με τρόπο λίγο πιο λεπτομερή από ό,τι έχει συζητηθεί μέχρι σήμερα. Βρίσκομαι εδώ σήμερα γιατί θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι αυτό είναι το καλύτερο δυνατό πακέτο μέτρο που μπορεί να προσφέρει η Ευρώπη ε, στο σημερινό οικονομικό κλίμα. Άκουσα με ενδιαφέρον τις αντιδράσεις του Κοινοβουλίου όταν παρουσιάστηκαν οι προτάσεις από τους αντιπροέδρους ε, στις 2 Δεκεμβρίου. Πριν μπω σε λεπτομέρειες για τη δέσμευτη μέτρων, θα ήθελα να κάνω δύο γενικά σχόλια. Πρώτον, Όσον αφορά τη συνελική μορφή της δέσμης μέτρων, το, η αρχική δέσμη μέτρων ανασχεδιάστηκε διότι θεωρήθηκε το η εφαρμογή τη ήταν πολύ στενό και η νέα μα πρόταση για την κυκλική οικονομία είναι σημαντικά διευρυμένη. Θα αντιμετωπίσει πραγματικά προβλήματα όπω το σχεδιασμό των προϊόντων καθώς ε, και τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να αλλάξουμε τα πρότυπα κατανάλωσης με στόχο την πρόληψη της πατάλης πρώτα απ' όλα ε, με επανεξέταση ολόκληρου του κύκλου του οικονομικού μας μοντέλου και όχι μόνο των τελευταίων σταδίων της κατανάλωσης αποτελεί ε, την κατάληξη μιας ε, μακροχρόνιας διαδικασίας διαβουλεύσεων εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μεταξύ ενδιαφερομένων καθώς και με το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η δεσμή μέτρων θα υλοποιηθεί από ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όχι μόνο μερικές γενικές διευθύνσεις. Δεν είναι δηλαδή ε, ένα στενό πακέτο είναι μια, ένα ευρύ θεματολόγιο διαφόρων μέτρων δεσμευτικών και μη ε, και με συγκεκριμένες ε, προθεσμίες. Το δεύτερο μου σχόλιο αφορά το επίπεδο φιλοδοξίας. Γνωρίζω και μπορώ φυσικά να προβλέψω διάφορες ερωτήσεις που θα προκύψουν για αυτό το ζήτημα, το πόσο φιλόδοξοι είμαστε θα σας παρουσιάσω κάποιες λεπτομέρειες για να σας αποδείξω ότι έχουμε βελτιώσει τις προσδοκίες μας όσον αφορά τη φιλοδοξία. Αλλά πρώτα απ' όλα θέλω να τονίσω ένα πράγμα. Το πακέτο που προτείνουμε θα φέρει πραγματικά αποτελέσματα για πραγματικούς ανθρώπους στην πραγματική ζωή. Θα φέρει αποτελέσματα αυτή η πρόταση. Αυτό είναι το ισχυρό της σημείο. Αυτό αποτελεί μια πραγματική φιλοδοξία, όχι απλά καλές θετικές προβλέψεις που θεωρητικά φαίνονται ικανοποιητικές. Έχουμε λοιπόν, ε, θα έχουμε λοιπόν τα μέτρα έτοιμα μέχρι τα Χριστούγεννα. Ας δούμε τι γίνεται μέσα σε αυτά. Γνωρίζετε το γενικότερο πλαίσιο του πακέτου αυτού, της κυκλικής οικονομίας, το οποίο όμως είναι περισσότερο από απλή περιβαλλοντική αναγκαιότητα έχει και από οικονομική άποψη νόημα να αξιοποιούμε τους φυσικούς πόρους με τρόπο πιο ευφυή. Το κυκλικό μοντέλο είναι το μόνο το οποίο έχει νόημα μακροχρόνια γενικά για την ευρωπαϊκή οικονομία αλλά και για τις επιχειρήσεις πιο συγκεκριμένα. Το ζήτημα δεν είναι αν θέλουμε να εφαρμόσουμε κυκλική ανάπτυξη στην Ευρώπη. Το ζήτημα είναι πώς θα βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις, τους πολίτες και τα κράτη-μέλη για να καταλήξουν σε αυτό το αποτέλεσμα και να τους δείξουμε και το δρόμο με τον οποίο θα καταλήξουν εκεί γρήγορα. Αυτό που χρειαζόμαστε ένα φιλόδοξο και ολοκληρωμένο πλαίσιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να δώσουμε μια όθηση στην κυκλική οικονομία και να επιταχύνουμε την μετάβαση και να την κάνουμε πραγματικότητα αυτή τη μετάβαση. Το πλαίσιο αυτό έχει την εικόνα ενός σχεδίου δράσης, ε, όπως αυτό που έχουμε προτείνει, που καταδεικνύει τους τομείς που πρέπει να καλύψουμε. Και αυτά που προτείνουμε καλύπτουν ολόκληρη τη διάρκεια ζωής ε, ε, των προϊόντων καθώς και των υλικών. Ξεκινάει από το σχεδιασμό ενός προϊόντος μέχρι τις διαδικασίες παραγωγής, ε, μέσω καλύτερα ενημερωμένων επιλογών, ε, καλύτερης κατανάλωσης, ε, αποτελεσματικής διαχείρισης των αποβλήτων και επιστρέφει στην παραγωγή. Όλες αυτές οι διαδικασίες θα υποστηριχθούν από χρηματοδοτικά μέσα και ταμεία. Ο σχεδιασμός είναι κεντρική σημασία για τις οικονομίες μας. Όλα ξεκινούν από το τραπέζι του σχεδιασμού και εμείς δεσμευόμαστε ότι τα προϊόντα θα βοηθήσουμε να γίνουν ευκολότερα στην επισκευή, στην αναβάθμιση, στην αποσυναρμολόγηση και στην ανακύκλωση μέσω του δικού μας υπάρχοντος πλαισίου για τον οικολογικό σχεδιασμό. Εμείς θα ξεκινήσουμε προτείνοντας κριτήρια για τις ηλεκτρονικές οθόνες. Ο σχεδιασμός ε, και ότι οι αλλαγές γίνουν σε αυτόν μπορούν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις ε, και πολύ συχνά τέτοιες αλλαγές μπορούν να γίνουν χωρίς επιπλέον κόστος. Ε, η ιδέα της κυκλικής οικονομίας χαίρει ευρείας υποστήριξη. Ε, εμείς θα παρέχουμε κάποια εργαλεία ώστε να βοηθήσουμε να ενημερώνουμε τους πολίτες για να κάνουν επιλογές γνωρίζοντας τι κάνουν. Αντιλαμβανόμαστε ότι χρειάζεται καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών. Είναι κάτι που επιθυμούν και οι ίδιοι και χρειάζονται ε, προϊόντα τα οποία θα είναι πιο επισκευάσιμα, θα διαρκούν περισσότερο και αυτό θα είναι καλύτερο όχι μόνο για τους καταναλωτές αλλά και για το περιβάλλον. Γι' αυτό το λόγο η Κομισιόν αναθεωρεί ήδη την ενεργειακή επισήμανση και εξετάζει το ενδεχόμενο συμπεριλήψη πληροφοριών που αφορούν τη βιωσιμότητα στις ε, υποχρεωτικές ε, επισημάνσεις ενέργειας. Θα είναι σημαντικές όμως και οι προαιρετικές ε, επισημάνσεις και ετικέτες όπως ε, η οικολογική ετικέτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θα αποτελέσει όλο και μεγαλύτερη σημασία για αυτό το σκοπό. Επίσης η Κομισιόν εξετάζει τη μεθοδολογία του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, κάτι που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον για καλύτερη μέτρηση και ενημέρωση όσον αφορά την περιβαλλοντική απόδοση των προϊόντων και των οργανισμών. Επίσης σκοπεύουμε να καταπολεμήσουμε τις, τους παραπλανητικούς ισχυρισμούς και να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να τηρούνται πλήρως τα υπάρχοντα πρότυπα. Εγώ είμαι ιδιαίτερα ενθουσιασμένος ε, με τη δυνατότητα που θα υπάρξει για κάποια ε, έρευνα της επιλογής ε, της τεχνητής γύρανσης, planned obsolescence όπως λέμε σήμερα, ώστε να μπορέσουμε να προσδιορίσουμε τέτοιες πρακτικές μέσα με τους ενδιαφερομένους. Οι δημόσιες αρχές ε, είναι ένας από τους μεγαλύτερους καταναλωτές ε, στην Ευρώπη. Οι δημόσιες προμήθειες αντιστοιχούν περίπου στο 20% του ε- ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα αποτελέσουν λοιπόν σημαντικό μοχλό αλλαγής. Θα ενθαρρύνουμε λοιπόν τις δημόσιες αρχές να χρησιμοποιούν περισσότερα κριτήρια κυκλικής οικονομία όταν κάνουν επιλογές αγοράς. Έτσι λοιπόν θα αναθεωρήσουμε τα κριτήρια για πράσινες δημόσιες προμήθειες και η Κομισιόν θα ε, δίνει πρώτη το παράδειγμα. Όταν ε, οι αντιπροέδροι παρουσίασαν τις προτάσεις εδώ στις αρχές του μήνα, οι αναθεωρημένοι στόχοι αποτελέσαν το επικεντρό της προσοχής. Γνωρίζουμε όλοι ότι υπάρχει ανάγκη για αλλαγή διότι η διαχείριση των αποβλήτων ακόμα δεν πραγματοποιείται βάσει της ιεραρχίας ε, για τα απόβλητα. Βάσει τον ε, το στοιχείο που έχουμε για το 2012, μόνο το 20% των αποβλήτων ανακυκλώνεται ε, αποτελεσματικά, ενώ ένα 37% απλά απορρίπτεται. Αυτό σημαίνει ότι χάνουμε πολύτιμους πόρους ε, ασκώντας περισσότερη πίεση στο περιβάλλον και χάνοντας σημαντικές επιχειρησιακές ευκαιρίες. Εμείς προτείνουμε να αντιστρέψουμε την κατάσταση αυτή μέσω ενός ε, σταθερού και σαφούς ε, πλαισίου πολιτικής ώστε να ενθαρρύνουμε το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα να αναπτύξουν μακροχρόνιες επενδυτικές στρατηγικές. Αλλάζουμε την επίκεντρο της προσοχής μας προς την πρόληψη των αποβλήτων, την επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων και την ανακύκλωση. Και θέλουμε να εξαλείψουμε σταδιακά του σχήτα και να αποφύγουμε την υπερφόρτωση των διαδικασιών ε, βιολογικού μηχανικού καθαρισμού και αποτέφρωσης. Σκόπος είναι να τα καταφέρουμε όλα αυτά με δεσμευτικούς μακροχρόνιους και μεσο, ε, μακροπρόθεσμους μεσοπρόθεσμους στόχους για την ανακύκλωση και μακροπρόθεσμους στόχους για σημαντική μείωση των χήτα για τα δημοτικά απόβλητα. Υπάρχει μια πολύ σημαντική ρήτρα αναθεωρήσεις που δεσμεύει την Κομισιόν να επανεξετάσει το πεδίο εφαρμογή ε, με ενδεχομένω την εφαρμογή υψηλότερων στόχων μέχρι το 2025. Επαναλαμβάνω, ο νέο στόχο για του ΧΙΤΑ είναι δεσμευτικό. Αυτό σημαίνει ότι μόνο το 10% των δημοτικών αποβλήτων μπορούν να απορρίπτονται σε ΧΙΤΑ μέχρι το 2030. Αυτό αποτελεί σημαντικό βήμα ε, προ τα εμπρό ε, από τους απλά θεωρητικούς στόχους που είχαμε στην προηγούμενη πρόταση. Δεν θα υπάρχει πλέον δυνατότητα ε, ύπαρξη διαφορετικών χήτα για ε, τα συλλεκθέντα απόβλητα. Αυτό είναι σημαντική πρόοδος. Επίσης και κάποια άλλα σημεία που θα βελτιωθούν θα είναι τα στατιστικά στοιχεία της ανακύκλωσης ώστε να υπάρχει πραγματικός ε, ε, ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού, ακριβή δεδομένα και ακριβείς εκθέσεις διατάξεις για την πρόθεση της χρήση των οικονομικών μέσων για καλύτερη διαχείριση των αποβλήτων και υποχρέωση ε, λήψης ε, μέτρων πρόληψης αποβλήτων για να αποφευχθούν ε, τα απόβλητα κουζίνα και να περικοπούν όλα τα απόβλητα από οικοδομές ε, και κατεδαφίσεις και από διαδικασίες εξόρυξης. Θα υπάρξει μια ενθάρρυνση επανάχρηση των προϊόντων πλωστοϊφαντουργία και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, ελάχιστε απαιτήσει για τη βελτίωση του σχεδιασμού και της λειτουργίας ε, σχεδίων ε, διευρυμένης ευθύνης παραγωγών, επέκταση της υπάρχουσας ε, υποχρέωσης για τα βιολογικά απόβλητα και διόρθωση του πλαισίου για τα βιολογικά προϊόντα και τον αποχαρακτηρισμό των αποβλήτων και ε, ένα πιο ελαφρύ πρόγραμμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τώρα θέλω να εστιαστώ σε συγκεκριμένους τομείς που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες προκλήσεις οι οποίοι πρέπει να αντιμετωπιστούν στοχευμένα ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των διαφόρων φάσεων του κύκλου θα λαμβάνονται υπόψη σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας. Να ξεκινήσω λοιπόν με τα απόβλητα κουζίνας. Ξέρω ότι όλοι ανησυχούμε όσον αφορά τα απόβλητα κουζίνας, τα απόβλητα διατροφής. Είναι οικονομικά, κοινωνικά και ηθικά απαράδεκτο τόσα πολλά τρόφιμα να σπαταλώνται. Περίπου το 30% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πράγματι σιγά σιγά η κοινή γνώμη αλλάζει, όπως είδαμε το Σεπτέμβριο όταν τα Ηνωμένα Έθνη υιοθέτησαν το στόχο ε, για ε, επίτευξη μισών, 50%, ε, μείωση κατά 50% των αποβλήτων κατά κεφαλήν. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη έχουν δεσμευτεί για την επίτευξη αυτού του στόχου. Ο στόχος αυτός λοιπόν είναι τώρα δικό μα στόχο. Οι δικές μα προτάσει εξετάζουν το τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στου τομεί όπου έχει αρμοδιότητα, συμπεριλαμβανομένων των ημερομιών λήξης που πολύ συχνά αποτελούν το αντικείμενο παρανόηση μεταξύ των καταναλωτών. Επίσης κάνουμε έκκληση στα κράτη-μέλη να δράσουν για την αντιμετώπιση των αποβλήτων κουζίνα σε όλα τα στάδια όπου έχουν αρμοδιότητα από την παραγωγή μέχρι την κατασκευή, μέχρι την μεταπίεση, από τη λιανική πώληση μέχρι τα εστιατόρια, ακόμη και μέσα στα νοικοκυριά. Εμεί θα συνεργαστούμε με τα κράτη-μέλη και με του ενδιαφορομένου σε ολόκληρη την αλυσίδα ε, φαγητού, τροφίμων, σε μια, με μια αφιερωμένη ειδική πλατφόρμα που θα μας βοηθήσει για να επιτύχουμε αυτό το στόχο. Πρότασή είναι να αναπτύξουμε μια αξιόπιστη μέθοδο ποσοτικού προσδιορισμού και κατανόησης των αποβλήτων τροφίμων. Έτσι θα μπορέσουμε να μετρήσουμε την πρόοδο σε σχέση με τους στόχους ώστε να επιτύχουμε μείωση των αποβλήτων τροφίμων στο μισό. Ένας άλλος τομέας με μεγάλες προκλήσεις είναι τα πλαστικά. Εδώ χρειαζόμαστε κατεπίγουσα δράση. Ενώ η χρήση των πλαστικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξάνεται ε, σταθερά. Λιγότερο από το 25% των ε, συλλεκτών των αποβλήτων πλαστικών ανακυκλώνεται και περίπου το 50% καταλήγει σε χύτα. Όπως ε, ανέφερα προηγουμένως, η νομοθετική πρόταση θα αυξήσει τους υπάρχοντες στόχους ανακύκλωσης για τα δημοτικά απόβλητα και για απόβλητα πλαστικών συσκευασιών μαζί με τα μέτρα μείωσης των ΧΙΤΑ και βελτίωσης ε, του διαχωρισμού της συλλογή ε, θα καλυφθεί η υποχρέωση αύξηση των ποσοστών ανακύκλωση για τα πλαστικά. Αλλά οι καλές προθέσεις δεν αρκούν. Χρειάζεται να κάνουμε περισσότερα για να δούμε αποτελέσματα. Το σχέδιο δράση, θα βοηθήσει μέσω μέτρων για την ενίσχυση του οικολογικού σχεδιασμού και για την εγκαθίδρυση πιο αυστηρών προτύπων ποιότητα για, τα για τι δευτερεύουσε πρωτεσίλε συμπεριλαμβανομένων των πλαστικών. Στο πλαίσιο μια συγκεκριμένη προσέγγιση για τα πλαστικά, η Κομισιόν θα προετοιμάσει μια συγκεκριμένη στρατηγική για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούν τα πλαστικά σε ολόκληρη την αλυσίδα αξία. Μέσω αυτή τη στρατηγική θα εξεταστούν οι, πιθανές, οι πιθανοί προβληματικοί τομεί, όπω η παρουσία χημικών που προκαλούν ανησυχίε και θα καλυφθεί ολόκληρη η διάρκεια ζωής του πλαστικού ώστε να διασφαλιστεί μια πραγματικά κυκλική προσέγγιση. Θα υπάρξει συμπερίμνα ώστε τα καινοτόμα ανταγωνιστικά ανακυκλώσιμα και ασφαλή πλαστικά του μέλλοντος να προέλθουν πρώτα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ ερχόμαστε τώρα στα θαλάσσια απόβλητα. Πολύ, υπερβολικά μεγάλη ποσότητα πλαστικών καταλήγει δυστυχώς στις θάλασσες. Έχουμε να ασχοληθούμε λοιπόν και με αυτό το ζήτημα για διάφορους λόγους ε, συμπεριλαμβανομένη της νέας διεθνούς δέσμευσης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για στο πλαίσιο των στόχων αηφόρων ανάπτυξης για σημαντική μείωση των θαλασσιών αποβλήτων μέχρι το 2015. Η δράση μας για τις πλαστικές σακούλες αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα προς τα μπρος και οι προσπάθειες ε, για την μείωση των χήτα και την αύξηση της ανακύκλωσης θα μας βοηθήσουν ακόμη περισσότερο. Η Κομισιόν θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα με συγκεκριμένε δράσει για τα θαλάσσια απόβλητα στη στρατηγική τη για τα πλαστικά στο πλαίσιο τη κυκλική οικονομία. Έχουν ήδη ξεκινήσει εργασίε για να επιτύχουμε τον φιλόδοξο στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση των θαλασσιών αποβλήτων κατά 30% μέχρι το 2020. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να κλείσω με λίγα λόγια ε, για κάτι που ανέφερα προηγουμένως ως ε, ε, υποστηρικτικό πλαίσιο. Έχουμε μία σειρά μέτρων υποστήριξης στο νου μας, όπως το Ορίζοντα 2020, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το ΕΦΣΙ και τα διαρθρωτικά ταμεία. Στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020, για παράδειγμα, μια σημαντική πρωτοβουλία ύψους 650 εκατομμύριων ευρώ έχει ξεκινήσει για τη βιομηχανία 2020 στην κυκλική οικονομία. Προγράμματα περιφερειακής πολιτικής επίσης θα βοηθήσουν να πραγματοποιηθούν αλλαγές επιτόπου με υποστήριξη για επενδύσεις ε, στον διαχωρισμό των αποβλήτων κατά τη συλλογή τους και για τις υποδομές ανακύκλωσης. Μέχρι το 2020, 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν μόνο για τη διαχείριση αποβλήτων. Επίσης, ε, στέλνουμε ένα ηχηρό μήνυμα ότι τα διαρθρωτικά ταμεία θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τη χρηματοδότηση των υψηλότερων επιπέδων της ε, ιεραρχίας αποβλήτων. γεγονό που σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση απομακρύνεται σιγά σιγά από την αποτέφρωση και ταχύτητα εκτός εάν αυτό αιτιολογείται επαρκώς. Επίσης θα χρειαστούμε σημαντικές επενδύσεις από τον ιδιωτικό τομέα για αυτές τις νέες ευκαιρίες. Έτσι, η Κομισιόν θα ενθαρρύνει αιτήσει προ το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, οι οποίε θα βοηθήσουν να βρεθούν ιδιωτικά κονδύλια χρηματοδότηση. Πριν δύο εβδομάδε, εγώ παρουσίασα τη δέσμη μέτρων στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η απάντησή του ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντική. Ο πρόεδρος Χόιερ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ενημέρωσε ότι ο οργανισμός του έχει ήδη συγχρηματοδοτήσει προγράμματα κυκλικής οικονομίας αξίας περίπου 15 δισεκατομμύριων ευρώ ε, τα τελευταία δεκαετία. Η τράπεζα αυτή τη στιγμή αναθεωρεί τις δραστηριότητές της ώστε να βρει του καλύτερου δυνατού τρόπου για την επιτάχυνση τη μετάβαση προ μια κυκλική οικονομία. Την περασμένη εβδομάδα η τράπεζα συμφώνησε να επεκτείνει τα κριτήρια επιλεξιμότητας για την Innofin, ένα πρόγραμμα ύψους 24 δισεκατομμύρων ευρώ για την προσέλκυση προγραμμάτων κυκλικής οικονομίας. Αυτά είναι καταπληκτικά νέα για τα προγράμματα όπου το στοιχείο του αντιληπτού κινδύνου είναι λίγο υψηλότερο. Έχουμε εδώ λοιπόν έναν πολύ ισχυρό σύμμαχο, το μεγαλύτερο δανειοδότη ε, πολύπλευρο διαδημιοδότη του κόσμου που συνεργάζεται για λύσεις ε, που θα έχουν εφαρμογή στον πραγματικό κόσμο και θα βοηθήσουν στο να επιταχυνθεί η αλλαγή, η μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία. Αγαπητοί συνάδελφοι, να σας ευχαριστήσω για το ενδιαφέρον που έχετε δείξει για αυτό το θέμα και ελπίζω να έχετε πιστεί ότι το σχέδιο δράσης και οι προτάσεις θα παράσχουν φυκτά, ε, φιλόδοξα και μακροχρόνια αποτελέσματα. Ακόμη πιο σημαντικό θέλω να επαναλάβω ότι αυτές οι προτάσεις είναι ρεαλιστικές. Έχουν μελετηθεί μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια ώστε να ανταποκρίνεται στην οικονομική πραγματικότητα του καιρού μας. Αλλά προς το παρόν δεν είναι παραπροτάσεις. Το τελικό αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό και από τη δική σας συμμετοχή. Θέλω, δράτω λοιπόν τη ευκαιρία για να ζητήσω τη συνεχή σας συνεργασία και δέσμευση στους πλαίσιο διαλόγων με άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές, με κράτη-μέλη, με τις περιφέρειες, με τους δήμους και με όλους τους ενδιαφερομένους. Επίσης θα ήθελα εδώ να επισημάνω ότι όταν παρουσίασα τη δέσμευτη μέτρων στο Συμβουλίο τα κράτη-μέλη την υποδεχτήκαν με πολύ θετικά σχόλια. Υπολογίζω λοιπόν σε όλους τους ενδιαφερομένους και ειδικότερα σε εσά ώστε να συνεχίσουμε το διάλογο και να διασφαλίσουμε ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες θα μπορέσουν να υποφεληθούν πλήρως από την ταχύτατη μετάβαση σε μια πραγματική ε, κυκλική οικονομία. Αυτή θα είναι η Ευρώπη του μέλλοντος, αυτή θα είναι η Ευρώπη που χρειάζεται η οικονομία μας. Σας ευχαριστώ όλους για το χρόνο σας και για την προσοχή σας. Thank ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε για την εξαιρετική σας παρουσίαση. Αρχίζουμε τώρα με τον πρώτο γύρο μιλητών. Οι εκπρόσωποι των πολιτικών ομάδων. Κάλεν Φλόρενς πρώτα. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε που είστε εδώ και μας παρουσιάζετε για άλλη μια φορά την έκθεσή σας. Δεν είστε από εκείνου που πριν από ένα χρόνο απέσυραν την ε, έκθεση αυτή εκ μέρους της Επιτροπής με την ε, αμφίβολη διατύπωση ότι θέλουν μια πιο φιλόδοξη έκθεση, ε, πρόταση. Την ε, διατυπώνετε λοιπόν εσείς τώρα, σήμερα. Πρέπει να είναι λοιπόν πιο φιλόδοξα αυτά τα οποία μας ε, είχε υποσχεθεί ο Αντιπρόεδρος, έτσι μας το είχε υποσχεθεί, αλλά δεν τη βλέπω να είναι πιο φιλόδοξη η πρόταση. Λέτε ότι είναι ευρύτερη. Ναι, ευρύτερη διατύπωσή της. Αλλά έχει και πιο πολλά κενά με το να έχει πιο ευρεία διατύπωση και φάσμα θεμάτων. Και αυτές οι οικολογικές και οικονομικές ε, συνέπειες της ε, κυκλικής ε, οικονομίας δεν μου φαίνονται πολύ σαφείς. Και ξέρετε ότι όλος ο κλάδος της παραγωγής στην Ευρώπη ανησυχεί ότι μπορεί αυτή η κυκλική οικονομία να οδηγήσει σε πολύ περισσότερες δαπάνες και κόστες με οικολογική και οικονομική δραστηριοποίηση. Πρέπει να έχουμε ή μη τι άλλο πιο πολλές οικονομίες. Δεν μπορούμε να έχουμε περισσότερο κόστος. Αυτό πρέπει να διευκρινιστεί. Επίσης, όλο μιλάμε για αυτό το παλιό ποδήλατο που θα πάμε στην ανακύκλωση, που όμως μπορεί τελικά να θεωρούμε ότι έχει ξεκινήσει από ένα ορυχείο μεταλλευμάτων, από ένα μεταλλορυχείο σε κάποιον ξένο πλανήτη σχεδόν. Φαίνεται συνέχεια σαν να πρόκειται για μια νέα οδηγία για απόβλητα, αλλά νομίζω θα πρέπει να κοιτάξουμε τον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη αντιμετωπίζει τα απόβλητα που είναι πολύ καλά οργανωμένος εάν δούμε τις ε, συνθήκες στα πρώτα κράτη-μέλη, δεν χρειάζεται να πάμε στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, εκεί πρέπει να κοιτάξουμε πού βρίσκονται τα προβλήματα. Και σε σχέση με την απαγόρευση της χρήσης της λέξης χωματερή, κάθε φορά που γίνεται λόγος για απαγόρευση χωματερών, ακόμα και στη Γερμανία, οι πολιτικοί αρχίζουν να ανησυχούν πολύ καταργούνται λένε οι χωματερές, δεν θα υπάρχουν και χωματερές. Όχι, είναι λάθος αυτό. Απλώς στη χωματερή δεν πρέπει να φτάνει τίποτα που να μην έχει περάσει από τη σχετική διαλογή πια. Γι' αυτό λοιπόν αυτό πρέπει να διατυπωθεί και να εξηγηθεί καλύτερα. Στο πρόγραμμα δράσης. Νομίζω ότι θα πρέπει να βρείτε πιο εφάνταστες λύσεις. Ναι και είναι και η περίοδος των Χριστουγέννων και ζούμε λίγο στον κόσμο της φαντασίας, θα σας παρακαλούσα να διατυπώσετε το κείμενο έτσι ώστε να γίνει ένα συνολικό έγγραφο. Έγγραφο συνολικό, διότι διαφορετικά κύριε Επίτροπε, διερωτώ με, πόθεν αντλείτε το θάρρος να έρχεστε εδώ να μας παρουσιάσετε αυτά τα πράγματα όταν γνωρίζουμε ότι από αυτά που ήδη υπάρχουν τώρα από τις οδηγίες για τα απόβλητα δεν έχουν αντιμετωπιστεί. Και πάλι μιλάω για τη δική μου την πατρίδα. Ναι κύριε Πρόεδρε, ξέρω. Παρακαλώ όμως να δείξετε μια ανοχή. Τόσες οδηγίες που έχουν διατυπωθεί, εγκριθεί, περάσει σε εθνικό δίκαιο και δεν έχουν εφαρμοστεί από τις περιφέρειες, γιατί εκεί βρίσκεται η αδυναμία και εκεί εσείς κύριε Επίτροπε πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη έμφαση. Αλλά βέβαια υπάρχουν όλοι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται στο επιτελείο σας, οι οποίοι θα πρέπει να τηρήσουν τελικά τις οδηγίες αυτές και την νομοθεσία. Ευχαριστώ κυρία Μποναφέ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε για αυτή την πολύ λεπτομερική ακριβή παρουσίαση αυτού του πολύπλοκου ε, τομέα που αφορά πολλά θέματα. Να σε ευχαριστήσω όμως επειδή και εσείς και η Κομισιόν κρατήσατε το λόγο σας. Είπατε ότι θα αποσύρατε την παλιότερη οδηγία και ότι η ναι, νέα θα ήταν έτοιμη πριν το τέλος του έτους. Οπότε βρισκόμαστε εδώ έχοντας την μπροστά μα Μπροστά Παρ' όλα αυτά εγώ παρατηρώ ότι εργάστηκαν πολλέ ε, γενικέ διευθύνσει για αυτή τη δέσμη μέτρα. Αυτό είναι, μέτρο. είναι πολύ θετικό αυτό. Αυτό σημαίνει ότι κανένα δεν διέφυγε από την προσέγγιση που χαρακτηρίζει την ε, κυκλική οικονομία. Δηλαδή μια ολιστική προσέγγιση που χαράσει έναν κύκλο τον οποίο κλείνει όπως έχει υποθεί επανειλημμένος. Ίσως πράγματι η πρώτη οδηγία να ε, μην ήταν απολύτω ισορροπημένη. Οπότε εδώ λαμβάνεται υπόψη και το κομμάτι της υλοποίησης. Ε, το κυριότερο όμως ε, είναι ότι αυτή η προσέγγιση της κυκλικής οικονομίας ε, δεν αποτελεί μόνο μια οικονομία για τα απόβλητα, ούτε απλά περιβαλλοντική, όπως λέτε και εσείς ο ίδιος. Είναι μια πραγματική οικονομική πολιτική που εμπλέκει όλους τους ενδιαφερομένους από τα θεσμικά όργανα, μέχρι τους καταναλωτές, μέχρι τις επιχειρήσεις, Μπορούμε δηλαδή να αναφερθούμε σε ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο και μέσω νέων βιομηχανικών μοντέλων φυσικά που λαμβάνει υπόψη φυσικά την ανταγωνιστικότητα αλλά και τις πρώτες ύλες, την περιβαλλοντική διάσταση κτλ. Είναι μια καλή ευκαιρία για να πούμε όχι μόνο ότι μέσω αυτής της κυκλικής οικονομίας θα δημιουργηθούν και νέες θέσεις εργασίας αλλά ότι θα αποτελέσει και μια ευκαιρία να ξαναδούμε τα ζητήματα τα οποία θα πρέπει να αναλύσουμε ενδεχομένω λίγο περισσότερο, διότι εντάξει τώρα δεν θέλω εγώ να κρίνω εδώ το βαθμό φιλοδοξία σα, παρότι απογοητεύτηκα λίγο από αυτή την οδηγία, όσον αφορά του στόχου βασικά, σε αυτού αναφέρομαι, αλλά πιστεύω ότι, αν μη τι άλλο, εδώ έχουμε μια ευκαιρία να δούμε τα αδύναμα σημεία. Είναι μια πρώτη ευκαιρία για να τα δούμε αυτά τα αδύναμα σημεία και εγώ θέλω να ξεκινήσω από την ιεραρχία των αποβλήτων, διότι πράγματι η πολιτική αυτή δεν αφορά μόνο τα απόβλητα, η κυκλική οικονομία αφορά τη βέλτιστη και αποτελεσματική ε, διαχείριση του ολόκληρου του κύκλου των αποβλήτων και εγώ ξεκινώ από την ιεραρχία. Εγώ ξέρετε πιστεύω στο αξίωμα ότι ο πιο αποτελεσματικό χρήσο, η πιο αποτελεσματική χρήση ενό σπόρου είναι η μη χρήση τη. Ε, αν θέλουμε να κάνουμε οικονομία στο ηλεκτρικό κλείνουμε το διακόπτη. Οπότε και για τα απορρίμματα και για τα απόβλητα όλα εξαρτώνται από τον τρόπο που εμείς παράγουμε και χρησιμοποιούμε ένα προϊόν και πώς το επαναχρησιμοποιούμε, πώ το ανακυκλώνουμε, πώ το επισκευάζουμε αυτά είναι τα νέα χαρακτηριστικά της νέας αυτής κυκλικής οικονομίας ε, και το λέω εθαρσός ε, εγώ πιστεύω ότι σε αυτά τα θέματα είναι αδύναμη αυτή η οδηγία δεν έχει συγκεκριμένους στόχους και αυτή η ιδέα ε, των καταξιοδότηση πράξεων από το 2017 και μετά είναι λίγο χαλαρό και Κάτι άλλο που απασχολεί ιδιαίτερα το Κοινοβούλιο είναι το food waste, είναι η σπατάλη τροφίμων. Δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό, αλλά είναι και θέμα ηθικής. Δεν επιτρέπεται λοιπόν να αποκλίνουμε από αυτές τις οδηγίες σε θέματα αυτά. Αλλά και όσον αφορά επίσης και την, ε, το διαχωρισμό των, της συλλογής των ε, αποβλήτων, δεν υπάρχουν αρκετές λεπτομέρειες. Χρειάζονται υποχρεωτικά μέτρα με συγκεκριμένες ε, βέβαιες προθεσμίες. Είναι αυτός ο μόνος τρόπος για να καταλήξουμε σε θετικά αποτελεσματικότητα, ε, για να ε, επιτύχουμε αποτελέσματα όσον αφορά τους σπόρους και όσον αφορά την ενέργεια. Και επίσης και οι best practices, οι βέλτιστες πρακτικές μπορούν να χρησιμοποιηθούν τώρα για τους στόχους, το ξαναείπα προηγουμένως. Εμείς θεω, δεν θεωρούμε ότι το 5% πάνω ή κάτω από το στόχο είναι το μέτρο αξιολόγησης της φιλοδοξίας αυτής της μέτρων. Ωστόσο θεωρούμε ότι όλα θα παιχτούν ε, στο γήπεδο της αξιοπιστίας. Αν θέλουμε λοιπόν να είμαστε αξιόπιστοι πρέπει να ε, βελτιώσουμε τις προσδοκίες και φυσικά ναι σίγουρα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα ρεαλιστικά στις χώρες που σήμερα αντιμετωπίζουν δυσκολίε, αλλά δεν μπορούμε εμείς να είμαστε πρώτοι που εφαρμόζουμε εξαιρέσεις όσον αφορά τις φιλοδοξίες. Για να κλείσω, ε, μας υπενθυμίσατε τις ευαισθησίες σα όσον αφορά τις προτάσεις που θα κάνει το Κοινοβούλιο. Ξέρετε, σε αυτή την οδηγία ε, πολλοί κόσμος αναμένει να σχολιάσει, πολλοί κόσμος περιμένει να τη δει στο βιομηχανικό τομέα, οπότε εμείς πρέπει να βιαστούμε εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο και να υποβάλουμε κάποιες καλές ιδέες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Δέμες Μέκερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ που ήρθατε εδώ στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Και εμείς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για τις προσπάθειές σας, για την ευρεία ενημέρωση που μας κάνατε και να ξέρετε ότι πιστεύουμε και εμείς τις ευκαιρίες που έχουμε τώρα μπροστά μας. Είναι όμως και ανάγκη η κυκλική οικονομία για το περιβάλλον, για την ευημερία μας. Με έξι μήνες καθυστέρηση δυστυχώς, κρίμα. Και για μένα παραμένει σαφές το γιατί υπάρχει αυτή η καθυστέρηση. Πρέπει να δούμε όλη την αλυσίδα η χρήση των ε, ορυκτών αυξάνει. Δεν μειώνεται με το χρόνο που περνάει, οπότε θα πρέπει να βιαστούμε περισσότερο. Πρέπει να δώσουμε τώρα δυνατότητες σε πειράματα, σε νέα μοντέλα. Το πρόγραμμα δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όμως για μένα παραμένει ασαφές όσον αφορά αυτό το σημείο το πακέτο αποδυναμώνει επίσης και κάποια σημεία. Στις 2 Δεκεμβρίου υπέβαλα διάφορες ερωτήσεις πρόεδρες στη συζήτηση που είχαμε στην ε, Ολομέλεια και ακόμα δεν έχω απαντήσεις. Πρώτον, οι διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των χωρών μελών όσον αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας που ήδη υπάρχει για τα θέματα αυτά που εξετάζουμε. Έχουμε κάποιους στόχους για το 2020 που είναι και η μεγάλη πρόκληση για όλους μας. Πώς λοιπόν θα τεθούν σε εφαρμογή τόσα ήδη προβλέπονται. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν καταρχήν πρέπει να κάνει προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση. Έπειτα, δεν πρέπει να πέφτει το επίπεδο φιλοδοξίας μας όσον αφορά το 65% ε, να πέσει το επίπεδο των ε, οικιακών αποβλήτων. Σύμφωνοι, να δούμε κατά περίπτωση, αλλά οι χώρες εκείνες που δυσκολεύονται είναι η μία κατηγορία και άλλη κατηγορία είναι εκείνες που μπορούν να κάνουν περισσότερα. Η Φλάνδρα για παράδειγμα περιοχές, περιφέρειες που χρειάζονται ενθάρρυνση, που πρέπει να έχουν κάθε ευκαιρία, να δώσουν κάθε ευκαιρία στην καινοτομία. Σε αυτά θέλουμε τη στήριξή σας. Και τρίτον, αν θέλουμε να βάλουμε τις βάσεις για μια πιο πράσινη οικονομία, τότε πρέπει να σταματήσουμε να εμποδίζουμε την ανακύκλωση κάποιων ε, προϊόντων. Τα ανακυκλώσιμα πρέπει να μπορούν να ανακυκλώνονται χωρίς περιορισμούς. Το πακέτο αναφέρεται κυρίως στα οικιακά απόβλητα. Τι θα κάνει όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα απόβλητα των επιχειρήσεων. Η Φλάνδρα έχει εμπειρίες με την ανακύκλωση και κατά προτεραιότητα προϊόντων όπως αναφέρατε εσείς. Θα πρέπει να βοηθήσουμε λοιπόν τις επιχειρήσεις αυτές που έχουν αυτή την εμπειρία. Ξέρω ότι το φλαμαδικό μοντέλο μπορεί να προσφέρει έμπνευση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όμως δεν θα πρέπει να νομίζουμε ότι ήδη έχουμε καταφέρει κάτι. Όχι, βρισκόμαστε μόνο στην αρχή. Πρέπει να ενθαρρύνουμε την καινοτομία τώρα. Είναι ζωτική σημασία λοιπόν η πρόταση που θα κάνουμε να μπορεί να αποφέρει αποτελέσματα, να είναι δηλαδή κάτι το ρεαλιστικό στην πράξη. Έχετε τη συνεργασία μας, ξέρετε ότι είμαστε φίλοι και τέροι και θέλουμε και εμείς να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να πετύχουμε. Ευχαριστούμε κύριος Γκερμπραντή τώρα. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον Επίτροπο που ήρθε. Φοβάμαι ότι όλοι συμφωνούμε για το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πυροβόλησε στα πόδια της βασιστικά όταν απέσυρε την πρότασή της πέρυσι. Ήταν λάθος. Και έχοντας δει τις νέες προτάσεις, γίνεται ακόμα πιο κατάφορο ότι έκανε λάθος πέρυσι. Φοβάμαι ότι όσοι πήραν αυτή την απόφαση για την απόσυρση πέρυσι, το κάναν για πολιτικούς λόγους ή δεν ξέρανε καλά τι κάνουν. Για να διορθωθεί τώρα το σφάλμα αυτό, η Επιτροπή υποσχέθηκε να μας έρθει με ακόμα πιο φιλόδοξες προτάσεις πριν τα τέλη της χρονιάς. Αν κοιτάξω λοιπόν το νέο πακέτο για τα πόβλητα και το πρόγραμμα δράσης, φοβάμαι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έκανε αυτό που είπε, δεν τήρησε την υπόσχεσή της για πιο φιλόδοξες προτάσεις. Κυρίως αν λάβουμε υπόψη μας το πρώτο αντιπρόεδρο της Επιτροπής, τον κύριο Τίμερμανς και όσα μας είπε και κατά την Πράσινη Εβδομάδα και κατά τη συζήτηση για την έκθεση ποιοτικά είναι στην Ολομέλεια, όντως ήταν πολύ πιστικός για το πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν τέτοιες προτάσεις και οικονομικά και περιβαλλοντικά, ότι η κυκλική οικονομία είναι ζωτική σημασίας από πολλές απόψεις και δημοσιεύτηκε και η μελέτη Μακιάνση τον Ιούνιο που επιβεβαίωνε αυτά τα λεγόμενα, ότι δηλαδή δεν πρόκειται μόνο για ένα πακέτο για το περιβάλλον, αλλά πρόκειται για κάτι πολύ περισσότερο. Πρόκειται για τη νέα οικονομική ατζέντα, τους νέους στόχους δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωραία, εγώ δεν θα μιλήσω για τα απόβλητα και το τι λέει για αυτά στην πρόταση. Γενικά μιλώντας είδε τα ίδια λίγο πολύ όπως είχαμε και πριν από ένα χρόνο, ενάμιση. εδώ και εκεί βλέπουμε λιγότερη φιλοδοξία. Αλλού πάλι είναι καλύτερα όσον αφορά τον ορισμό, την ευθύνη. Και εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορούμε να ενισχύσουμε, να αυξήσουμε τα ποσοστά εδώ και εκεί και να διορθώσουμε ε, το κακό που έχει γίνει. Θα αναφερθώ κυρίως στο πρόγραμμα δράσης, γιατί εδώ είναι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας υποσχέθηκε τα περισσότερα, που είναι η άλλη πλευρά της κυκλικής οικονομίας. Και για να είμαι ειλικρινής, στις 2 Δεκεμβρίου είπα ότι ήταν copy-paste, αντιγραφή και επικόλληση δηλαδή του χαρτιπορίας του 2011, αλλά είναι ακόμα χειρότερα. Είναι πιο αποδεινωμένο το πρόγραμμα αυτοδράσης από εκείνο του 2011, πριν από τέσσερα χρόνια δηλαδή. Συνεπώς εδώ δεν μιλάμε για μια καθυστέρηση ένα-δύο χρόνια. Πριν από τέσσερα χρόνια είχαμε το προηγούμενο με πολύ συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα φιλόδοξο για τα επόμενα βήματα. Θα σας δώσω κάποια παραδείγματα για τις διαφορές που διαπιστώνουμε ανάμεσα στο χάρτη πορείας του 2011 και τις μερινές προτάσεις. Όσον αφορά τον οικολογικό σχεδιασμό, έλεγε το 2011 ότι θα πρέπει να υπάρξουν προδιαγραφές για να ενισχυθούν ε, προϊόντα τα οποία είναι πιο αποδοτικά. Το πρόγραμμα δράσης του 2015 μιλάει για ένα σχέδιο ομάδα εργασίας για οικολογικό σχεδιασμό το 2017 που θα δει πώς θα τεθούν αυτά σε εφαρμογή. Μου φαίνεται πιο αδύναμη αυτή η διατύπωση από την προηγούμενη. Έπειτα, ε, περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Πάλι η διατύπωση ήταν πιο έντονη για τις δημόσιες συμβάσεις. Το 2011 μιλούσαμε για ενίσχυση των απαιτήσεων. Ενώ εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι θα εξετάσει μόνο. Και τέτοια παραδείγματα θα μπορούσα να σας δώσω πολλά και για τα δευτερογενή υλικά. Τη δευτερογενής πρώτας Ο πρόεδρος βλέπω ότι ετοιμάζεται να με κόψει, γιατί έχω μιλήσει πολύ. Αλλά το βασικό ζήτημα είναι το εξή. Το πρόγραμμα δράσης μπορείτε να το κάνετε πιο συγκεκριμένο από ό,τι είναι τώρα. Γιατί πολλά από τα στοιχεία τα οποία ονομάζονται δράσεις θα πρέπει να υλοποιηθούν ε, σύντομα, όχι σε μερικά χρόνια. Ζητώ λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας έρθει με ένα πιο δεσμευτικό νομοθετικό κομμάτι και πιο συγκεκριμένο από αυτό που έχουμε τώρα μπροστά μας. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Κυρία Κύλωνα. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε. Μας είχαν υποσχεθεί πολλά πράγματα. Μάλιστα κάποιοι είχαν μιλήσει και για μια σχέση πάθους με το θέμα αυτό. Αλλά αυτό το πάθος δεν το βλέπουμε δεν έχουμε πολύ θερμή σχέση από ό,τι φαίνεται με την υπόθεση αυτή και το λέω εγώ, προέρχομαι και από ψυχρή ζώνη. Η κυκλική οικονομία δεν μπορεί να στηρίζεται κατά την άποψή μου στην πιο απλή λύση. Η πιο απλή λύση θα πρέπει να μας επιτρέπει να πάμε ε, πιο πέρα στους, ε, στην κατανάλωση, στον τρόπο με τον οποίο καταναλώνουμε. Δηλαδή χρησιμοποιούμε τα προϊόντα ώστε να έχουμε λιγότερες συνέπειες για το περιβάλλον, για τους πόρους, τις πρώτες ύλες, λιγότερες δαπάνες, λιγότερη κατανάλωση περιττή των ε, τροφίμων, όλα αυτά. Κατανάλωση τροφίμων και τρόπος παραγωγής τροφίμων επί παραδείγματι στα δυτικά κράτη που είναι απαράδεκτο απαράδεκτη σπατάλη με 30% των τροφίμων στα σκουπίδια το 30% αυτό που θα επέτρεπε τρεις φορές να βάλουμε ένα τέρμα στην πείνα σε όλο τον κόσμο. Στην πρόταση λοιπόν της Επιτροπής βλέπω να λείπει ένα πολύ συγκεκριμένο πράγμα στόχος για μια καλύτερη αποτελεσματικότητα στη χρήση των πόρων. Και θα έλεγα όχι καλύτερη αποτελεσματικότητα, για φρόνηση στην χρήση των πόρων. Να χρησιμοποιούμε λελογισμένα τους πόρους του πλανήτη μας για να είναι και αηφόρος η χρήση τους. Αυτή η φρόνηση μπορεί να περάσει από την κυκλική οικονομία, την χρήση των υλικών σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής, την καλύτερη χρήση της ανανεώσιμης ε, ενέργειας, αλλά αυτό δεν πρόκειται να συμβεί εάν παρακολουθούμε απλώς τις εξελίξεις άπρακτη. Πρέπει να δράσουμε. Και γι' αυτό κύριε Επίτροπε και μάλιστα πριν από τα Χριστούγεννα θα περίμενα να δω περισσότερο πάθος από πλευρά σας. Πάθος που θα μας επέτρεπε να δράσουμε. Πρέπει να σταματήσουμε να παρακολουθούμε και να παρατηρούμε τις εξελίξεις. Ο καθένας μας οφείλει και, πρέπει να και μπορεί να δράσει. Ευχαριστώ κύριος Εκχάουτ. Ευχαριστώ πρόεδρε και κύριε επίτροπε. Ευχαριστώ που μας εξηγήσατε τη δέσμη. Ελπίζω βέβαια να είναι αυτή και η τελευταία φορά που συζητούμε ε, το, τους ισχυρισμούς Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι τάχα έχει πιο φιλόδοξα σχέδια κτλ. Ε, ξέρουμε ότι κάνατε λάθος πέρσι. Και προσπαθείτε το λάθος αυτό το διορθώσετε ισχυριζόμενο τώρα προτείνετε μια πιο φιλόδοξη πρόταση. Εξκυζέ μου όμω, ε, ας σταματήσουμε τι αειδίε, να το πω και στα γαλλικά, λέει ο μιλητή. Χρειάζεται ένα πακέτο για τα απόβλητα, συγκρίσιμο σε τελευταία ανάλυση με αυτά που έχουμε, αλλά όχι αδύνα, πιο αδύναμο από αυτά που έχουμε, γιατί αυτό μα προτείνεται τώρα. Και έχουμε πολλά άλλα ζητήματα στα οποία δεν έχετε δώσει απαντήσει. Αυτή είναι η κατάσταση τώρα. Είμαστε λίγο πολύ δηλαδή και που ήμασταν πριν από 1,5 χρόνο, η διαφορά είναι ότι όλο και πιο πολλού ανθρώπου ενδιαφέρει η κυκλική οικονομία. Ε, φαίνεται ότι άρχισε λίγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βρει το δρόμο τη, ήταν κάπω έμεσο ο δρόμο μέσα στον μέσα από τον οποίο μπήκε στη συζήτηση για την κυκλική οικονομία. Τα βρήκε όμω, βρήκε το δρόμο τη εν τέλει. Σα ευχαριστούμε. Αλλά δεν χρειάζεται να αποσυρθούν οι προτάσει του τελευταίου 1,5 έτου. Έστω όμω, κάνατε αυτό, προσπαθείτε να ισχυριστείτε για να πιστέψει ο έξω κόσμο ότι είσαστε πιο φιλόδοξοι κτλ. Πολύ ωραία να σα επικροτήσουμε επικοινωνιακά τουλάχιστον για τις υπηρεσίες επιτροπής ήταν επιτυχία δεν μπορώ να πω αλλά ας κάνουμε και λίγη δουλειά τώρα για το νομοθετικό πακέτο αυτό θα το αντιμετωπίσουμε γιατί ως νομοθέτες θα κάνουμε τη δουλειά μας θα το καλύψουμε, θα διορθώσουμε κάποια από τα λάθη σας αυτά που βλέπουμε στο νέο πακέτο μέτρων αλλά για το πρόγραμμα δράση έχω κάποιε ερωτήσει, γιατί δεν είναι καθόλου σαφέ το τι μπορούμε να περιμένουμε. Και θέλω σαφεί απαντήσει από πλευρά σα. Πρώτον, το γενικό στόχο για την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων. Στην τελευταία ανακοίνωση, αν κοιτάξουμε την ιεράρχηση των αποβλήτων και τα λοιπά και το ποιο είναι το πιο σημαντικό πρέπει να γίνει, σημειώνετε κι εσείς ότι πρέπει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στη χρήση των πόρων. Υπήρχαν και στα προηγούμενα πακέτα σαν στόχοι η καλύτερη αποτελεσματικότητα ε, στη χρήση των πόρων, αλλά τώρα δεν βλέπω να το λέτε. Και στην ανακοίνωση αναφερόταν την περασμένου έτους ότι θα μπορούσε να μπει αυτός ο στόχος της ε, αποτελεσματικής χρήσης των πόρων και στο εξάμεινο, το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Τώρα χάθηκε, δεν το βλέπουμε να το λέτε αυτό. Μας εξηγείτε λοιπόν πώς το γενικό θέμα της αποτελεσματικής χρήσης των πόρων θα καλυφθεί γιατί δεν αναφέρεται ο στόχος ο συγκεκριμένο σε αυτό το στάδιο. Πρώτο αυτό. Δεύτερον, για τα απόβλητα για τα απόβλητα αποτρόφιμα και τη σχετική σπατάλη. Αυτό που λέτε στο παράρτημα μόνο είναι ότι αναφέρετε πως για το 2016 θα εντοπίσετε την ε, ευρωπαϊκή νομοθεσία που έχει να κάνει με την ε, σπατάλη ή τα απόβλητα σε τρόφιμα και ζωοτροφές. Ε, τι σημαίνει αυτό. Ήδη έχουμε ένα πρόγραμμα δράσης μετά τη συνομοθεσία διαδικασία όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε υποσχεθεί πως θα καταθέσει μια ε, πλήρη μελέτη για την αντιμετώπιση της πατάλης στα τρόφιμα. Αυτό είναι μετά τα, το 7ο πακέτο. Και τώρα, και ήταν πολύ πιο σαφές από αυτά που βλέπουμε τώρα στις προτάσεις σας. Πολύ ε, ασαφής η διατύπωσή σας και παρακαλώ να μας εξηγήσετε πιο συγκεκριμένα. Τρίτον, τίθεστε να καταθέσετε του χρόνου μία πρόταση για την αποτελεσματική χρήση της ενέργειας. Ναι. Το πιο ανόητο όμως το μπορούσε να κάνει κανείς σε σχέση με τα απόβλητα, πέραν της χωματερής ή μετά τη χωματερή, είναι η αποτέφρωση των αποβλήτων. Και φαίνεται ότι στο στόχο της ενέργειας έχετε ακριβώς την ε, διοχέτευση των αποβλήτων στους αποτεφρωτήρες. Πώς θα το κάνετε αυτό λοιπόν, ή εξηγήστε μας, είναι συγκεκριμένο στόχος. Επίσης, πέντε είναι τα σημεία μου, πρόεδρε, και θα καταλήξω όπου να είναι. Για το FC. Το πρόγραμμα Juncker. Μας λέτε ότι θα ενθαρρύνουμε στόχους που ισχύουν για το πρόγραμμα επενδύσεων Juncker. Ναι, αλλά κάθε φορά που γίνεται συζήτηση για το FC, μας λέτε ότι δεν πρέπει να πολιτικοποιηθεί και να το αφήσουμε στα διαχειριστικά του όργανα, στα management boards, στα διοικητικά ε, όργανα. Άρα τι ισχύει και με ανησυχεί αυτή σας η αναφορά. Επίσης ε, για την παραποίηση του κυκλικού, ε, για τα χημικά στο κυκλικό μοντέλο. Λέτε ότι πρέπει τα χημικά να μπαίνουν στο κυκλικό μοντέλο, αλλά ταυτόχρονα χορηγείται για την ευθαλάτη DHP την ε, δυνατότητα να αξιοποιηθεί για PVC ε, ήπιας ανακύκλωσης όπως το λέτε. Κάτι το οποίο έχει απορρίψει μόλις πριν από μερικές εβδομάδες η Ολομέλεια του Κοινοβουλίου. Δηλαδή το ξαναβάζετε μέσα ενώ είναι επικίνδυνη ουσία και το ξαναβάζετε στην ε, αλυσίδα της ανακύκλωσης Λοιπόν, παρακαλώ να κάνετε κάποιες διορθώσεις ουσιαστικές για να μην ε, ε, κηρύσετε τα αντίθετα από αυτά που έχετε υποσχεθεί. Ο πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ και χαίρομαι που δεν είχες δέκα σημεία. Έχω και δεύτερο γύρο, πρόεδρε. Θα επανέλθω. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν θα επαναλάβω τόσο υπόθηκαν ήδη σε σχέση με τις μεγαλύτερες φιλοδοξίες που μας ανακοινώθηκε επαγγελμένως από πλευρές κομισιών, το είπαν ήδη όλοι. Αλλά θα ήθελα να αναφερθώ πιο συγκεκριμένα στη διευρυμένη ευθύνη καθώς και στην πρόληψη των αποβλήτων. Εμείς ανέκαθεν θεωρούσαμε ότι η διευρυμένη ευθύνη αποτελεί βασικό εργαλείο για τη μείωση των αποβλήτων και τη σωστή τους διαχείριση. Και πιο συγκεκριμένα υποστηρίζουμε το αίτημα να πληρώνουν πλήρως η παραγωγή το κόστος ανακύκλωσης των αποβλήτων καθώς και το κόστος εκπαίδευση των πολιτών για τη σωστή του διαχείριση. Ταυτόχρονα όμως θεωρούμε ότι θα πρέπει να υποστηρίζουμε τους παραγωγούς στη μεταβατική φάση ε, κατά την οποία θα πρέπει να πληρώνουν λιγότερο για τα πιο αποτελεσματικά προϊόντα και τα προϊόντα που έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και για εκείνα φυσικά τα οποία είναι ανακυκλώσιμα και παραχρησιμοποιούμενα. Όσον αφορά τα απόβλητα, εμεί συμφωνούμε με τα όσα είπε ο Πρόεδρο και ο Επίτροπο. Θεωρούμε ότι πρέπει να αποτελέσει πολιτική προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, στο πλαίσιο τη ε, διαχείριση των αποβλήτων. Στην πρόταση λοιπόν τη Κομισιόν βρίσκουμε μόνο μία σειρά από συστάσει προ τα κράτη-μέλη που δεν έχουν καμία δεσμευτική αξία. Οπότε έχω να ρωτήσω τα εξή. Τι μέτρα έχει προβλέψει η Κομισιόν ώστε τα κράτη-μέλη να διαβεβαιωθούν ότι καταβάλουν το πλήρες κόστος των αποβλήτων η σχετική παραγωγή δεδομένου της πατάλα 100 τόνους ε, τροφίμων η Ευρωπαϊκή Ένωση ετησίως πώς θα το αντιμετωπίσει το πρόβλημα τρίτον αφού ε, ο στόχος δεν ε, ευθυγραμμίζεται με την ιεραρχία αποβλήτων και επειδή ορισμένα δημοτικά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πώς πιστεύετε εσείς ο Κομισιόν ότι μπορείτε να προωθήσετε την επαναχρήση χωρίς δεσμευτικούς ε, στόχους. Τέλος, γι' αυτό το 10% των δημοτικών αποβλήτων μέχρι το 2030 που αναφέρετε δεν πιστεύετε ότι έχουν γίνει πολύ λίγα ε, μέχρι στιγμής ε, ώστε να διευκολύνεται πράγματι τη μετάβαση προς την κυκλική οικονομία. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Ντονάνο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, η ευρωπαϊκή οικονομία σπαταλάει πάνω από το ίμιση των πρώτων υλών που θα μπορούσαν να ανακυκλωθούν Πιστεύω ότι πρέπει να σας ρωτήσουμε πάνω σε αυτό το θέμα. Βέβαια πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι κάθε ρύθμιση πρέπει να προσφέρει συγκεκριμένο ωφέλη προς τις χώρες μέλη. Δύο ερωτήσεις μου. Τι στοιχεία θετικά για την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών οικονομιών προβλέπονται στα μέτρα που προτείνεται. Στο νομοθετικό πακέτο προτείνεται μια τροποποίηση της οδηγίας του 98 για τα απόβλητα όπου προβλέπονται διάφορες εξαιρέσεις για διάφορες χώρες όσον αφορά την προθεσμία που έχουν για να πετύχουν τους στόχους ανακύκλωσης. Δεύτερον, τι λόγους μπορείτε να μας δώσετε γιατί είναι ευπρόσδεκτη αυτή η ελαστικότητα. Γιατί δεν προτείνεται ένα πιο ελαστικό σύστημα γενικά ώστε να μπορούμε να ενισχύσουμε την αντοχή των διαφόρων πλευρών. Και όσον αφορά την ανακύκλωση των ηλεκτρονικών μηχανημάτων και των ε, μπαταριών, εδώ και πάλι ε, μπαίνει το θέμα και υπάρχουν πολλές δράσεις και στην αυτοκινητοβιομηχανία και αλλού σε διάφορες κλίμακες. Ποιοι φορείς της οικονομίας ή της κοινωνίας των πολιτών ε, ρωτήθηκαν από εσά με ποιους διαβουλευτήκατε και γιατί δεν υπάρχει αρκετή προβολή αυτού του θέματος. Ευχαριστώ. Αυτές ήταν οι ερωτήσεις μου. Πρόεδρος. Ευχαριστούμε. Ο Επίτροπος τώρα. Παρακαλώ, έχετε 10 λεπτά για να απαντήσετε. Ευχαριστώ. Θέλω να αναφερθώ πράγματι σε διάφορα σημεία από πλευράς ε, της Επιτροπής για αυτά που είπατε όσον αφορά την ελληνική φιλοδοξία κλπ. Κοιτάξτε, είναι δύσκολο να συγκρίνει κανείς αυτά που προτείνουμε τώρα με αυτά τα οποία αποσύραμε. Γιατί αποσύραμε την οδηγία για τα απόβλητα που ήταν ε, το τέλος μιας ε, γραμμικής διαδικασίας, ενός γραμμικού μοντέλου και τώρα προτείναμε ένα πακέτο για την κυκλική οικονομία που είναι σφαιρικό. Πιστεύουμε ότι είναι πιο ισορροπημένη η προσέγγιση αυτή. Τώρα, γιατί είναι πιο φιλόδοξο το πακέτο αυτό. Πρώτον, γιατί πρόκειται για ένα πρόγραμμα δράση, πρόκειται για το εύρο εφαρμογή. Το εύρο εφαρμογή έχει να κάνει και με την ε, παραγωγή και την ε, κατανάλωση, την ε, ανακύκλωση των αποβλήτων. Πρόκειται δηλαδή για πολλαπλούς τομείς που είναι από το, την οικολογική, τον οικολογικό σχεδιασμό, πρόκειται για τους διαγωνισμούς, για τις δημόσιες προμήθειες κλπ. Μιλάμε για μέτρα επίση στήριξη, τα οποία ευθυγραμμίζουν όλα τα μέτρα τα οποία πρέπει να λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να βοηθήσει. Είναι λοιπόν ένα θεματολόγιο πολύ φιλόδοξο πιστεύω εμεί που θα μα απασχολήσει για ολόκληρη την εντολή μα. Τώρα όσον αφορά την νομοθετική πρωτοβουλία για τα απόβλητα. Χρειαζόμαστε διαχείριση αποβλήτων, βοηθάει την κυκλική οικονομία. Οι πρώτε ύλε το να καταλήγουν στις χωματερές είναι πράγματι θλιβερό, ενώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην οικονομία μας. Και αυτό το έχουμε λάβει υπόψη μας. Τώρα έχουμε δεσμευτικούς στόχους για τους χώρους υγιεινής γεωνομικής ταφής. Απλοποιούνται οι κανόνες. Είναι κάτι πιο εύκολο, πιο προσιτό για το χρήστη και λαμβάνει υπόψη πολύ περισσότερο και καλύτερα τις επιδόσεις των χωρών μελών. Και έχουμε ήδη πει ότι έχουμε 28 χώρες μέλη με 28 διαφορετικές ταχύτητες. Η επιλογή που έχουμε είναι είτε να επιλέξουμε το ίδιο επίπεδο φιλοδοξίας και να βοηθήσουμε τις χώρες μέλη που καθυστερούν περισσότερο ή εξαιτία των χωρών αυτών που βρίσκονται πιο πίσω, έχουν καθυστερήσει επίτευξη των στόχων, να κατεβάσουμε και τι φιλοδοξίε μας. Ε, όχι, προτιμήσαμε το πρώτο. Οι χώρες που βρίσκονται πιο πίσω θα βοηθηθούν από εμά για να κερδίσουν τη χαμένη απόσταση. Όσον αφορά το πρόγραμμα δράσης, γιατί πολλοί από εσά αναφέρθηκαν στο πρόγραμμα δράσης, βεβαίως και έχουμε πολλές νέες ιδέες και κίνητρα. Και πρώτα απ' όλα έχουμε τον στόχο διοχέτευσης πολλών κονδυλίων και πόρων υπέρ της κυκλικής οικονομίας. Είπαμε για τον ορίζοντα 2020 ε, που είναι 650 εκατομμύρια. Είναι τα διαστροτικά ταμεία και όταν λέμε για διαστροτικά κάποιος από σας μίλησε για την αποτέφρωση. Μα όταν μίλησε για τα διαστροτικά ταμεία πριν είπα ότι από την αποτέφρωση των αποβλήτων θα αλλάξουμε. Πολλοί από εσά αναφέρθηκαν στις σπατάλη τροφίμων. Ναι, μα υπάρχουν οι στόχοι και στους στόχους της ε, βιώσιμης ανάπτυξης. Όλοι οι στόχοι τώρα είναι δεσμευτικοί και πρέπει οι χώρες μέλη να υποβάλουν σχέδια για να μας δείξουν πώς θα μειώσουν τις σπατάλη τροφίμων. Είναι μέτρα τα οποία θα συζητηθούν στη συνέχεια. Παράδειγμα, Υπάρχει μεγάλη σύγχυση για την ημερομηνία λήξης ενός προϊόντος. Όλοι λένε ότι αν δούνε η ημερομηνία 1 31η Δεκεμβρίου, αυτό σημαίνει ότι την επόμενη μέρα πρέπει να πετάξεις αυτό το προϊόν. Δεν ισχύει όμως. Ίσως χρειαζόμαστε κάτι που να λέει ότι είναι καλύτερο πριν και μία ημερομηνία λήξη. Γιατί η ημερομηνία που λέει ότι είναι καλύτερο πριν δεν σημαίνει ότι λύγει το προϊόν την επόμενη. Πολλές οργανώσεις επίσης φοβούνται να δίνουν τα τρόφιμα τα οποία είναι μετά την ημερομηνία που αναφέρεται ως το προϊόν είναι καλύτερο πριν από. Και αυτό θα το κοιτάξουμε. Επίσης, εκπονούμε μεθοδολογία για να δούμε πώς μπορούμε να υπολογίσουμε τη σπατάλη τροφίμων. χρόνο, ποσότητα κλπ. Αναφερθήκατε στην ανακύκλωση. Φυσικά και θα αναπτύξουμε την αγορά ανακύκλωσης, γιατί ακόμα και σήμερα, μετά την διαλογή και την ανακύκλωση, πολλά από τα υλικά, τα, ανακυκλου, τα ανακυκλωμένα, δεν βρίσκουν το δρόμο τους και πάλι στην παραγωγή. Αναφερθήκατε επίσης στην καλύτερη επιλογή των καταναλωτών. Μα και εδώ ο οικολογικός σχεδιασμός και το να αντέχουν περισσότερο στον χρόνο τα προϊόντα είναι κάτι που θα συμπεριλάβουμε ο οικοσχεδιασμός δεν έχει μόνο την ενεργειακή απόδοση όπως είχε μέχρι τώρα. Τώρα μιλάμε και για την ανθεκτικότητα και για την αβάθμιση, για ένα σωρό άλλα πράγματα. Μέχρι τώρα ο οικολογικός σχεδιασμός ήταν κυρίως ενεργειακή απόδοση. Τώρα το συνδυάζουμε αυτό. Την ενεργειακή απόδοση δηλαδή με την ε, χρήση διαρκείας των πόρων, των υλών. Επίσης αναφερθήκατε στην προγραμματισμένη παλαίωση λήξη ζωή ενό προϊόντος, ότι μερικά προϊόντα προγραμματισμένα για να αντέξουν στον χρόνο δύο χρόνια, τρία χρόνια. Ε, λοιπόν, με την έρευνά μας θα εντοπίσουμε ποια είναι αυτά τα προϊόντα και θα φροντίσουμε να αναλάβουμε δράση. Για τα πλαστικά. Όλοι γνωρίζουμε το δίλημα που έχουμε με το πλαστικό. Η στρατηγική για το πλαστικό στην κυκλική οικονομία πιστεύω ότι είναι πολύ καλή γιατί θα αντιμετωπίσει και τις ε, επικίνδυνες ουσίες και την βιοαποδόμηση κλπ. Έπειτα, για τα θαλάσσια απόβλητα. Και εδώ υπάρχει δέσμευση να βελτιωθεί αυτό και να μειωθούν 30% τα σκουπίδια που έχουμε στη θάλασσα μέχρι το 2030. Αναφερθήκατε στα τρόφιμα αλλά εκτό από τις πατέλες τροφίμων πρέπει να δούμε τι γίνεται και με τις κατασκευές και εκεί θα ασχοληθούμε. Κάποιος επίσης αναβέρθηκε και στην καινοτομία και την έρευνα. Εξετάζουμε τις παγκόσμιες προκλήσεις της κυκλικής οικονομίας, γιατί δεν έχει νόημα για μια πολυεθνική, μια διεθνή επιχείρηση να λειτουργεί στην Ευρώπη με μια κυκλική οικονομία ενώ αλλού δεν υπάρχει κυκλική οικονομία. Ευτυχώς υπάρχουν και χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που ήδη έχουν υιοθετήσει την κυκλική οικονομία. Επάρκεια πόρων. Ο Μπάς το είπε. Ναι, είναι κάτι που το έχουμε ζητήσει και πολλοί ευρωβουλευτές. Η μεταβίβαση τώρα στην κυκλική οικονομία πρέπει να δούμε πώς θα γίνει. Η μέτρηση της επάρκειας σπόρων είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, της απόδοσης των πόρων είναι πάρα πολύ δύσκολο. Υπάρχει πολιτική στήριξη πάντως. Θέλουμε ναι, την πρόοδο στην κυκλική οικονομία και το πρόγραμμα δράσης ακριβώς αυτό δείχνει ότι θα υπάρξει τέτοιο πλαίσιο. Όσον αφορά τώρα την σπατάλη ενέργειας, όντως ε, δεν θέλουμε ούτε και εμείς να επενδύσουμε στην ε, αποτέφρωση των σκουπιδιών, εκτός αν αυτό είναι αναγκαίο και αιτιολογείται. Το έχουμε συμπεριλάβει και αυτό. Επίσης, να ξέρετε ότι έχουμε σημειώσει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για όλα τα θέματα και το συζητάμε αυτό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πάντως, η ανακύκλωση δεν θα πρέπει να έχει σαν αποτέλεσμα επικίνδυνα προϊόντα να παραμένουν σε αυτά που χρησιμοποιούμε. Η οικονομική μας στρατηγική είναι τέτοια που θέλουμε να αντιμετωπίσουμε και το θέμα της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αρχίσει ήδη συζητήσεις με την ΕΚΑ προκειμένου να δει πώς ε, μπορεί να βελτιωθεί το θέμα των αδειών στα διάφορα προϊόντα. Επίσης, όσον αφορά την ερώτηση τη κυρία Μποναφέ για του στόχους και για το πώς μπορούμε να τους μετρήσουμε, εγώ πιστεύω ότι ο πιο βασικός στόχος που έχουμε θέσει εμείς είναι το 10% όσον αφορά την υγειονομική ταφή. Μπορούμε να αντιστρέψουμε το επιχείρημα και να σας πω ότι αν επιμείνουμε στο 10% για την υγειονομική ταφή, κοίταξτε, είναι ο στόχος αυτός ο οποίος θα προωθήσει περισσότερο την κατάσταση ώστε τα απόβλητα να ανακυκλώνονται. Δηλαδή το 90% των σκουπιδιών θα πρέπει να είτε να ανακυκλωθούν είτε να επαναχρησιμοποιηθούν μόνο αν είναι αναγκαίο να καταλήξουν στην υγειονομική ταφή. Είπε η κυρία Μποναφέ ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να συζητάει και να υποβάλει προτάσεις. Και εμείς θα συνεχίσουμε να σας ακούμε. Μάρκ, ένα από τα καλά πράγματα που είπε ο Μάρκ είναι ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα στην πηγή του. Και είναι ακριβώς αυτό που κάνουμε. Δεν μπορούμε να χάνουμε το δάσος για το δέντρο και να συγκρίνουμε το 65% το στόχο ανακύκλωσης. Γιατί, γιατί πριν φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο, ακριβώς αυτό κάνουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα στην πηγή. Δηλαδή, αποφεύγουμε τα πόβλητα. Είναι χίλιες φορές καλύτερο. Ποια είναι η χρήση του να μην κάνουμε τίποτα για την παραγωγή σκουπιδιών, αλλά ασχολούμαστε με το πώς θα τα διοχετεύσουμε καλύτερα. Άρα λοιπόν ξεκινάμε από την αποφυγή συσσόρευσης σκουπιδιών και μετά προχωράμε στη διαχείρισή τους. Έρχομαι τώρα και στην ομοθεσία. Στη φιλοδοξία, αν είναι αρκετή ή όχι. Κοιτάξτε, μπαίνουμε σε ένα διέξοδο ή που θα έχουμε υπερβολική νομοθεσία και καθόλου εφαρμογή ή το αντίθετο. Εγώ νομίζω ότι η κατεύθυνση που έχουμε πάρει είναι να έχουμε μια καλή ισορροπία στην νομοθεσία και στην εφαρμογή της. Προσπαθούμε δηλαδή να έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε από την νομοθεσία που έχουμε υιοθετήσει. Για τις εξαιρέσεις τώρα που έχουν δοθεί σε διάφορες χώρες μέλη, Έχω εξηγήσει ότι η ιδέα μας δεν είναι να τιμωρήσουμε τις χώρες που δεν έχουν πετύχει τους στόχους, αλλά να εντοπίσουμε γιατί δεν έχουν εφαρμόσει τους στόχους και από εκεί και πέρα να τις βοηθήσουμε να τους πετύχουν. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν πολύ καλά παραδείγματα στη Φλάνδρα όπως είπατε, αλλά δεν συμφωνώ ότι πυροβολήσαμε τον εαυτό μας τα πόδια όταν αποσύραμε την προηγούμενη πρότασή μας. Ναι, είμαστε καινούργοι και το έχουμε πει από την αρχή ότι την κυκλική οικονομία δεν θα τη δούμε μόνο από την περιβαλλοντική οπτική γωνία αλλά και από οικονομική. Τι είπαμε από την αρχή ότι ακριβώς αυτό είναι το χαρακτηριστικό παράδειγμα μίας λύσης και για το οικονομικό σκέλος και για το περιβαλλοντικό. Αν τώρα από πλευρά ε, οικονομικής θα πετύχουμε τους στόχους μας για περισσότερες επενδύσεις, για περισσότερη οικονομική ανάπτυξη και απασχόληση, τότε σίγουρα πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί. Δυστυχώς δεν μπορούμε να πετύχουμε μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα μειώνοντα τους μισθούς, δεν είναι αυτό που θέλουμε, αλλά μπορούμε να πετύχουμε περισσότερη ανταγωνιστικότητα μέσω αυτού του συστήματος μεγαλύτερη και καλύτερης απόδοσης των ε, υλών, των πόρων. Είμαστε ισχυροί και πλούσιοι σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο, αλλά είμαστε πολύ φτωχοί όταν μιλάμε για πρώτες ύλες και γι' αυτό και πρέπει την απόδοση των πόρων στην κυκλική οικονομία να είναι κάτι που θα το πάρουμε πάρα πολύ σοβαρά. Το, ότι συγκρίνουμε το χάρτη πορείας που είχαμε με το πρόγραμμα δράσης, ε, ο χάρτης πορείας παραμένει χάρτης πορείας. Τώρα έχουμε ένα πρόγραμμα δράσης. Είναι κάτι άλλο. Και αν συνεργαστούμε όλοι, τότε θα μπορέσουμε να πετύχουμε και το αποτέλεσμα που πραγματικά θέλουμε. Ο κύριος Πιεντιτσίνη ήταν εκείνος ο οποίος αναφέρθηκε στην ε, ευθύνη παραγωγής. Υπάρχει στο πρόγραμμα δράσης μας και ελπίζουμε να δώσουμε κίνητρα για καλύτερα προϊόντα που να ανακυκλώνονται, να επιδέχονται ανακύκλωση και ότι η παραγωγή θα πληρώνουν λιγότερα για την ανακύκλωση, όσο καλύτερο δηλαδή για ανακύκλωση είναι το προϊόν τους, τόσο λιγότερο θα πληρώνουν. Τι άλλο, ε, τον Άνω. Κύριε τον και συμφωνώ. Γιατί το είπα, ότι 50% δεν ανακυκλώνεται ακόμα από τα απόβλητα. Βέβαια υπάρχουν κάποιες χώρες μέλη που έχουν προδιαγραφές τέτοιες που αποτελούν ένα καλό παράδειγμα, αλλά δυστυχώ υπάρχουν άλλες χώρες που δεν το κάνουν. Και όσον αφορά την ευελιξία, πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε ευέλικτοι και γι' αυτό δεν μπορούμε να πούμε ότι ένα μέτρο το ίδιο για όλους, γιατί το έχουμε να κάνουμε με διαφορετικά προϊόντα, με διαφορετικά υλικά και το κάθε προϊόν και το κάθε υλικό προφανώς και έχει δικούς του στόχους. Θα ολοκληρώσω ευχαριστώντας σας για την στήριξη που μας προσφέρετε. Ελπίζω να μπορέσουμε να συζητήσουμε το θέμα με περισσότερες ακόμα λεπτομέρειες να ξέρετε ότι θα στηρίξουμε τους συνομοθέτες προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι και δράτω με τις ευκαιρίες αυτής για να ευχηθώ σε όλους σας ό,τι επιθυμείτε. Καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο τον καινούριο χρόνο, αλλά ο πρόεδρος διακόπτει. Μη δεν φεύγετε ακόμα κύριε Επιτροπέ, μη βιάζεστε. Δεν φεύγετε. Γιατί έχω εδώ ένα κατάλογο με 12 ακόμα ομιλητές. 20 λεπτά. Ένα λεπτό λοιπόν ο καθένας, γιατί πρέπει να φύγει ο Επίτροπος. Πρέπει να πάρω αεροπλάνο, γι' αυτό το λέω. Ωραία, Ιβο Μπελέτ. Πολύ σύντομο παρακαλώ. Όντως ένα λεπτό μόνο, κύριε Επίτροπε. Και ευχαριστώ πολύ που δέχεστε να μείνετε και για το δεύτερο γύρο. Βεβαίως, συμφωνούμε ότι έφτασε με καθυστέρηση και δεν έχει και πολλές φιλοδοξίες αυτή η δεύτερη ε, πρόταση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέει και ο Καρλ Χάιντς Φλόρενς ότι πρέπει να μιλούμε και για την οικονομία όχι μόνο για το περιβάλλον και θα πρέπει να αποφεύγονται βέβαια οπωσδήποτε οι αποτεφρώσεις και όλα αυτά. Το πλαστικό έχει πολύ μεγάλη σημασία, το 25% μόνο και λιγότερο μάλιστα ε, του πλαστικού συλλέγεται και είναι πολύ ανησυχητικό στοιχείο. Θα θέλαμε λοιπόν πιο πολλές λεπτομέρειες σε αυτό. Δεν θα αναφερθώ στο βελγικό μοντέλο βεβαίως γιατί έχει ήδη αναφέρει ο Μάρκο ο οποίος έχει φύγει εντωμεταξύ. μεταξύ αλλά στην οδηγία για την ε, διακίνηση αποβλήτων, μεταφορά αποβλήτων. Λέμε ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας ώστε να ε, αποφύγουμε την ιαδήποτε διαρροή από την ευρωπαϊκή οικονομία οποιοδήποτε υλικού ανακύκλησης και ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να δημιουργήσουμε αυτή την εσωτερική θα λέγαμε αγορά του, των δευτερογενών υλικών. Ε, τι έχετε να πείτε γι' αυτό, Ματίας Γκρότε τώρα. Ευχαριστώ και εγώ πολύ σύντομα. Τι, έχετε να πείτε για την ε, απόθεση σε χωματερές υλικού το οποίο βρίσκεται στο τέλος της αλυσίδας και δεν πρέπει να αποτίθεται σε χωματερές που δεν έχει δηλαδή αξιοποιηθεί πλήρως. Αυτό πρέπει ιδιαίτερα να το ε, κοιτάξουμε για την προγραμματισμένη παλαίωση δηλαδή προγραμματισμένη σπατάλη, θέλω να, να δώσετε συγκεκριμένες προτάσεις κύριε Επίτροπε. Αντίστοιχα με αυτά των συστημάτων καθαρισμού των καυσαερίων. Εάν ε, φτάνει ένας καταλήτης στο τέλος της ζωής του, ύστερα από κάποιον αριθμό χιλιόμετρων, τότε θα πρέπει να ξέρουμε και γιατί πρέπει να χαλάσει ένα, ε, μια συσκευή, ένα μηχάνημα που χρησιμοποιούμε στα σπίτια μας πρόωρα. Το πλαστικό επίσης που βλέπουμε στις θάλασσες. Βλέπουμε ότι στη Βόρεια Θάλασσα οι αλείς βρίσκουν πλαστικές σακούλες και μεγάλα κομμάτια πλαστικού και τα μαζεύουν από τη θάλασσα. Υπάρχει όμως το Life Plus που προβλέπει, κάποια, που προβλέπει την, ε, τον καθαρισμό των θαλασσών και πρέπει να γίνει αυτό. Διαφορετικά κάποια στιγμή αυτό το πλαστικό θα φτάσει στο πιάτο μας. Ευχαριστώ, Μπέλντερ. Όχι. Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε. Θα μιλήσω Ολλανδικά, μια και είναι τεχνικό το θέμα. Οι επιχειρήσεις, ναι, πρέπει να υιοθετήσουν την κυκλική οικονομία. Φυσικά, οι πρώτες ύλε σπανίζουν, φυσικά. Η γεωργία όμως παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για την πράσινη οικονομία. Οι επιχειρήσεις όμως είναι αυτές οι οποίες παράγουν τα τρόφιμα κρέας για παράδειγμα. Είναι κρίμα που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελάχιστα πράγματα ε, λέει και δεν νομίζω ότι θεωρεί την γεωργία τη λύση για την κυκλική οικονομία και την πράσινη οικονομία και είναι κρίμα, είναι μια χαμένη ευκαιρία αυτή. Χρειάζεται περισσότερη νομοθεσία, καλύτερη ρύθμιση που να λαμβάνει υπόψη και τις νέες τεχνικές. Για μένα το βασικό είναι η σχέση των πρώτων υλών με, την, ε, τα λοιπάσματα και πώς από τα λοιπάσματα μπορούμε να πάρουμε τις πρώτες ύλες. Πρέπει λοιπόν να προσαρμοθούν οι τεχνικές ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ύλε αυτές και να μπορούν να φτιαχτούν και πάλι λοιπάσματα. Τα βασικά μέταλλα, για παράδειγμα, τα οποία παίρνουμε από διάφορες ε, ύλες με την ανακύκλωση, να χρησιμοποιούνται μετά στα λοιπάσματα. Έτσι θα έχουμε μια κατάσταση από την οποία όλοι έχουν να κερδίσουν και η οικονομία και η οικολογία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Φλάνναγκαν. Κύριε Φλάνναγκαν. Ζητά συγγνώμη κύριε Φλάνναγκαν. Όπως φαίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση η κυκλική οικονομία είναι σαν ένα σκύλο που κυνηγάει την ουρά του. Κάνει κύκλους όλη την ώρα. Ε, πραγματικά είναι κυκλική η διαδικασία αλλά δεν επιτυχαίνει ποτέ τίποτα. Άκουσα διάφορα σχόλια εδώ σήμερα και ειδικότερα τον κύριο Κερπράντη. Είναι σαφές ότι αυτό κάνουμε. Έχουμε μπει σε ένα φαύλο κύκλο. Από τη δική μου εμπειρία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορείτε να οργανώσετε τίποτα. Πώς θα οργανώσετε την ανακύκλωση. Είπε εδώ κύριος συνάδελφος ότι ο κόσμος το συζητάει. Ναι, ξέρετε, μακάρι να το συζητούσαν. Γιατί είναι μάλλον το σημαντικότερο πράγμα που έχουμε κάνει ποτέ. Αλλιώς θα καταλήξουμε να ζούμε μέσα στα σκουπίδια μας. Ε, το θέμα αυτό αφορά το μέλλον μας. Αλλά ξέρετε, κανείς δεν το συζητάει. Ελάχιστο είναι το ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί γι' αυτό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνουμε τους ανθρώπους να ενδιαφερθούν. Οπότε πρέπει να κάνουμε κάτι γι' αυτό και το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να το βιώνουμε, να δίνουμε ένα ε, ποτήρι στους ανθρώπους να πιούν από έναν ψύκτη, αντί να τους δίνουμε ένα μπουκαλάκι, όταν πάνε να πάνε ένα καφέ, να τους δίνουμε μια κανάτα με καφέ, αντί για πράγματα που δεν είναι ανακυκλώσιμα πρέπει να αρχίσουμε να το εφαρμόζουμε εδώ. Πρέπει το φαγητό που ανακυκλώνεται, που βιοδιασπάται να το βάζουμε ξεχωριστά. Μόλις μπήκαν σε αυτό εδώ το κοινοβούλιο παρατηρεί αμέσω ότι όλο λόγια είμαστε αλλά δεν κάνουμε τίποτα. Και ξέρετε κάτι, δεν μπορούμε να οργανώσουμε ούτε καν μια συνάντηση σωστά. Αν είχε οργανωθεί σωστά θα είχε τελειώσει τώρα. Οπότε και εγώ θα πάω να ακούσω την κόρη μου να λέει τα κάλαντα. Έπρεπε να είχαμε τελειώσει με το αυτό δεν μπορείτε να κανονίσετε. Πείτε με κοινικό, αλλά ούτε αυτό δεν μπορείτε να καταφέρετε. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ κυρία Σέβη. Κυρία Εύη, συγγνώμη. Ναι, ευχαριστώ. Λοιπόν, ε, το να λέμε ότι αυτή η νέα πρόταση είναι φιλόδοξη Είναι ε, σαν να ξεχνάμε ε, τις αναλύσεις, τις εκθέσεις, τις έρευνες ε. που μας λένε πως υψηλές φιλοδοξίες μπορούν να δημιουργήσουν δραστηριότητα, θέσεις εργασίας και μείωση του κόστους κτλ. Όλα αυτά εμένα μου φαίνονται αντιφατικά. Η πρόταση εδώ που έχουμε μπροστά μας ε, είναι, δεν είναι και τόσο φιλόδοξη. Κάτι άλλο που ήθελα να πω, χωρίς να επαναλαμβάνω τα όσα είπαν οι συναδελφοί. Αν θέλατε να είναι φιλόδοξη αυτή η πρόταση, ε, έπρεπε να προτείνετε και μείωση των υλικών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ενός προϊόντος ε, με επιλογή των ε, περισσότερο περιβαλλοντικά φιλικών προϊόντων. Ε, ε σκέφτομαι τώρα τα πλαστικά λέγοντα αυτό. Αυτό πρέπει να κάνετε. Ένα άλλο φιλοδοξό στόχο θα ήταν ε, όταν επελθέδεται η επίτευξη των στόχων της ανασκύκλωσης να υπολογίζαμε το κλάσμα των υλικών που προέρχεται από ε, απόβλητα τα οποία προέρχονται από πρωτεσίλες που δημιουργούνται για πρώτη φορά αλλιώς δεν έχει νόημα Κάτι άλλο που θέλω να υπογραμμίσω. Όταν δημιουργούμε μια αγορά δευτερευόντων υλικών, ε, αν δεν κάνουμε μια θετική διάκριση μεταξύ δευτερευόντων υλικών, δηλαδή ανακυκλωμένων, ε, αν δεν υπάρχει διάκριση αυτών των υλικών από αυτά που δημιουργούνται για πρώτη φορά, που χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά, δεν θα καταφέρουμε να ορίσουμε ε, κανονικά ε, χρήσιμα μέτρα για μια αγορά που θα χρησιμοποιεί ανακυκλώσιμα υλικά. Ευχαριστώ κύριε Όσλεντ. Ναι. Ο κύριος Τίμερμανς ήθελε να μας παρουσιάσει πιο φιλόδοξα σχέδια. Δεν βλέπω λοιπόν πού είναι τώρα η διαφορά και η φιλοδοξία σε σχέση με αυτά που είχατε καταθέσει το 2014. Γιατί εγώ δεν βλέπω καμία διαφορά. Και βλέπω ότι θέλετε το 2020 να κάνετε τη διαφοροποίηση των αποβλήτων οργανικά από μη. Αλλά φαίνεται ότι απαντούν κάποιοι πως αυτός ο διαχωρισμός δεν έχει οικονομικά, ε, οικονομικό συμφέρον και άρα μπορεί να απορριφθεί για τέτοιους όρους. Λυσμονώντας βέβαια ότι υπάρχει η ιστορία του μεθανίου στην υπόθεση αυτή και για την ε, σπατάληση τρόφιμα. Εάν δεν καταθέσουν ε, και τα κράτη-μέλη προτάσεις, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Έχει κάνει το Κοινοβούλιο τις ε, δικές του ε, για το πώς μπορούμε να περιορίσουμε την παραγωγή και τη σπατάλη, αλλά βλέπουμε σχέδια όχι φιλόδοξη, για να το πω ευγενικά. Ευχαριστώ πολύ. Γκαρτίνη. Ευχαριστώ πολύ γρήγορα γιατί δυστυχώς ε, άργησε η πτήση μου και έχασα την αρχή της συνεδρίας. Λοιπόν, εμένα θα με ενδιαφέρει να καταλάβω πώς μπορούμε να τα εντάξουμε όλα αυτά σε μια ολιστική προσέγγιση. Γιατί εγώ να επικροτώ την κυκλική οικονομία, αλλά δυστυχώς συχνά παρατηρούμε ότι εδώ στην Ευρώπη ε, αντιμετωπίζουμε τα πράγματα κατά ε, αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη και όλα αυτά που λέτε να τα εφαρμόσουμε πιο ολιστικά. Όταν μιλάμε για χάλιβα, που είναι ένα υλικό κατεξοχήν υλικό της ε, κυκλικής οικονομίας, μπορεί να ανακυκλώνεται επάπειρον. Όταν λοιπόν σε άλλα μέτωπα έχουμε πολιτικές ε, που υπάρχει κίνδυνος ε, ε, για, το ETS, ε, για τα ETS, για την περιβαλλοντική πολιτική υπάρχει κίνδυνος ε, να προκαλέσουν απώλεια ενός τόσο σημαντικού βιομηχανικού τομέα δεν θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιο σύστημα συντελεστών ώστε τελικά να γίνεται μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση με τα πλεονεκτήματα και τα των διαφόρων τομέων σε σχέση με τις αντίστοιχες πρώτες που χρησιμοποιούμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μελίωρ. Όχι. Μου το μου δόθηκε απάντηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ναι, εμένα με ικανοποιεί η κυκλική οικονομία. Κύριε Πίτρο Πεβέλα, τη γεωργία. Εδώ αναφέρεται πράγματα από το 2003. Αν Αναφέρθηκε και ο συνάδελφο πριν ότι πολλέ φορέ έχουμε ρωτήσει και στον Επιτρόπο Χόγκαν όσον αφορά την, ε, τα οργανικά λοιπάσματα και τα... για την Ολλανδία είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα των ε, λοιπασμάτων και όχι μόνο τα φωσφορικά. Τελικά, η συγκεκριμένη μου ερώτηση είναι, μπορείτε όσο γίνεται πιο γρήγορα να μας πείτε περισσότερο όσον αφορά την γεωργία και για τα πόβλητα και την ανακύκλωση. Το 10% όμως θα πρέπει να καίγεται, έτσι δεν είναι. Πρέπει να γίνει αυτό. Δεν είναι δυνατό να μην το κάνετε. Τέλος. Για τα πλαστικά απόβλητα. Υπάρχουν μεγάλες επιχειρήσεις που ασχολούνται με αυτά. Μην είμαστε τόσο αρνητικοί. Υπάρχουν επιχειρήσεις που ασχολούνται ακριβώς με την αφαίρεση των ε, πλαστικών. Οπότε, καλό θα ήταν να μάθουμε περισσότερο πώς θα αγοράζουμε και πώς θα μαγειρεύουμε. Είναι προτιμότερο αυτό γιατί νομίζω ότι έτσι μπορούμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα και να μην πετάμε τρόφιμα. Μπορούμε να πετύχουμε πολλά έτσι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Σελίμωβιτς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε που ήρθατε και που μας προτείνατε μας εξηγήσετε τις προτάσεις σας. Συμφωνώ με όλοι ότι πρόκειται για μια απαραίτητη δέσμη. Κάποιοι εξημών όμως και μου συμπεριλαμβανομένου θεωρούν ότι δεν αρκούν και ότι είναι αρκετά, είναι μάλλον ασαφή αυτά που μας λέτε. Αλλά κυρίως αυτό που δεν βλέπω είναι μια ευρωπαϊκή προοπτική σε αυτή τη δέσμη. Δηλαδή όλοι αντιλαμβανόμαστε πιστεύω ότι αν θέλουμε να έχουμε αξιόπιστη κυκλική οικονομία με τις προτάσεις θα πρέπει το φάσμα, δηλαδή η κλίμακα της οικονομίας να αξιοποιηθεί, δηλαδή τα απόβλητα σε μια χώρα η ενέργεια, ε, να μετατραπούν σε ενέργεια ή σε υλικό που θα αξιοποιηθεί και σε μια άλλη χώρα. Αν δεν ανοίξουμε λοιπόν το γεωγραφικό πεδίο της Ευρώπης, χάνουμε κάθε πλεονέκτημα. Συγκεκριμένο παράδειγμα. Δεν έχει νόημα να μετατρέπουμε τα απόβλητα σε ενέργεια αν δεν μπορούμε να τα μεταφέρουμε σε κάποια άλλη περιοχή. Δεν υπάρχει λόγος να παράγονται ηλεκτρικά αυτοκίνητα στο Βέλγιο εάν μόνο στο Βέλγιο μπορούν να φορτιστούν. Δεν έχει νόημα να παράγεται ολική ενέργεια στην Ισπανία εάν η Γαλλία παρεμποδίζει τη μεταφορά της και χρήση στη δική της επικράτεια. Ερωτώ λοιπόν, πού είναι η ευρωπαϊκή προοπτική αυτής της δέσμης και πώς μπορείτε να ανοίξετε αυτό το πεδίο εφαρμογής, αυτό το ευρωπαϊκό γεωγραφικό πεδίο προ όφελο των ε, χωρών, αλλά όλων των χωρών. Ευχαριστώ πολύ Πέταρλε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ για την παρουσίαση, για τι απαντήσει σας. Σε ένα βαθμό έχετε δώσει απαντήσει σε ερωτήσεις μου. Αλλά πρέπει να πω πως ε, λυπούμε γιατί δεν βλέπω να έχουν ε, τηρηθεί ούτε καν τα επίπεδα της προηγούμενης πρότασης για την ανακύκλωση. Για το 70% στα δημοτικά ε, απόβλητα που έχει πέσει στα 65%, τα συσκευασίες από 80% πέφτει στο 75%, τα τρόφιμα ε, χάνονται τελείως τα ποσοστά για το 2025. Άρα η λέξη ρεαλισμός φαίνεται να προβάλλεται ιδιαίτερα, αλλά δεν νομίζω ότι ρεαλισμός σημαίνει κάνω λιγότερα. Τι λέτε λοιπόν εσείς, η φιλοδοξία μπορεί να είναι και ελκυστική και μπορούμε να το επιτύχουμε αυτό και αυτό ισχύει και για την πολιτική για τις κλιματικές αλλαγές. Δεν θέλω να έχω διδακτικό ύφος, αλλά θα υπενθυμίσω ότι την ίδια συζήτηση είχαμε και στην Ιαπωνία πριν από χρόνια για το τι είναι ε, ρεαλιστικό και τι μπορεί να είναι φιλόδοξο. Όταν η Ιαπωνία όμως εισήγαγε πιο υψηλούς ε, περιβαλλοντικούς στόχους, επέτρεψε στην οικονομία της να γίνει πιο ανταγωνιστική. Και ελπίζω να μπορέσουμε να κάνουμε το ίδιο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πίτροπα. Και χρόνια πολλά και σε εσάς μια και μας Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο. Ολοκληρώσαμε. Μπορούμε να σα ακούσουμε τώρα. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο κύριο Βέλλα. Πρώτα απ' όλα, για τα πλαστικά και, την, ε, και τα απόβλητα από πλαστικά. Εδώ ακριβώς βλέπουμε την κυκλική οικονομία. Εάν θέλουμε να μειώσουμε τα απόβλητα, δηλαδή πλαστικά στους ωκεανούς ή μετατροπή των αποβλήτων σε ενέργεια ή μια ανακυκλημένα υλικά που μπορούν να οδηγήσουν σε ενέργεια. Στην πρώτη ερώτηση αναφέρθηκε η οδηγία για τη μεταφορά αποβλήτων. Συμφωνώ απολύτως ότι είναι ενεργητικό και όχι παθητικό πια τα απόβλητα. Κάποτε λέγαμε ότι όσο πιο πολλά τα απόβλητα τόσο πιο μεγάλο το παθητικό. Τώρα συμβαίνει το αντίστροφο και δεν πρέπει να συνεχίσουμε να χάνουμε πόρους, όπως είναι ακριβώς τα απόβλητα. Γιατί μπορούμε να τα ξαναχρησιμοποιήσουμε. Να τα χρησιμοποιήσει ο δικός μας βιομηχανικός τομέας για να ενισχύσουμε και την ανταγωνιστικότητά μας. Για τον κύριο Γρότε που μίλησε για την προγραμματισμένη παλαίωση. Συμφωνώ μαζί του. Θα μπορέσουμε να καταλήξουμε ασφαλώς σε συγκεκριμένες προτάσεις για την προγραμματισμένη παλαίωση που αναφέρεται σε μια σειρά από τομείς, όχι μόνο ηλεκτρικές συσκευές, αλλά και υπολογιστές, τηλέφωνα και πολλά άλλα. Επίσης ο κύριος Κρότε αναφέρθηκε στην ανάγκη να αντιμετωπίσουμε σοβαρότητα όλα αυτά τα πράγματα. Με βεβαίω και το πράττουμε σοβαρότητα. Η Μάρε, επί παραδείγματι, και η Διευθυνσή Θαλασσών, όταν κοιτάει πώς μπορούμε να διαχειριστούμε καλύτερα τους ωκεανούς μας ε, και τις θάλασσες, που είναι το ίμιση περίπου των ωκεανών και θαλασσών της Ιφιλίου. Όλοι μας μας υπεύθυνοι. Και τελικά κανείς όμως αυτή τη στιγμή. Αυτό πρέπει να αλλάξουμε. Θα πρέπει βεβαίως να, αποφύγουν και, να αποφεύγεται σε πρώτο βαθμό η απόρριψη αποβλήτων στη θάλασσα. Έτσι θα βελτιωθεί η κατάσταση. Αναφέρεστε επίση στην οδηγία για τα, για τα λοιπάσματα. Όταν μιλούμε για την γεωργία στην κυκλική οικονομία ή κυκλική οικονομία στη γεωργία, υπάρχει ένας πολύ σημαντικός σύνδεσμος τώρα που έχουμε περάσει, ιδιαίτερα στην επαναχρησιμοποίηση των υδάτων και ανακύκλωση των υδάτων. Πρέπει να ξέρουμε ότι το, είδος, το είδωρ χρησιμοποιείται ως πόρος και ανακυκλείται στην οικονομία, στην ε, γεωργία. Και αναζητούμε όλο και πιο καινοτόμους τρόπους για καλύτερη χρήση και ανακύκλυση του ύδατος. Δεν κατάλαβα τι είπε ο κύριος Φλάναγκα ναι, σε σχέση με την οργάνωση μιας συνεδρίασης, αλλά όταν λέτε ότι δεν το συζητάει ο κόσμος, μα δεν είναι αυτό δεν είναι ότι το συζητάνε μόνο, είναι ότι επενδύουν οι επενδυτές. Αυτό είναι κυκλική οικονομία. Έχουμε τον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος τρέχει παρασάγκας μπροστά μας, καινοτομή, και αυτή τουλάχιστον είναι η δική μας ιδέα για τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να υποστηρίξουμε την κατάσταση, δηλαδή να στηρίξουμε τον ιδιωτικό τομέα, γιατί τελικά αυτός θα είναι ο υπεύθυνο για την εξασφάλιση των πλεονεκτημάτων, των αποτελεσμάτων αυτής της κυκλικής οικονομίας. Και επίσης είχα αναφέρει νομίζω και τα δισεκατομμύρια που ήδη έχει ρίξει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στη χρηματοδότηση ε, έργων κυκλικής οικονομίας. Ναι, δεν το, δεν το συζητούμε μόνο, δεν περιοριζόμαστε στα λόγια. Υπάρχουν ήδη οι δράσει, υπάρχουν όλοι αυτοί που το έχουν υλοποιήσει και το υλοποιούν και χρειάζονται την υποστήριξή μα. Θέσει εργασία, ανταγωνιστικότητα, φιλοδοξίε. Βεβαίω. φιλοδοξία. Τι είναι. Ακούμε τι έχει να μα πει το Κοινοβούλιο, ακούμε τι έχει να μα πει το Συμβούλιο, αλλά κοιτούμε και άλλου σημαντικού φορεί. Γιατί εάν κοιτάξουμε την κυκλική οικονομία από την οικονομική της διάσταση, οφείλουμε να ακούσουμε τι έχει να πει ιδιωτικός τομέα και από την περιβολητική διάσταση οφείλουμε να ακούσουμε και τι έχουν να πούν και τα κράτη-μέλη για τον κύριο Χόισλιν προς όφελος οικονομίας. Ναι, δεν θα επαναλάβω τη σημασία του ιδιωτικού τομέα, γκαρντίνη, ολιστική προσέγγιση. Ναι, βεβαίως και έχουμε μια ολιστική προσέγγιση. Γι' αυτό και ανοίγουμε το πεδίο η κυκλική οικονομία είχε ξεκινήσει με το πλαστικό, το χαρτί, το γυαλί. Τώρα πάμε σε ολόκληρη την οικονομία, στην οικοδομική, στα, στην φαντουργία, στα πάντα. Μίλησα για συνδέσμους. Ένα από τα κύρια ε, πλεονεκτήματα που δεν ανέφερα στο σημείο αυτό ήταν ότι είναι μικρότερο το κόστος σε ενέργεια για την επεξεργασία στην ανακύκλωση. Ένα παράδειγμα από το αλουμίνιο. Χρειάζεται δεκαπλάσιο χρόνο η επεξεργασία του ε, παρθένου λεγόμενου αλουμινίου, δηλαδή η πρώτη επεξεργασία παρά η ανακύκλωση του. Αυτό μας δείχνει πόσο σημαντικό είναι το ε, συγκριτικό πλεονέκτημα. Επίσης μίλησε ήδη για τα οδηγία για τα λοιπάσματα, είπαμε ότι θα γίνει αναθεώρηση των κανονισμών για τα λοιπάσματα, πλαστικά και απόβλητα θαλασσών. Και μάλιστα δεν ξέρω και γιατί να τα λέμε απόβλητα θαλασσών, γιατί είναι στερεά, στερεάς μάλλον απόβλητα, από τη στεριά δηλαδή φεύγουν και πάνε στη θάλασσα, άρα στη στεριά πρέπει να γυρίσουν. Θέλω επίσης να τονίσω ότι όλες οι περιβαλλοντικές ε, προκλήσεις έχουν σημασία όχι μόνο για περιβαλλοντικό λόγο. Είναι προκλήσεις ως προς το περιβάλλον που ταυτόχρονα μπορούν να μας προσφέρουν οικονομικές, ε, οικονομικά ωφέλη ή ευκαιρίες. Πρέπει βεβαίω να συνοηθούμε και να εξηγήσουμε και στον καταναλωτή η σήμανση, η επισήμανση παραδείγματι, η οικολογική επισήμανση, διάφοροι τρόποι που θα επιτρέψουν στον καταναλωτή να αντιλαμβάνεται καλύτερα τι επιλογέ του. Απόβλητα σε ενέργεια, ναι βεβαίω μια πρόκληση που έχουμε και σε σχέση με την παλιριακή ενέργεια για την εναρία των κυμάτων. Αυτά θα πρέπει να τα δούμε, γιατί χρειάζεται η ανάπτυξη των υποδομών που θα, επιτρέπουν τη μετάδοση, μεταφορά αυτή τη ενέργεια. Βέβαια, μπορούν κάποια κράτη-μέλη ήδη να διαθέσουν την ενέργεια που παράγουν στα υφιστάμενα δίκτυα διανομή. Για τον κύριο Πέτερλε δεν νομίζω ότι μειώσαμε τους στόχους για τα ανακυκλωμένα υλικά. Αυτό που πράξαμε όμως, και είναι πιο σημαντικό για μένα, ε, ήταν ότι μειώσαμε τους στόχους στην παραγωγή αποβλήτων. Και συγκρίνουμε τώρα τους στόχους ως προς τους όγκους των υποανακύκλησης υλικών, λησμονώντας όμως ότι η κυκλική οικονομία περισσότερο ακόμη στηρίζεται στην μείωση των στόχων παραγωγής αποβλήτων σε πρώτο επίπεδο. Και βέβαια, οι στόχοι που υποστηρίζουμε δεν είναι του μόνο. Έχουμε και σχέδια, έχουμε και οικονομική υποστήριξη. Σας ευχαριστώ και πάλι καλά σας Χριστούγεννα. Και λυπούμε, αλλά πρέπει να φύγω πολύ γρήγορα. Uh, ευχαριστούμε πολύ. Ξέρουμε ότι πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε, αλλά συνεχίζουμε την συνεδρίασή μας. Δεν έχει ζητήσει κανείς άλλος το λόγο. Να ευχαριστήσουμε τον Επίτροπο που βρέθηκε εδώ μαζί μας και που απάντησε σε πάρα πολλές ερωτήσεις για πάρα πολλή ώρα. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερως. Dear colleagues, we can... Αγαπητοί συνάδελφοι, μπορούμε να συνεχίσουμε τώρα κάνοντας ένα βήμα προς τα πίσω, προς το σημείο 3 τη ημερήσιας διάταξη, Είναι η υποβολή έκθεση ε, σχετικά με τις τρέχουσες διοργανικές διαπραγματεύσεις για τους ελέγχους και λοιπές δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής νομοθεσία για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές ο πρώτος και δεύτερος τριμερής διάλογος που έλαβαν χώρα ε, στις 9 Νοεμβρίου πιο συγκεκριμένα έδωσαν στους νομοθέτη τη δυνατότητα να συζητήσει σημεία για τα οποία υπάρχουν ήδη συγκλίνουσες θέσεις όπως ε, το πολλαπλασιαστικό φυτικό υλικό, ώστε να αποφασιστεί η μεθόδος εργασίας και το χρονοδιάγραμμα και το, η πρώτη ομάδα άρθρων. 16 Δεκεμβρίου έγινε ο πρώτος τριμερής διάλογος και αυτό έδωσε δυνατότητα στους νομοθέτη να συζητήσει τις διατάξεις για τους ελέγχους σε συγκεκριμένους τομείς και να συμπεριληφθούν τα διατάξει στην βασική δευτερεύουσα νομοθεσία. Ο τέταρτος τριμερής διάλογο προγραμματίζεται για τις 27 Ιανουαρίου. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, στο σημείο 5. 5 και 6 τα οποία μπορούμε να συζητήσουμε μαζί αφορούν την αποδοχή των τροποποιήσεων του πρωτοκόλου του 1998 της Σύμβασης του 1979 για την διασυνοριακή ατμοσφαιρική ρήπανση μεγάλης απόστασης που οφείλεται στους μόνους οργανικούς ρήπους είναι στο σημείο 5 και στα βαρέα μέτρα είναι στο σημείο 6 οπότε θα περάσω στα Ιταλικά και είναι πολύ πιο εύκολο για μένα είναι πολύ πιο απλά να τα εξηγήσω στα Ιταλικά. Λοιπόν, η σύμβαση αυτή για την διασυνοριακή ατμοσφαιρική ρήπαχη σε μεγάλη απόσταση αποσκοπεί στην προστασία του περιβάλλοντος από τη ρήπανση. Είναι μια μακροχρόνια διαδικασία που ξεκίνησε βάσει μελετών που έγιναν από το 1972 μέχρι το 1977 και που οδήγησαν την ε, σύνευση της σύμβασης που συζητάμε που υπογράφηκε το 1979 και τέθηκε σε ισχύ το 1983. Υπήρξε αυτή το πρώτο διεθνές νομικά δισμευτικό μέσο για τον τομέα αυτών. Αυτή η σύμβαση δημιουργεί ένα πλαίσιο για τον έλεγχο και τη μείωση των βλαβών από τη διασυνοριακή ρήπανση. Ακολουθήθηκε από 8 πρωτόκολλα τα οποία αφορούν θιούχες ε, εκπομπές, επτητικές οργανικές ενώσεις, βαρέα μέταλλα και το 8ο πρωτοκόλλο ε, αντιμετωπίζει την ε, οξύνηση, το τροποσφαιρικό όζον και τον ευτροφισμό και το επόμενο πρωτόκολλο αφορά τους έμονους ε, ε, ρήπους ε, και που τροποποιήθηκε με πρωτόκολλο από την Κομισιόν. Εξετάστηκε η καταλληλότητα και η αποτελεσματικότητα των υποχρέωσεων που προβλέπεται και το 2007 άνοιξαν οι διαπραγματεύσεις για αναθεώρηση του κειμένου και των σχετικών τροπολογιών. Το πρωτόκολλο τροποποιήθηκε με αποφάσεις του 2009 και οι αποφάσεις αυτές πρέπει να αποκηρυθούν από τα συμβαλόμενα μέρη επικύρωση των τροπολογιών που διατυπώθηκαν με αποφάσεις του Συμβουλίου θα αποτελεί σημαντικό βήμα μπροστά προς ένα υψηλότερο επίπεδο προστασίας ε, της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από τη διασυνοριακή ατμοσφαιρική ρήπανση. Τόσο όσον αφορά τους οργανικούς ρήπους ε, αλλά και όσον αφορά τα βαρέα μέταλλα η πρόταση του εισηγητή είναι να εγκρίνουμε τις τροπολογίες που έχουν πραγματοποιηθεί μέσω απόφαση του Συμβουλίου και έτσι να δώσουμε τη συνένεσή μας τόσο για το σημείο 5 όσο και για το σημείο 6 της ημερήσης διάταξης. Υπάρχει κάποιος που θα ήθελε το λόγο. Κανένας δεν θέλει να σχολιάσει. Ωραία, ας δώσουμε το λόγο λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι. Συμφωνούμε άπαντες. Πολύ ωραία. Ας προχωρήσουμε λοιπόν ώστε να ανακτήσουμε το χαμένο χρόνο, το χρόνο που χάσαμε με το προηγούμενο σημείο. Λοιπόν, περνάμε. Λοιπόν, Τώρα πρέπει να ακολουθήσει κοινή συζήτηση για τα σημεία 7, και 9. Πρόκειται για ενστάσεις ε, σύμφωνα με το άρθρο 105 του κανονισμού για τα παρασκευάσματα για βρέφη και παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικία για... στο σημείο 7. Αλλά όπως φαίνεται ο συνάδελφος που διατύπωσε την ένσταση δεν είναι παρόν. Αλλά έρχεται. Οπότε σας προτείνω να συζητήσουμε πρώτα τα σημεία 10 με 15 που αφορούν την απαλλαγή. Οπότε να κάνουμε λίγο δουλειά. Uh, λοιπόν, ο συνάδελφος, μέχρι να έρθει ο συνάδελφος Τέιλορ, α ασχοληθούμε με τα σημεία τη απαλλαγή του 2014, τη ΕΦΣΑ, τη ΕΚΑ, της ΕΑ, τη ΕΣΥΔΙΣΗ... Τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων. 10 με 15 είναι τα σημεία αυτά στην ημερήσια διάταξη. Ξεκινάμε λοιπόν με κάποιες γενικές πτυχές, δεδομένου ότι και εγώ είμαι εισήγητη ε, τη γνωμοδότησης, οπότε θα με ακούσετε λιγάκι. Λοιπόν, σε γενικέ γραμμές θα έλεγα ότι αυτή η εξέταση τη εκτέλεσης και του προπολογισμού λαμβάνει υπόψη την ετήσια έκθεση του ερευνητικού Συνεδρίου και των επαφών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των λοιπόν θεσμικών οργάνων που συνεργάστηκαν με το Κοινοβούλιο και που έδωσαν ικανοποιητικέ απαντήσεις στα δικά μα αιτήματα ενημέρωσης και διευκρινήσεων. Να υπενθυμίσω ότι το 2014 έτος που αφορά αυτές οι απαλλαγές ήταν το πρώτο έτος εφαρμογής του νέου δημοσιονομικού, πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου το οποίο είχε ως στόχο την κατανομή των πόρων της Ένωσης ε, για το διάστημα 2014-2020. Το επίπεδο εκτέλεσης λοιπόν, επειδή ήταν το πρώτο έτος του πολίτου δημοσιονομικού πλαισίου, ήταν χαμηλότερο από ότι τα προηγούμενα έτη, παρότι πολύ ψηλό για ζητήματα που αφορούν τις δικές μας αρμοδιότητες. Πράγματι, η Γενική Διεθνής Περιβάλλοντος από τα 352 εκατομμύρια ευρώ δεσμευτικών ε, ε, πιστώσεων ε, είχε εκτέλεση 99,7 και οι πιστώσεις, πιστώσεις πληρωμών 99,2%. Το ποσοστό εκτέλεσης αυξήθηκε και όσον αφορά την DG Κλίμα με ποσοστό 99,7% όσον αφορά τις αναλήψεις περιεχομένων και 93,1% για τις ε, πιστώσεις πληρωμών. Όσον αφορά τη Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΤΕ, ήταν αρμόδια το 2014 για την υλοποίηση 244 εκατομμυρίων ευρώ για τη δημόσια υγεία. 95% ε, εκτελέστηκε ικανοποιητικά. Το 75% του προπολογισμού ε, δόθηκε σε αποκεντρωμένες ε, ε, οργανισμούς και το επίπεδο εκτέλεσης έφτασε το 98%. Απόλυτη λοιπόν ικανοποίηση εκ μέρους του εισηγητή όσον αφορά τα επίπεδα ανάληψη υποχρεώσεων και πληρωμών στα θέματα που αφορούν την ε, Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, τη Γενική Διεύθυνση Κλίματος και τη Γενική Διεύθυνση Υγείας. Τώρα, όσον αφορά την διατροφική ασφάλεια και κυρίως ε, τους ε, οργανισμούς όπου θα σταθώ, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι πολύ σημαντικό ρόλο ανέλαβαν για τεχνικά και επιστημονικά και διοικητικά καθήκοντα. Οι οργανισμοί αυτοί βοηθούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των σχετικών πολιτικών. Απαιτούν ανθρώπινους πόρους και οικονομικούς πόρους για να επιτύχουν τους στόχους. Βλέπουμε γενική βελτίωση της ε, κατάστασης του προϋπολογισμού. Εισήχθηκαν διορθωτικά μέτρα μετά από τις παρατηρήσεις του Κοινοβουλίου και του Ελεκτικού Συνεδρίου τα προηγούμενα έτη με ειδικότερη αναφορά στην αυτο, γενική αυτοαξιολόγηση και στη βελτίωση των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και των ετήσιων προγραμμάτων εργασιών με περισσότερη ανάλυση των δημοσίων διαγωνισμών και των επιχορηγήσεων. Το ίδιο ισχύει όσον αφορά την παρατήρηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την απολογή του 2013 που αφορούσε τους τομείς όπου οι που αφορούσαν τους οικονομικούς ελέγχους και όπου αναφερόμενοι στην ΕΦΣΑ η εσωτερική έλεγχη και το σύστημα ε, που αφορούσε τους εσωτερικούς εμπειρογνώμονες. Θεωρώ λοιπόν ότι βάσει των διαθέσιμων στοιχείων της έκθεσης του ελεκτικού συνεδρίου μπορεί να χορηγηθεί η απαλλαγή στην Επιτροπή όσον αφορά τις δαπάνες του τομείς της περιβαλλοντικής κλιματολογικής πολιτικής, πολιτικής δημόσιας υγείας και ασφάλειας των τροφίμων για το 2014 καθώς και στους πέντε οργανισμούς που εντάσσονται στην πέντε αρμοδιοτητών της Επιτροπής μας. Οι γνωμοδοτήσεις λοιπόν που έχουν συνταχθεί εδώ εκφράζουν μια θετική άποψη όσον αφορά την ε, χορήγηση της απαλλαγής. Μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση και δίνω αμέσω το λόγο στον συνάδελφο Σελίμωβιτς που την ζήτησε. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σύμφωνο με όλα όσα αναφέρονται στις νομοδοτήσεις, τις διάβασα προσεκτικά. Και όταν προσπαθούσαμε να κάνουμε την τελευταία τροπολογία, είχε πέσει το σύστημα. Οπότε θα προσπαθήσω τώρα να πω κάτι που πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό. Είτε προφορικά, είτε το χρόνου, δεν ξέρω, αλλά πάντως αξίζει τον κόπο να το αναφέρουμε. Και όλους αυτούς τους οργανισμούς, τους πέντε. Όλοι έχουν πολιτικές καταπολέμησης της ε, διαφθοράς και της απάτης. Οι υπόλοιποι όμως δεν το έχουν αυτό. Και εφόσον το λεκτικό συνέδριο το λέει, λέει ότι κάπου υπήρξαν κάποιες ε, παρατυπίες, θα μπορούσαμε να συστήσουμε η Επιτροπή μας δηλαδή να γνωμοδοτήσει προς αυτή την κατεύθυνση, ότι συστήνουμε να υπάρχουν πολιτικές κατά των απατών. Σε ορισμένους από αυτούς τους οργανισμούς, όπως σας είπα, υπάρχει ε, στους άλλους θα έπρεπε να υπάρχει. Δεν ξέρω αν είναι εφικτό. Σας λέω, όταν προσπαθήσαμε να υποβάλουμε τέτοια τροπολογία έπεσε το σύστημα και δεν το κάναμε. Ζητώ συγγνώμη. Αν δεν γίνεται φέτος να το κάνουμε, να το κάνουμε του χρόνου. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να το λέμε. Πρέπει να υπογραμμίσω εδώ, λέει ο Πρόεδρος, ότι μέχρι αύριο στις 12 το μεσημέρι μπορεί να υποβληθεί η τροπολογία. Με τη συνήθη διαδικασία λοιπόν ε, μπορείτε να υποβάλλετε την τροπολογία αυτή και θα ψηφίσουμε αργότερα στην Επιτροπή μας. Άλλος κανείς θέλει το λόγο για αυτό το θέμα. Όχι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακαλώ αν είναι εδώ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Απλώς θέλω να πω ότι μας ικανοποιεί η χρήση 2014 όσον αφορά το περιβάλλον και το κλίμα. Και όπως είπατε και εσείς δεν ήταν μια εύκολη χρονιά. Ήταν η πρώτη χρονιά που είχαμε τις νέες δημοσιονομικές προοπτικές, το νέο πολιετές δηλαδή δημοσιονομικό πλαίσιο, με κάποιες καινοτομίες. Ιδιαίτερα υπήρχαν οικονομικά μέσα νέα για το περιβάλλον ένα, για το κλίμα το άλλο και τα οικονομικά αυτά μέσα ξεκίνησαν ε, τώρα. Μας ικανοποιεί επίσης η χρήση προπολογισμού όσον αφορά την Γενική Διεύθυνση Κλίμα. Είναι μια Γενική Διεύθυνση που δημιουργήθηκε το 2010. Τώρα, το 2014, έχει φτάσει στην κανονική της ταχύτητα, με ένα ποσοστό χρήσης κανονικό. Η αρχή ήταν κάπως δύσκολη βέβαια όσον αφορά τη χρήση των κονδυλίων, αλλά τώρα νομίζω ότι πάει πολύ καλύτερα. Το 2014 ήταν μια χρονιά που μας ε, δυσκόλεψε και όσον αφορά τις πιστώσεις πληρωμών και χρειάστηκε να γίνουν διάφορες μεταφορές το 2015. Έγιναν όμως αυτές τον Ιανουάριο του 2015 πληρωμές. Τώρα η κατάσταση έχει τακτοποιηθεί. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλα σχόλια από κάποιον άλλον, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όχι, καλώς. Συνεχίζουμε λοιπόν και πάμε πίσω πάλι Υπενθυμίζω ότι η προθεσμία για τροπολογίες είναι αύριο στις 12 το μεσημέρι. Θα ψηφίσουμε στις 21 Ιανουαρίου. 23 Μαρτίου εικόνου. Τώρα, είδα κάπου τον κύριο Τέιλορ. Ήρθε. Καλώς. Οπότε πάμε πίσω στη γενική συζήτηση όσον αφορά τις ενστάσεις πέντε υπάρχουν για τα τρόφιμα, φάρμακα, ε, βρεφικές τροφές και η τρίτη έχει να κάνει για δημητριακά και βρεφικές τροφές. Για εξηγήστε μας παρακαλώ κύριε Τέιλορ τις ενστάσεις σας και μετά θα αρχίσουμε τη συζήτηση. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα αναφερθώ και στις τρεις ε, ενστάσεις μαζί. Με τη σειρά βέβαια που υπάρχουν στην ημερήσια διάταξη. Πρώτα απ' όλα θέλω να αποσαφηνίσω ότι παρόλο που υπάρχουν αυτές οι ενστάσεις, οι φρεβικές στροφές είναι ο καλύτερος τρόπος για να τρέφονται τα βρέφη. Εγώ με τίποτα δεν είμαι κατά του μπιμπερό αντί για τον θυλασμό. Το σέβομαι απόλυτα. Αλλά οι ενστάσεις αυτές τις υποβάλλω για να προστατεύσω τα παιδιά και εκείνα που θυλάσσονται και εκείνα που παίρνουν γάλα με μπιβερό. Θέλω να προστατεύσω και αυτά τα παιδιά και τους γονείς από εμπορικές πρακτικές και παραπληροφόρηση από τις διαφημίσεις. τους πρώτους έξι μήνες μπορούν τα παιδιά να τρέφονται με θυλασμό και από τους έξι μήνες και μετά μπορούν να προσθεθούν και άλλες ουσίες συμπληρωματικά δηλαδή συστατικά στο γάλα. Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι από τις 21 χώρες στον ΠΟΕ μόνο 13% των μωρών τρέφονται αποκλειστικά από τον θυλασμό στους έξι μήνες. Ο θυλασμός σίγουρα έχει πάρα πολλά ωφέλη για τα παιδιά και για τις μητέρες τους και θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει περισσότερα για να ενθαρρύνει την πρακτική αυτή. Δυστυχώς όμως ο σχετικός κανονισμός δεν το κάνει. Δεν περιλαμβάνει τίποτα για να αποφευθεί ο αθέμητος ανταγωνισμός απέναντι στο θυλασμό. Η διεθνή διοντολογία όσον αφορά τα υποκατάστατα του ΠΟΕ λοιπόν είναι κάτι που υπάρχει και πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Η ρύθμιση όμως ε, αυτή που έχουμε τώρα δεν ενισχύει αυτή τη ρύθμιση αλλά την αποδυναμώνει και δεν φροντίζει οι χώρες μέλη να προστατεύουν, να θαρρύνουν το θυλασμό και να προστατεύουν τα παιδιά και τις μητέρες. Ενώ ο Διεθνής Κώδικας λέει ότι δεν πρέπει να γίνονται διαφημίσεις ή με άλλο τρόπο να προωθείτε προς το κοινό κάτι που να είναι εκτός του κώδικα. Παρόλα αυτά, εδώ με το σχέδιο αυτό κανονισμού επιτρέπεται η διαφήμιση ενώ θα έπρεπε οι χώρες μέλη να απαγορεύουν να περιορίζουν τέτοια διαφήμιση. Δεν περιορίζει επίσης την διαφήμιση υποκαταστάτων. Ούτε ενθαρρύνει τις χώρες οι οποίες θέλουν να απαγορεύσουν ε, τέτοιου είδους διαφημίσεις. Γι' αυτό λοιπόν εγώ λέω ότι κάθε ε, διαφήμιση για προϊόντα που αντικαθιστούν τον οθυλασμό πρέπει να περιορίζεται σε δημοσιεύσεις που περιλαμβάνονται μόνο σε περιοδικά που είναι ειδικευμένα και επιστημονικά για το θέμα αυτό. Αλλιώς πρέπει να περιορίζονται, να απαγορεύονται οι διαφημίσεις για τέτοια προϊόντα. Οι ισχυρισμοί επίσης που γίνονται για τα ωφέλη από τέτοια προϊόντα πρέπει επίσης να περιορίζονται. Τέτοιοι ισχυρισμοί πρέπει να επιτρέπονται μόνο εφόσον η Επιτροπή τους επιτρέπει και ο κανονισμός 1925 για τα παρασκευάσματα δεύτερης βρεθικής τροφής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν εξετάζει την άδεια για τέτοια προϊόντα. Είτε πρόκειται για την βιταμίνη σε που λέει ότι βοηθάει την απορρόφηση νεόλων προϊόντων. Όλοι οι ισχυρισμοί μπορεί να είναι σωστοί, αλλά αν επιτρέπουμε να γίνονται διαφημίσεις για αυτά τα χαρακτηριστικά όσον αφορά τις, ε, τα βρεφικά αυτά παρασκευάσματα, αυτό είναι διαφήμιση και θα έπρεπε να εμποδίζονται. γιατί υπονομεύουν το θυλασμό. Εγώ πιστεύω ότι η Επιτροπή μας θα πρέπει να στήσει να απαγορεύονται τέτοιες διαφημίσεις και τέτοιοι ισχυρισμοί. Άλλες αιτίες που μας οδηγούν στο να πρέπει να αποφεύγουμε τέτοια διαφήμιση είναι το DHA που είναι ένα λιπαρό οξύ ωμέγα 3 που περιλαμβάνεται στο βρεφικό γάλα σε θελοντική βάση. Τα ωφέλη δεν έχουν αποδειχτεί. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν διαφημίσεις με ισχυρισμού ότι είναι προς όφελος των βρεφών. Τέτοια πράγματα είναι που θέλουμε να απαγορεύσουμε. Και τέλος, υπολείμματα από παριστοκτόνα ή άλλες ε, τέτοιες ουσίες δεν πρέπει να υπάρχουν καθόλου 0% ανοχή. Θέλουμε να απαγορευτούν τέτοια προϊόντα. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Είναι, όπως ε, καταλαβαίνετε, για την ασφάλεια των βρεφών Το δεύτερο θέμα περιλαμβάνει κάτι και για ιατρικούς λόγους. Ο λόγος που έχω αντίρρηση για τα τρόφιμα για ιατρικούς λόγους έχουν να κάνουν με τις ε, απαιτήσεις όσον αφορά τη διατροφή των βρεφών είναι ευάλωτη ομάδα. Η διαφήμιση λοιπόν ειδικών ε, φαρμάκων για αυτά δεν θα έπρεπε να επιτρέπεται. Πρέπει να περιοριστεί μόνο στον επιστημονικό κόσμο και να αναφέρονται μόνο στοιχεία. Επιτρέπεται όμως η διαφήμιση για προϊόντα ιατρικούς λόγους για τα βρέφη. οι έγκυοι, οι μητέρες, οι πατεράδες, οι νέοι γονείς μπορεί να παρασυρθούν και να προσπαθήσουν να διαγνώσουν από μόνοι τους κάποιο πρόβλημα υγείας που μπορεί να έχει το μωρό τους. Χρειάζεται λοιπόν περιορισμός τέτοιων διαφημίσεων και τέτοιων πρακτικών, κάτι που αναφέρεται στο άρθρο 10 του κατεξουσιοδότηση κανονισμού όσον αφορά τα προϊόντα αυτά. Όμως η διατύπωση κάνει μια διάκριση στο σημείο 18 του κατεξοδότηση κανονισμού. Ανάμεσα στην τροφή των βρεφών και την επόμενη όσον αφορά την απαγόρευση ή τον περιορισμό που το κάνει μόνο για τα βρέφη και όχι μετά. Εδώ δεν υπάρχει συνοχή, δηλαδή ανάμεσα στον κατεξουσδότηση κανονισμό και την διατύπωση εδώ που μπορεί να οδηγήσει σε παρεξηγήσεις. Ένας άλλος λόγος για τον οποίο έχω την αίσθηση είναι ότι ενώ το, ο κατεξοδότης κανονισμού δεν επιτρέπει ισχυρισμούς για τα ωφέλη, διάφορες μάρκες de facto χρησιμοποιούν τέτοιους ισχυρισμούς. Αυτός ο κανονισμός θα πρέπει να λέει ότι τα ονόματα των, από τις μάρκες δεν θα πρέπει να περιλαμβάνουν, υπονοούν τέτοιους ισχυρισμούς. Επίσης όσον αφορά τα υπόλοιπα παρεσιτοκτόνου σε όλες τις ε, τροφές για βρέφη πρέπει να απαγορευτούν τη στιγμή που πρόκειται για ευάλωτες ομάδες, τα βρέφη και τα μικρά παιδιά. Ελπίζω η Επιτροπή μας να το στηρίξει στην ψηφοφορία που θα γίνει τον Ιανουάριο. Τέλος. Έρχομαι στα επεξεργασμένα δημητριακά. Το τρίτο θέμα που έχουμε στον κατάλογο. Εδώ 30% της ενέργειας δίνεται με ζάχαρη που είναι 30%. Θα αναγνωρίσετε εδώ ότι σε αντίθεση με όλες τις συμβουλές που έχουμε από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας κλπ που θέλει να περιορίζονται σε λιγότερο από 10% οι ελεύθερες ζάχαρες, αν αυτό το συγκρίνεται με το σχέδιο κανονισμού που μιλάει για 30% επί 3 δηλαδή τη σύσταση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας καταλαβαίνετε ότι είναι υπερβολικό. Επίσης ο ΠΟΕ λέει ότι από 6 μήνες το μητρικό γάλα πρέπει να συμπληρώνεται με συμπληρώματα χωρίς όμως πρόσθετα άλατα και ζάχαρη. Οι επιστημονικές επιτροπές στις χώρες μέλη έχουν επίσης συστήσει σημαντική μείωση της ζάχαρης. Ζάχαρη σε τόσο νεαρή ηλικία οδηγεί σε παχυσαρκία, κάτι το οποίο πρέπει να αποφεύγεται. Ιδίω τα μικρά παιδιά η πρόσθετη ζάχαρη πρέπει να περιορίζεται όσο γίνεται περισσότερο. Η ζάχαρη είναι μαζί με το ενόπνευμα και την μη άσκηση είναι αυτά που οδηγούν στις περισσότερες περιπτώσεις θανάτου. Όμως στον κανονισμό αυτό το προτινόμενο δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία που να προστατεύουν την υγεία των ε, μικρών παιδιών και να βοηθούν να αποφεύγεται η αρκεία. Η περιεκτικότητα σε ζάχαρη θα έπρεπε να είναι όπως συστήνει ο ΠΟΕ και όχι παραπάνω. Εγώ ζητάω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καθυστερήσει την έγκριση της κατεξιδότησης αυτής της πράξης μέχρι να έχουμε περισσότερες δημοσιεύσεις και να περιμένουμε την ΕΦΣΑ να έχει δημοσιεύσει τα δικά της συμπεράσματα όσον αφορά τα επεξεργασμένα τρόφιμα που προορίζονται για μικρά παιδιά. Αλλαγές στην ένστασή μου μιλούν επίσης για την προσέγγιση 0% στα παρασιτοκτόνα, περιεκτικό σε παρασιτοκτόνα, δεδομένου ότι τα βρέφη και τα νεαρά παιδιά αποτελούν μια ευάλωτη ομάδα καταναλωτών. Η σήμανση επίσης των προϊόντων αυτών θα πρέπει να δείχνει ότι δεν είναι κατάλληλα για βρέφη κάτω των έξι μηνών. Αυτά. Να απορρίψετε λοιπόν αυτή την πρόταση κανονισμού. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ας αρχίσει η συζήτηση. Κύριε Γκροστέτ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Μου φαίνονται αβάσιμες να θα σας αυτέ αυτές οι τρεις αντιρρήσεις και θα σας εξηγήσω γιατί προτείνω να τις απορρίψουμε. Κατά την έγκριση του κανονισμού του 2012, πολλοί ήμασταν εκείνοι που είχαμε αγωνιστεί μαζί με διάφορους συναδέλφους, την κυρία Ρίσφερμπιν, ώστε να επιβληθούν υψηλές προδιαγραφές ασφάλειας τροφίμων για να προστατεύονται οι πιο ευάλωτοι, στους οποίους απευθύνονται τα προϊόντα αυτά. Η καταξιοδότηση πράξη τη Επιτροπή ε, τίνουν προ την καλύτερη ενημέρωση του καταναλωτή, την ενισχυμένη επισήμανση, τι πιο αυστηρέ απαγορεύσει προ τη διαφήμιση. Και φρονώ ότι τα μέτρα αυτά τίνουν προ την ορθή κατεύθυνση. Γι' αυτό και θα συμμεριζόμαι την ακραία θέση των πρασίνων για, τις, ε, για τα σκευάσματα πρώτης ηλικίας και τα ε, δεύτερης ηλικίας. Η θέση των πρασίνων σε σχέση με τον μητρικό θυλασμό με παραξενεύει και με ανησυχεί. Προοδευτική λένε ότι είναι οι πράσινοι, άρα υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών. Αλλά θέλουν να ε, δημιουργήσουν ενοχικά σύνδρομα σε όποια γυναίκα δεν θυλάζει και πολλές φορές δεν είναι σε θέση καν να θυλάζει το ε, βρέφος της. Απαράδεκτο αυτό. Βεβαίως και όλοι αναγνωρίζουμε την υπεροχή του μητρικού θυλασμού και του γάλακτος, αλλά πρέπει να προσφέρονται υγιείς και ασφαλείς εναλλακτικές στη διάθεση των μητέρων. Το να προσπαθούμε στο βαθμό αυτό, να, το προσπαθούν κάποιοι στο βαθμό αυτό να απαγορεύσουν την ε, διάθεση στην αγορά ε, ε, κατασκευασμάτων που αντικαθιστούν το μητρικό θυλασμό είναι πολύ επικίνδυνη. Ταυτόχρονα ισχυρίζεται ψευδός ότι δεν θα πρέπει να επιτρέπεται η ε, ενημέρωση. Είναι πολύ πιο περιορισμένη η ενημέρωση του παρακοκού για τα γάλατα αυτά τα ηλικία. Δεν μπορούν να ισχυριστούν δηλαδή ότι είναι καλύτερα από το μετρικό θυλισμό. Τα γαλάτα πρώτης και δεύτερης ηλικίας σαφώς διακρίνονται με ειδική επισήμανση ώστε να μπορεί να τα διαφοροποιεί ο καταναλωτής και με τις διατάξεις που προβλέπονται είναι νομίζω εγγυημένη η προστασία του καταναλωτή. Για δε τα τρόφιμα που απευθύνονται που αφορούν συγκεκριμένους ιατρικούς στόχους και παραγόνται με βάση τα σιτηρά ή τρόφιμα για ε, βρέφη, τα γκέρμπερ που λέμε, είναι νομίζω αβάσιμα τα επιχειρήματα. Ας δούμε λίγο τις αιτιολογικές σκέψεις και συγκρίνουμε με τα άρθρα. Εν ώψη των δύο αντιρρήσεων του συναδέλφου, η μηδενική ενοχή σε σχέση με την ε, περιεκτικότητα σε ζυζανιοκτώνα, που τώρα είναι πάρα πολύ χαμηλή, 0,01 το πολύ, μικρογραμμάρια ανακυλό και ισχύει για κάθε είδους ζυζανιοκτώνου και πρέπει να πω ότι δυστυχώς και μέσω του μυστηρικού θυλασμού θα μπορούσε μια μητέρα να μεταδώσει στο ε, βρέφος της ε, ζυζανιοκτώνα που ίδια θα είχε ενδεχομένω καταναλώσει με την τροφή της. Άρα η απόλυτη απαγόρευση θα ήταν και αδύνατο να υλοποιηθεί. Γιατί υπάρχουν κατάλοιπα ζυζανιοκτώνα στο περιβάλλον και σε που μπορούν να εμφανιστούν και, στην, και στα τρόφιμα. Είναι μη ρεαλιστικό λοιπόν να ζητούμε μηδενική ενοχή. Επίσης τα παρασκευάσματα με βάση ε, σιτηρά και τρόφιμα για βρέφη είναι ρυθμισμένα με περιορισμένο και το άλλες και τα α, πολυακόριστα και το, τα σάχαρα. Επίσης, για να ολοκληρώσω, από τις τρεις αυτές αντιρρήσεις αντιλαμβάνομαι ότι η διαδικασία της επιτροπολογίας ορθά επισημαίνεται πως δεν είναι πολύ σαφής. Πρέπει ωστόσο να Επισημάνουμε ότι οι κατεξουδότησες πράξεις προχωρούν κατόπιν συνεννοήσεως και ε, ομοφωνίας μεταξύ επιτροπής, εμπλεκόμενων φορέων και ε, από τα κράτη. Εάν θέλουμε να καταστρέψουμε λοιπόν τη σχετική παραγωγή στην Ευρώπη, Βεβαίω θα ασχοληθήσουμε αυτό το δρόμο, αλλά πρέπει και να δώσουμε στις νεαρές μητέρες που δεν έχουν για λόγους είτε ε, παθολογικούς είτε οικονομικούς τη δυνατότητα ή άλλους να ε, θρέψουν τα παιδιά τους με το μητρικό θυλασμό ή αργότερα δεν έχουν καν το χρόνο ενδεχομένω να μαγειρέψουν για τα βρέφη τους και θέλουν το βαζάκι τύπου Γκέρμπερ. Ε, πρέπει να του εξηγήσουμε γιατί το πράττουμε αυτό. Α είμαστε όσο το δυνατόν πιο αυστηροί σε σχέση με την ε, παραγωγή των τροφίμων και το σχετικό κλάδο, αλλά μέχρι τότε δεν δέχομαι εγώ αυτέ τι αντιρρήσει. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Μόζερ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ήταν ενδελεχέστατη η παρουσίαση των αντιρρήσεών σας, κύριε συνάδελφε. Κύριε Χάσπρου ήταν σκιώδη συγκίτρια το 2006. Θέλαμε λοιπόν να υποστηρίξουμε δύο από τις ε, ενστάσεις. Η πρώτη αφορά το γάρα στη σκόνη. και τα μείγματα. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί ως προς την ε, διαφήμιση και τους ισχυρισμούς τους σχετικούς με την υγεία σε αυτό επιμένουμε και πρέπει να δίνονται οι επιλογές στον καταναλωτή, να, να έχει την ενημέρωση που θα το επιτρέπει να επιλέγει. Μην ξεχνάμε ότι το βρέφος είναι μια, πολύ, μια ιδιαίτερα ευάλωτη ομάδα. Απαιτείται η μέγιστη λοιπόν ε, προσοχή στο τι θα καταγράφεται στις διαφημίσεις. Δεν πρέπει να γίνεται υπερβολική. Ε, δεν πρέπει να επενούνται υπερβολικά τα προϊόντα αυτά Και επίσης σε σχέση με τα τρόφιμα που έχουν ειδικού ιατρικούς στόχους μπορούμε επίσης να συμφωνήσουμε. Για τα κατεργασμένα όμως τρόφιμα πιστεύουμε ότι θα ήταν λάθος η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταλήξει, να επιτρέψει την διάθεση στην αγορά τροφίμων που περιέχουν πάνω από 30% ζάχαρη, μέχρι και 30% ζάχαρη, όταν μια από τις κύριες προκλήσεις των κοινωνιών μας είναι η παχυσαρκία και μάλιστα η παιδική παχυσαρκία. Άρα πρέπει κάτι να κάνουμε. Μέχρι τώρα η ΕΦΣΑ δεν είχε τη δυνατότητα να εξετάσει τη σύνθεση των, των επεξεργασμένων τροφίμων. Δεν πρέπει να επιτρέπεται λοιπόν να κυκλοφορούν τρόφιμα, ε, μάλιστα βρεφικές τροφές με τέτοια υψηλή περιεκτικότητα. Εγώ προτείνω στους σοσιαλιστές και δημοκράτες να υποστηρίξουν την πρόταση. Άρα περιμένουμε να δούμε τα Ευχαριστώ κύριε Σελίμωβιτς, ευχαριστώ πολύ. Ε, θα μιλήσω εκ μέρους του Φρέντερικ Ρέις και όδους, γιατί που δεν μπόρεσε να βρεθεί εδώ σε αυτή την τελευταία συνάντηση του έτους και συμφωνώ με τα όσα μου μετέφεραν σας πω. Υπήρξε εισηγητή πριν από 2,5 χρόνια για το βασικό κανονισμό για τον οποίο συντάχθηκαν αυτέ οι τρει ενστάσεις και υπάρχουν κάποιε επιφυλάξει με αυτό το κείμενο. Πρώτα απ' όλα μερικά γενικά σχόλια θεωρεί ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για ένσταση αλλά για την ανάγκη απόλυτης αναδιατύπωσης ε, ε, του κειμένου αυτού που ε, ενέκρινα το 2013 η πράσινη και η λυπή και που το 2016 θα τεθεί σε εφαρμογή. Καταλαβαίνουμε γιατί οι ενστάσεις του κυρίου Τέιλορ ε, αναφέρονται σε αυτή την νομοθεσία που υιοθετήθηκε το 2013 και εκ μέρους του κ. ήθελα να τονίσω αυτή την αντίφαση με ένα απόσπασμα της ομιλίας του στην Ολομέλεια του Καρ Σλέιτερ και η των Πρασίνων αλλά και του Μισελ Ριβασί. Παραθέτω, καλωσορίζουμε την εισαγωγή της αρχής της προφύλαξης στο κείμενο αλλά επίσης θέλουμε συγκεκριμένους κανόνες για τη χρήση των ανοηλικών και αυστηρότερους κανόνες επισήμανσης και διαφήμισης. Είναι σημαντικό να μην γίνεται παραπλάνηση των καταναλωτών και συνεπώς θα ψηφίσουμε υπέρ του κειμένου αυτού. Τέλος της παράθεσης. Ε, ίσως για πολιτικούς λόγους να έχουν αλλάξει άποψη οι πράσινοι με πραγματικό κίνητρο, την αποκλειστικό θυλασμό μετά τους ε, έξι μήνες όπως προτείνεται από τον Παγκοσμίο Οργανισμό Υγείας και εμείς καταλαβαίνουμε ως φιλελεύθεροι ε, αντιτιθέμεθα στην, ε, στον περιορισμό της ελεύθερης επιλογής των γυναικών να, να ή όχι για διάφορους λόγους γιατί μερικές φορές δεν μπορούν να ε, το κάνουν παράλληλα με την επαγγελματική του ζωή ή γιατί ορισμένε φορές δεν μπορούν. Ε, τώρα για να δούμε κάποιες λεπτομέρειες για την πρώτη ένσταση για τα βρεφικά τρόφιμα και τα τρόφιμα παρασκευάζοντα δεύτερης βρεφικής ηλικίας για να περάσουμε στο πρώτο επιχείρημα οι πράσινοι προσπάθησαν να μας κάνουν να πιστέψουμε ότι υπάρχει νομικό πρόβλημα, νομική ε, αντίφαση μεταξύ της σύσταση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αυτό είναι λάθος, Όχι μόνο γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διασφαλίζει τη συνοχή του κειμένου, αλλά και για τα κράτη-μέλη Εφαρμόζονται τις κατευθυντές γραμμές του ΠΟΕ και δεν τίποτα νέο δεν έχει συμβεί από τη δημοσίευση του νέου κανονισμού στην επίσημη εφημερίδα. Το δεύτερο επιχείρημα είναι του συνήθε. Θέλουν να επεκτείνουν την απαγόρευση των διαφημίσεων για τα παρασκευάσματα δεύτερη βρεφική ηλικία. Συγκεκριμένα ε, γάλα για βρέφη από 6 μέχρι 8 επειδή αυτό το επιχείρημα ήδη απορρίφθηκε με 100 ψήφους και το 2012 γιατί θα δημιουργήσει αθέμητο ανταγωνισμό για τα παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας όπου τα βρέφη χρειάζονται μεικτή ε, διατροφή. Και επίσης κάτι άλλο για ένα οριζόντιο ζήτημα ε, επιμολυντών. Φυσικά έχουμε τις ίδιες απόψεις όσον αφορά το περιορισμό των φυτοφαρμάκων στα ε, βρεφικά τρόφιμα, αλλά να σας πω ότι έχουμε τους πιο αυστηρούς κανόνες στην Ευρώπη με ελάχιστο όριο καταλήπων. 0,01 μιλιγράμμα ανά κιλό βάσει της αρχής προφύλαξης. να το να ζητάμε μηδενική ανοχή φυτοφαρμάκων ως γενική αρχή είναι εντελώ μη ρεαλιστικό. Όλοι γνωρίζουμε ότι ορισμένε φορέ ε, το περιβάλλον ε, είναι μολυσμένο με διάφορα φυτοφάρμακα ε, και κατάλοιπά Μπορεί λοιπόν να υπάρξουν κατάλοιπα σε ορισμένα προϊόντα, δυστυχώ. Επίση, αληθεύει, όπω είπε η Κομισιόν, υλοποιώντα τον κανονισμό, ότι θα προσέχει τα CMA και γι' αυτό αναμένουμε ακόμα δράση για αυτό το θέμα και η Γι' αυτό το λόγο η Κομισιόν έχει πιέσει την ΕΦΣΑ για να ενημερώσει, να επικαιροποιήσει τον κατάλογο των φυτοφαρμάκων με αυστηρότερα ε, όρια από το 0,01 μιλιγκράμμα ένα κιλό. Τέλος, όσον αφορά την τελευταία ένσταση μέσω του σκιώδους μας, σε αυτή την περίπτωση δεν αναφερόμαστε σε κανονικούς ε, καταναλωτές, αλλά σε ασθενείς, μερικές φορές πολύ με χρόνιες ασθένειες που οδηγούν και σε αναπηρία. Έγινε διευκρίνηση μεταξύ του κανόνα, ε, μεταξύ της ενημέρωσης στον κανονισμό και της διαφήμισης που πρέπει να περιορίζεται. Τώρα έχουμε μια σαφή πρόταση ότι η ενημέρωση των επαγγελματών της υγείας δεν πρέπει να είναι διαφημιστική αλλά ενημερωτική. Για άλλη μια φορά ο κύριος Τέιλορ δείχνει ότι θέλει πλήρη ε, αναδιατύπωση της νομοθεσίας που δεν μπορεί να είναι στόχος της ένστασης σε μια κατεξοδότηση πράξη. Γι' αυτό το λόγο προτείνουμε να απορρίψουμε και τις τρεις ενστάσεις του κ. Τέιλορ. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Γκοντίν. Ναι, ευχαριστώ. Λοιπόν, οι τρεις ενστάσεις του κυρίου Τέιλορ για τα παρασκευάσματα για βρέφη ασθενείς ε, και ε, μικρά παιδιά δημιουργούν ανησυχίες όσον αφορά τα κατάλληλα αυτοφαρμάκων όσον αφορά και την επισήμανση επίσης το μητρικό γάλα είναι η καλύτερη λύση βέβαια, οπότε οι συστάσεις του ΠΟΕ για τους πρώτους 6 μήνες, ε, για τον απόλυτο θυλασμό, τόσο όσον αφορά την επισήμανση των ε, παρασκευασμάτων, Για αυτή την επισήμανση λοιπόν υποστηρίζουμε τον κύριο Τέιλερ. Όσον αφορά το θυλασμό, μια γυναίκα που θέλει να θυλάσει δεν θα επηρεαστεί από την ύπαρξη δειγμάτων. Αντιθέτως όμως μπορεί να επηρεαστεί μετά δημιουργώντας έτσι μια ειδικευμένη αγορά. Τώρα για τη μηδενική παρουσία φάρμακών στα προϊόντα αυτά, η σύσταση της Κομισιόν είναι όντω συζητήσιμη ακόμη και στη διατύπωση και συμφωνούμε με τον κύριο Τέιλορ στο ότι λείπει όσον αφορά την απουσία του γλυφοσάτ στα περιορισμένα φυτοφάρμακα παρότι είναι αυτό που χρησιμοποιείται όπως γνωρίζουμε όλοι περισσότερο στον κόσμο. Τέλος, τα ε, γενετικό τροποποιημένα προϊόντα θα πρέπει να προσθεθούν. Όσον αφορά το DHI που είναι λιπαρό οξύ για την ανάπτυξη ε, των παιδιών, βάσει των μελετών υπάρχει κατάχρηση εδώ. Το DHI αντικατάστασης δεν ε, είναι συγκρίσιμο με το μετρικό. Επίσης είμαστε υπέρ της δημοσίευσης του καταλόγου των ενδιαφορεμένων με τους οποίους έγινε συζήτηση για να δημιουργηθούν αυτές οι ενστάσεις. Ε, συμφωνούμε με τον κίνδυνο παχυσαρκίας ε, λόγω της υπερβολικής δόσης ζάχαρης ε, που είναι τριπλάσια δόση από αυτή του ΠΟΕ. Τέλος για τα παρασκευάσματα για δικούς ιατρικούς σκοπούς. Συμφωνούμε με τον εισηγητή. Τα προϊόντα αυτά δεν πρέπει να αποτελούν το αντικείμενο καμίας διαφήμισης και δεν πρέπει να περιλαμβάνουν διατροφικούς ισχυρισμού. Τέλος, συμφωνούμε με πολλά αυτά τα ζητήματα που θέτει ο κ. Τέλορ, αλλά δεν έχουμε ακόμα οριστικοποιήσει τη θέση μα για αυτά τα τρία κείμενα και για να διαπιστώσουμε κατά πόσο πρόκειται για ε, κείμενα που βοηθούν να, προχωρήσουμε λίγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Γκαρδίνη. Ευχαριστώ εντάχει. Λοιπόν, Κοιτάξτε τώρα, ακούγοντα το συνάδελφο, ο οποίο περιέγραψε τι τρεις ενστάσεις και τι υποστήριξε με σημαντικά επιχειρήματα, Τώρα βέβαια δεν θυμάμαι ήταν παρόν σε όλες τις εργασίες ε, στην προηγούμενη θητεία για να καταλήξει σε, για να, που είχαν ως αποτέλεσμα τα έγγραφα τα οποία ψηφίστηκαν. Ε, αυτές οι ανησυχίε μας είχαν απασχολήσει στην αρχή για να κάνουμε όλες αυτές τις εργασίες, οι οποίες διέρχεσαν δύο έτη και έγιναν σε βάθος. Οπότε τώρα είναι σαν να ε, Και τώρα είμαστε σαν να κάνουμε τα πρώτα σαν την Πινελόπη, η οποία έφτιαχνε το ύφασμα και το, και το υφάδι και μετά το χάλαγε. Ε, ενώ δεν έχουμε ξαναγυρίσει στο σημείο όλα αυτά έχουν ελεγχθεί, τα έχουμε εμβαθύνει, τα έχουμε λάβει υπόψη και πιστεύω ότι τελικά το αποτέλεσμα που έχει επιτευχθεί είναι το βέλτιστο διότι βασίστηκε στο ότι θελήσαμε να καθισχάσουμε όλες αυτές τις ανησυχίες και να δώσουμε μια απάντηση σε αυτές. Επειδή είπε συνάδελφος προηγουμένως ότι τα κράτη-μέλη ενδεχομένως μπορούν να επιβάλλουν περαιτέρω περιορισμού στη διαφήμιση. Είναι πράγματι, ξέρετε αυτό, είναι ήδη ένα ενδεχόμενο που συζητείτε τα κράτη-μέλη να μπορούν ε, να εφαρμόσουν περαιτέρω περιορισμούς όσον αφορά τη διαφήμιση ε, η οποία διαφήμιση θα γίνεται μόνο σε ειδικευμένα περιοδικά. Για το ω3, ξέρετε, είναι ένα υλικό πολύ γνωστό που ο κόσμος το βλέπει πολύ θετικά. παλιότερα το χρησιμοποιούσε ο κόσμος προαιρετικά και παρατηρήθηκε ότι αυτό δημιουργούσε ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα για αυτούς που δεν το χρησιμοποιούσαν. Γι' αυτό το λόγο επινοήθηκε αυτή η εισαγωγή για να έρθουν ορισμένα πλεονεκτήματα που ήταν πλεονεκτήματα στην αγορά ουσιαστικά. πιστεύω ότι αν περάσουν αυτέ τι τρει ενστάσει θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Γιατί επαναλαμβάνω, ε, τι ίδιε ανησυχίε είχαμε και εμεί. Ε, τι εξετάσαμε, τι εμβαθύναμε, εργαστήκαμε με σοβαρότητα. Και τώρα, άμα να πάμε να τα ξαναρχίσουμε όλα την αρχή. Να ξαναρχίσουμε από την αρχή μια τόσο σκληρή προσπάθεια που έγινε πριν δύο χρόνια, που διήρκησε δύο χρόνια, θα ακολουθήσει μια περίοδο νομική αβεβαιότητα και θα δημιουργήσουμε σοβαρά προβλήματα. Όχι μόνο στον τομέα Μην ξεχνάμε ότι αυτοί οι τομεί ε, που είναι και τόσο υψηλό επίπεδο, ε, αν υποστούν ε, βλάβη, θα έχουν μεγάλε απώλειε, χάνονται θέσει εργασία, αλλά θα υπάρξουν και προβλήματα και για του καταναλωτέ. Καταναλωτέ οι οποίοι δεν θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν αυτά τα νέα μέσα προστασία που προσφέρει αυτό ο νέο κανονισμό σε σχέση με το τι υπάρχει σήμερα Τώρα λοιπόν, ε, ξέρετε, ε, όλες αυτές οι ανησυχίες που αναφέρονται εδώ στις ενστάσεις, εμείς τις είχαμε εξετάσει. Τις είχαμε εξετάσει. Δεν το θυμάστε. Πολύ προσεκτικά ελήφθησαν υπόψη και με μεγάλη επιμέλεια τις εμβαθύναμε. Οπότε θα ήθελα να παρακαλέσω άπαντες να μην ε, διαπράξουν ένα τέτοιο σφάλμα. Ευχαριστούμε κυρία Τζεντήλια. Ναι, ευχαριστώ πρόεδρε παρεμβαίνω επειδή και εγώ είμαι παιδίατρος ε, ε, βέβαια ε, όχι προσωρινά φυσικά δεν ασκώται επάγγελμα αλλά εδώ βλέπω ότι εξολογούμε ένα ζήτημα Ε, των σοσιαλιστών και δημοκρατών εδώ διάβασα τις ενστάσεις επαναξιολόγησα τις ίδιες ενστάσεις και βάση του κειμένου και των εργασιών ε, που έγιναν ε, σε σχέση με τα έγγραφα ειλικρινά αυτή η θέση μου φαίνεται ε, λίγο ακραία. Βέβαια είναι σημαντικά τα ζητήματα και πρέπει φυσικά να έχουν την προσοχή μας. Ε, αυτό αναμφίβολα. Σίγουρα κάθε γυναίκα πρέπει να προτιμά όταν επιλέγει να βιώσει αυτή την ομορφότερη εμπειρία στον κόσμο, δηλαδή το να φέρει ένα παιδί στον κόσμο, θα πρέπει να ζει το θυλασμό. Αλλά ορισμένε παθολογίε δεν επιτρέπουν κάτι τέτοιο. Και μερικές φορές, ξέρετε, είναι και το ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο ζει μια γυναίκα που μπορεί να μην επιτρέπει κάτι τέτοιο. Ξέρετε, η οργάνωση της εργασίας, το πόσο εύθραυστα είναι τα συστήματά μας ε, κοινωνικής πρόνοιας ε, ε, λόγω των επιχειρήσεων κανόνες που φαίνεται να είναι ισορροπημένοι αλλά που ως, στην καθημερινή ζωή επηρεάζουν αρνητικά τις γιοές γυναικών οι οποίες πρέπει να γυρίσουν στην εργασία τους πολύ νωρίς μετά από τη γέννηση αυτό τώρα αφορά της αντισμητρότητας αλλά δεν θα εξετάσουμε αυτό τώρα σήμερα εδώ αλλά πρέπει να το ξαναζητήσουμε κάποια στιγμή. Αυτό πρέπει να μας το υποσχεθείτε. Ε, εγώ λοιπόν ε, θα έλεγα ότι πρέπει να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη για να έχουν κάποιες πολιτικές πιο φιλικές προς το θυλασμό. Εντάξει το λέω κάπως, ακούγεται κάπως δημαγωγία τώρα αυτό. Ε, ο θυλασμός ως ε, ε, στοιχείο αντιμετώπισης της φτώχειας ακούγεται λίγο δημαγωγικό αλλά ξέρετε υπάρχουν επιστημονικά τεκμήρια γι' αυτό αλλά τέλος πάντων αυτή τη στιγμή ας προσπαθήσουμε να εξαφανίσουμε περιβάλλοντα που υποχρεώνουν τις γυναίκες να κάνουν τη μία επιλογή σε σχέση με την άλλη ε, όταν υπάρχουν τέτοιου είδου δυσκολίε. Ε, για παράδειγμα, αναρωτιέμαι γιατί τα νοσοκομεία στη δική μου τη χώρα, ε, τα νοσοκομεία στην Ιταλία, λαμβάνουν δωρεάν από τις βιομηχανίε του τομέα το δείγμα του γάλακτος που εύκολα παραδίδεται στα χέρια στις μικρά τέτοια θέματα, μικρές σκέψεις που θα μπορούσαν να μα βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα του φυλασμού να ακολουθήσουμε μια άλλη οδό ε, σε σχέση με το ζήτημα αυτό. Αυτά κύριε Πρόεδρε, αυτή είναι η μικρή μου συμβολή. Αλλά θα ήθελα να το ξανασκεφτούμε πριν αποφασίσουμε τι απόφαση θα λάβουμε συνολικά εδώ ως ομάδα. Κύριε Εκ. Μίστερ Εκ. Danke, Herr Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρόεδρε, θα ήθελα να επανέλθω σε ένα στοιχείο από τις τρεις ενστάσεις του κύριου Τέιλορ. Για τα παρασκευάσματα για βρέφη και δεύτερης βρεφικής ηλικία που περιλαμβάνουν πολύ ζάχαρη. Έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη. Η αδερφή μου και ο γαμπρός μου είναι νευρολόγος, πρώτος και ψυχίατρος ο δεύτερος. Και αναρωτιούνται γιατί αρέσουν τόσο πολύ τα γλυκά στα παιδιά. Και μου είπαν ότι αν τα παιδιά τα ταΐζουμε με πολύ γλυκά τρόφιμα, όταν τους στερήσουμε τα γλυκά αυτά, τότε στους νευρώνες δημιουργούνται κάποιες συνάψεις στον εγκέφαλο του παιδιού που έχουν σαν αποτέλεσμα διαταραχές και συνεπώς η κατανάλωση ζάχαρης και η στέρηση της ζάχαρης δημιουργούν αλλαγές στις ε, συνάψεις των νευρώνων. Δημιουργούμε δηλαδή γενιές παιδιών που τελικά θα εξαρτώνται από τη ζάχαρη. Όλοι ξέρουμε τις αρνητικές συνέπειες από υπερβολική κατανάλωση ζάχαρης και όχι μόνο για τα παιδιά, για όλους. Με αυτόν τον τρόπο είναι εύκολο για τους παραγωγούς τροφίμων. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούν ολόκληρες γενιές ανθρώπων που θα θέλουν να καταναλώνουν ζάχαρη. Μεγάλη περιεκτικότητα λοιπόν σε ζάχαρη, ε, σε τρόφιμα που προορίζονται για μικρά παιδιά είναι εγκληματικό. Κυρία Μίλλερ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η ναι, κυρία Μέλιορ. Εγώ δεν θα τα πω τόσο δογματικά όπως τα είπε ο κύριος Εκ. Όμως παρόλα αυτά με Πλήσει μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε αυτά που λέει ο ΠΟΕ, που μιλάει για 10% και σε αυτά που έχουμε εμείς στα δικά μας κείμενα, που είναι 30% περιεκτικότητα. Μα πώς είναι δυνατόν να υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά. Πώς είναι δυνατόν να μην τηρούμε πιο πιστά τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Όταν ε, πρόκειται μάλιστα για την διατροφή των βρεφών. Η διαρρεκτικότητα λοιπόν σε ζάχαρη πράγματι μου φαίνεται ιδιαίτερα υψηλή. Έπειτα η αρχή της μηδενικής ανοχής σε φυτοφάρμακα. Έχουμε και άλλους κανονισμούς και απευθύνουμε εδώ στην Επιτροπή. Και για άλλα πράγματα, αυτή η ιστορία της ανοχής μηδέν είναι κάτι το ρεαλιστικό. Μήπως θα ήταν καλύτερα να βάλουμε ένα πολύ χαμηλό όριο που να είναι όμως πιο ρεαλιστικό. Ευχαριστώ πολύ, λέει η κυρία Σόμερ. Με κάθε ειλικρίνεια πρέπει να σας πω ότι δεν είμαι καθόλου πεπισμένη από τα επιχειρήματα των πρασίμων. Οι ενστάσεις αυτές είναι καθαρά ιδεολογικού τύπου και τίποτα άλλο. Κι εγώ είμαι υπέρ ε, του μητρικού γάλατος, του θυλασμού έξι μήνες, θύλασα και εγώ τα παιδιά μου, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι δεν φτάνει πάντα για όλες τις γυναίκες. Κάποια μέρα έτσι καλλιώς θα πρέπει να περάσουμε στο πιπερό. Εγώ δεν δούλευα εκείνη την εποχή, αλλά πολλές φίλες μου που δούλευαν δεν μπορούσαν να επιτρέψουν στον εαυτό του την ίδια πολυτέλεια που επέτρεψα και εγώ στο δικό μου και σταμάτησαν να θυλάζουν τα παιδιά του γιατί έπρεπε να γυρίσουν στη δουλειά. Και είναι πολύ δύσκολο να δουλεύει κανεί και να συνεχίζει να θυλάζει. Είναι αδύνατον στην πράξη. Γι' αυτό και υπάρχουν αυτά τα παρασκευάσματα εξάλλου. Η κατεξουσδότηση πράξη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή το λένε ότι ο μητρικός θυλασμός είναι ο καλύτερος τρόπος διατροφής του νεογέννητου και οι αξιολογήσεις που γίνονται για τα παρασκευάσματα αυτά είναι πάρα πολύ αυστηρές. Ο καταναλωτής έχει σαφείς πληροφορίες, γίνονται διακρίσεις ανάμεσα στα παρασκευάσματα πρώτης ηλικίας, δεύτερης ηλικίας και όταν υπάρχουν υπόνοιες για βλάβες στην υγεία, έτσι κι αλλιώς ο μητρικός θυλασμός παρουσιάζεται σαν τον καλύτερο τρόπο για να θρέψει κανείς τα παιδιά του. Τώρα, κατά πόσο επιτρέπονται οι διαφημίσεις για τα γάλατα δεύτερης βρεφικής ηλικία, ναι, αλλά πολύ περιορισμένα, μόνο σε δικευμένα περιοδικά. Άρα είναι υπερβολικό να λέμε να απαγορευτούν πλήρως οι διαφημίσεις Μα αγοράζουν τέτοια ειδικευμένα περιοδικά οι γονεί για να ξέρουν ποιο γάλα δεύτερη ηλικία να δώσουν στα παιδιά του. Όχι. Οι γιατροί, οι παιδίατροι τα παίρνουν τα περιοδικά αυτά για να ενημερώνονται. Όχι οι γονεί. Και αν τα προϊόντα αυτά ε, χρησιμοποιούνται από ιατρικό προσωπικό, τότε προφανώς η κατάσταση είναι σαφής και το ότι λέγεται δεν είναι καν αναγκαίο. Έχουμε λοιπόν κανόνες και δεν υπάρχει λόγος να παριστάνουμε ότι είμαστε σε έναν χώρο εκτός δικαίου που ο καθένας θα έκανε ό,τι θέλει. Όχι, και όπως είπε και κάποιος άλλος συνάδελφος, οι χώρες μέλη μπορούν να θετήσουν πιο αυστηρά μέτρα αν το θεωρούν αναγκαίο. Ωραία, τι άλλο θέλουμε λοιπόν. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχουν ενστάσεις αυτές. Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας έχει υποβάλει συστάσεις που στο κάτω-κάτω δεν είναι και αυτές οι ιερές. Υπάρχουν πολλές συστάσεις από τον ΠΟΕ που όμως, ε, από τον που όμως δεν είναι επιστημονικού τύπου για τις χώρες μέλη. Και εμείς έχουμε τη δικιά μας επιστημονική αρχή η οποία υποβάλλει συστάσεις. Όσον αφορά τώρα την περιεκτικότητα στη ζάχαρη, εδώ δεν βλέπω συστηνόμενη περιεκτικότητα όσον αφορά την κατανάλωση στη ζάχαρη. Όντω, μπορούμε να συνηθίσουμε τα παιδιά να τρώνε όλο και περισσότερη ζάχαρη. Και συνήθω οι παππούδε είναι αυτοί που το κάνουν, που δίνουν ε, σοκολάτες και γλυκά στα παιδιά. Το λέω από προσωπική εμπειρία αυτό, εν πάση περιπτώσει. Κλείνω την παρένθεση. Πιστεύω ότι υπάρχει και η Γερμανική Ένωση για τη Διατροφή όπου συμμετέχουν επιστήμονες και υπάρχει η υπηρεσία αυτή εδώ και δεκαετίες. Συμβουλεύει όλους τους πολιτικούς και θεωρεί ότι οι συστάσεις του ΠΟΗ δεν είναι κάτι ιερό. Έπειτα ξέρουμε ότι η ζάχαρη είναι αναγκαία. Γιατί δίνει ενέργεια. Το σώμα μας χρειάζεται ζάχαρη. Δεν πρέπει να θεωρούμε τις συστάσεις λοιπόν του ΠΟΗ σαν κάτι που πρέπει να ακολουθήσουμε στα τυφλά. Και υπάρχει και η διαφορά ανάμεσα στις διάφορες μορφές. Άλλο η φρουκτόζη και άλλο άλλες μορφές ζάχαρης. Όλα αυτά λοιπόν προκαλούν σύγχυση. Και έχουμε και επιπλέον κόστος. Εγώ πιστεύω ότι η κριτική των πρασίνων είναι υπερβολική. Δεν μας πείθει. Κάτι το οποίο με πείθει είναι το ότι οι σημερινοί κανόνες είναι σίγουρα οι πιο αυστηροί που είχαμε ποτέ στην ιστορία μας. Άρα το να κάνουμε τους κανόνες αυτούς ακόμα πιο αυστηρούς... Όπως... Θα ήταν περιττό. Δεν το χρειαζόμαστε. Είναι αρκετά καλοί οι κανόνες. Πέραν αυτού, όπως υπόθηκε, σημειώνεται πάντα ε, ότι είναι καλύτερη η λύση του μητρικού θυλασμού σε κάθε προϊόν. Τι άλλο θέλετε λοιπόν. Είναι άλλωστε γνωστό ότι σπάσιμο ότι ο μητρησικός θυλασμός είναι ε, ε, η καλύτερη λύση για το βρέφος. Η επισήμανση και από γιατρούς και νοσοκόμες νομίζω ούτως ή άλλως ε, δεν χρειάζεται γιατί είναι γνωστό ότι σπάσιμο. Επίσης υπάρχουν γυναίκες οι οποίες δεν είναι σε θέση να φυλάσσουν. Δεν τα καταφέρνουν για λόγους λογικού ή πρέπει να εργαστούν. Δεν μπορούμε λοιπόν αυτές να τις βάζουμε στο εδόλιο του κατηγορουμένου, να τις, το τους δημιουργούμε ενοχικά σύνδρομα γιατί δεν μπορούν να προσφέρουν το θυλασμό. Δεν χρειάζεται να έχουν τύψεις πάνω από όλα τα προβλήματά τους. Ευχαριστώ Μπάλτσο. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε. Έχω μια ερώτηση. Όταν νομοθετούμε να ρωτήσω το εξής. Τι εννοούμε όταν λέμε διαφήμιση για τις ε, παιδικές τροφές, ε, γάλα πρώτης και δεύτερης ηλικίας. Αφού έχουμε δεδομένα. Εάν αυτά παρουσιάζονται αντικειμενικά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης αντικειμενικά, ε, επιστημονικά δοκιμασμένες γνώσεις μπορούν να θεωρηθούν ε, ως διαφήμιση. Γιατί αν απαγορεύεται κάτι τέτοιο, προφανώς ισοδυναμεί και με απαγόρευση του ίδιου του προϊόντος. Γιατί δεν μπορεί να προσφερθεί η πληροφορία που χρειάζεται ο καταναλωτής. Άρα πρόκειται για απαγορεύση του ίδιου του προϊόντος. Εάν υπάρχουν ισχυρισμοί ότι είναι πολύ πιο υγιεινή ως τροφή ή ότι μπορεί να είναι καλύτερη από κάτι άλλο, από τον μητρικό θυλασμό ιδιαίτερος. Αν λοιπόν υπάρχει κάποια τέτοια δήλωση ή ισχυρισμός για το ε, γάλα πρώτης και δεύτερης ηλικίας ή για κάποιο παιδικό σκεύασμα, ε, προφανώς δεν μπορεί να ευσταθεί, αλλά εάν δεν επιτρέπεται κανένα τύπου διαφήμιση, τότε είναι σαν να απαγορεύουμε το προϊόν. Η κυρία Μαγκίνε, Πρόεδρε, θέλω και εγώ να συμφωνήσω με του συναδέλφου Γκαρδίνη και Ζόμερ. Όχι με λεπτομέρειε, αλλά θέλω να εξηγήσω τη δική μου την περίπτωση. Ήμασταν 8 στην οικογένεια μου, 8 παιδιά. Ε, τη μητέρα μου φαντάζομαι θα έπρεπε να την έχουν βάλει φυλακή, γιατί όταν ήμασταν 6 μηνών ε, μα έβαζε και ζάχαρη στον πιμπερόν. και για όνομα του Θεού ακούσατε, ακούσατε, τσάι και αγελαδινό γάλα. Ε, νομίζω ότι δεν έγινα πια και κανένα τέρας. Ακούγοντας λοιπόν τον συνάδελφο από του πράσινου, ανησυχώ λίγο για τις ε, επιταγές αυτές τι οποίες εκδίδουν ορισμένοι ως διατάγματα και επίση από άλλη προσωπική σκοπιά. Έχω τέσσερα παιδιά, έχω θυλάσει και τα τέσσερα και τα δύο ήταν δίδυμα μάλιστα. Είμαι περήφανη γι' αυτό, αλλά δεν ήταν καθόλου εύκολο. Όσοι λοιπόν λένε breast is best, ο μητρικός θυλασμός είναι ό,τι καλύτερο, προφανώς δεν το έχουν δοκιμάσει. Εδώ πέρα εμείς δεν κάνουμε επιλογές ε, στη θέση άλλων. Εμείς εξετάζουμε κατά εξουσιοδότηση συμπράξεις όπως έχουν συνταχθεί για να δούμε αν εξυπηρετούν το στόχο τους. Και εγώ πιστεύω ότι εξυπηρετούν το στόχο τους. Τα υπόλοιπα της συζήτησης μπορούμε να τα πούμε σε άλλη χρονική στιγμή. Συμφωνώ απόλυτα με τα σχόλια των συναδέλφων και απορρίπτω πολλά από αυτά που ακούστηκαν από τους συναδέλφου των Πρασίνων, προς οποίους τρέφω κάθε σεβασμό βεβαίως. Αλλά δεν θέλω μια νέα μητέρα ή ε, μέλουσα μητέρα να ε, έχει ακόμη περισσότερο άγχος. Γιατί νομίζω ότι αυτό έχουν καταφέρει οι συναδελφοί εδώ. Όταν κανείς είναι σε τόσο νεαρή ηλικία, όταν έχει μητέρα είναι σε τόσο νεαρή ηλικία ή γενικά είναι μικρομάνα, προφανώς έχει πάρα πολύ άγχος. Και κύριε Τέιλορ, με συγχωρείτε που θα επανέλθω, αλλά μια και κάνατε ένα σχόλιο για τη διαφήμιση. υπενισόμενους ότι θα μπορούσαν να κρίνουν μόνοι τους οι γονείς. Ε, κοιτάξτε, ας εμπιστευτούμε και τους ανθρώπους. Μπορούν και να διαβάζουν και να βρούνε άκρη. Η μητέρα μου μπορεί να μην είχε κάπου να ψάξει, γιατί δεν υπήρχε και σχετική νομοθεσία που θα της έλεγε ή οδηγίες που θα της έλεγαν ότι δεν πρέπει να βάζει ζάχαρη στο πιπέρο. Αλλά πρέπει να κάνουμε αυτό που θα ήταν το καλύτερο στην τωρινή μας εποχή για τους γονείς αλλά και για τα βρέφη και δεν πρέπει να απορρίψουμε τις πράξεις. Ο Πρόεδρος ευχαριστώ πολύ και πρέπει τώρα να ακούσουμε την Επιτροπή πιστεύω να και διατυπώθηκαν κάποιες ε, ερωτήσεις προς αυτή. Um, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε τον λόγο και ευχαριστούμε για αυτή την πολύ ζωηρή συζήτηση. Το πρώτο που θα ήθελα να καταστήσω απολύτως σαφές είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνεί με την άποψη ολόκληρη της επιστημονικής κοινότητα ότι ο σου απαρέχει την καλύτερη τροφή για υγιή βρέφη και εμεί έχουμε δεσμευτεί για την υποστήριξη του θυλασμού και ήθελα απλά να αναφέρω ορισμένε από τι πρωτοβουλίε σε αυτό το τομέα Υποστηρίζουμε τα κράτη-μέλη στο σχέδιο δράσης πολέμηση της παιδικης παιξαρκιας παξαρκίας 2014-2020. Χρηματοδοτούμε ένα πιλωτικό έργο που ονομάζεται Together για να προωθήσουμε υγιέστερους τρόπους ζωής και το θυλασμό μεταξύ των μητερών. Επίσης γίνονται προσπάθειες μαζί με αναπτυσσόμενες χώρες όπως περιγράφεται στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο πολιτικής που θα ενισχύσει τη μητρική και ευρευτική διατροφή. Δεδομένων αυτών μην ξεχνάμε ότι κάθε γυναίκα έχει το δικαίωμα να επιλέξει το θυλασμό ή όχι. Και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι η τελική επιλογή είναι προσωπική. Εκεί επισέρχεται η ευθύνη τη Ευρωπαϊκή Ένωση και η ευθύνη δική μα στου τομεί αρμοδιότητά μα είναι να διασφαλίσουμε πρώτον ότι αυτή η επιλογή δεν επηρεάζεται αρνητικά από εξωτερικού παράγοντε, δηλαδή από ε, παροχή εσφαλμένων ή παραπλανητικών πληροφοριών σε γονείς ή ε, νοσηλευτές που μπορεί να τους απομακρύνει από το θυλασμό και ότι επίσης όταν μια μητέρα αποφασίζει να μην θυλάσει να υπάρχει ένα εναλλακτικό προϊόν με τις ίδιες ε, θρεπτικές ικανότητες για τα βρέφη ώστε να βοηθήσει την ανάπτυξή τους. Και στο, στο πνεύμα αυτό εμείς διατυπώσαμε τους κατεξοδότηση κανονισμούς οι οποίοι βασίζονται στις πιο πρόσφατες επιστημονικές συμβουλές της ΕΦΣΑ όταν υπάρχει και έγιναν και εξωτερικές διαβουλεύσεις με κράτη-μέλη και με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Επιτρέψτε μου να σας πω δύο λόγια για την ΕΣΑ, διότι έχουμε παρατηρήσει ότι στην πρώτη ψηφίσματος ε, εκφράζονται ανησυχίες περί διαφάνειας και θέλω να σας διασφαλίσω, να σας διαβεβαιώσω ότι έγιναν διαβουλεύσεις με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και με τις ΜΚΟ και η Κομισιόν ε, εφάρμοσε τη μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια ε, για την κατάρτιση των κατεξοδότηση πράξεων και χάρη στη συμβολή των ΜΚΟ εξελίχθηκε το κείμενο αυτό και ε, σε θέματα προστασίας των καταναλωτών και σας διαβεβαιώ ότι και οι ΜΚΟ που βρίσκονται εδώ σήμερα μπορούν να το επιβεβαιώσουν. Οι κατεξοδότηση κανονισμοί περιλαμβάνουν σημαντικά βήματα προς τα εμπρός για την προστασία των καταναλωτών και υποστήριξη του φυλασμού. Να αναφέρω μερικά όλοι οι θρεπτικοί ε, ισχυρισμοί και ισχυρισμοί υγείας έχουν απαγορευτεί από το βρεφικό γάλο. Ενισχύσαμε τους κανόνες ε, για να γίνεται διάκριση μεταξύ βρεφικού παρασκευάσματων για βρέφη και παρασκευάσματα για βρέφη δεύτερης ηλικία. Και επίσης ε, έχουμε μεριμνήσει για τις επισημάνσεις για ειδικού σκοπούς για βρέφη. Πέραν αυτών, εμπνευσμένους από αυτούς που αφορούν το βρεφικό γάλα. Όπως είπε και η Γκροστέτ, βλέπουμε ότι αυτό το, η πρόταση ψηφίσματος ξανανοίγει κάποια ζητήματα πολιτικής που έχουν ήδη συμφωνηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή όταν έγινε η διαπραγμάτευση του βασικού κανονισμού. Θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι όταν υιοθετήκαν οι Κομισιόν κατά εξώτηση πράξης πρέπει να τηρήσει την εντολή του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου και δεν μπορεί να παρεκκλίνει από αποφάσεις πολιτική των βασικών πράξεων. Αυτό θα σήμαινε ότι υπερεύαινε τις εξουσίες της. Για παράδειγμα, το αίτημα να μεταχειριστούμε το, στις διαφημίσεις το παρασκεύασμα δεύτερης βρεφικής ηλικίας της διαφημίσεις ως παρασκεύασμα για βρέφη είχε, ήταν τροπολογία που απορρίφθηκε με σχεδόν 100 ε, ψήφους ε, κατά διαπραγμάτευση της βασικής πράξης. Τώρα, όσον αφορά τη διευθύνηση, αληθεύει ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων έχει αναφέρει ότι η σύνθεση των παρασκευασμάτων δεύτερης βασικής ηλικία πρέπει να είναι παρόμοια, αλλά όχι όμοια με αυτή των παρασκευασμάτων για βρέφει. Ωστόσο, η γνωμοδότηση της ΕΦΣΑ αναφέρεται στις απαιτήσει σύνθεσης. Μην ξεχνάμε όμως ότι αυτά τα δύο προϊόντα ε, παίζουν διαφορετικό ρόλο στην διατροφή των βρεφών. Οπότε η λογική μας είναι σαφής. Ε, τα παρασκευάσματα για βρέφη είναι όντως τα πρώτα μόνα ε, προϊόντα που, χρησιμο... αντικαθιστούν το μητρικό γάλα για βρέφη από μηδόν ετών. Αλλά όσον αφορά τα παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας και τις λοιπές τροφέ για βρέφη που καταναλώνονται μετά από τον τέταρτο ή τον έκτο μήνα, όταν ξεκινάει συμπληρωματική διατροφή ενδεχομένως πρέπει να φροντίσουμε για αυτά τα παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικία, ότι άλλα φυσιολογικά τρόφιμα που μπορεί να καταναλώσουν τα βρέφη θα πρέπει να έχουν ισχυρισμούς υγείας οπότε εκεί γίνεται μια διάκριση Οπότε μπορεί κανείς να φανταστεί το σενάριο όπου γονείς μπορεί να προτιμήσουν κανονικά τρόφιμα ακόμα και αν η συνολική του σύνθεση είναι κατάλληλη για βρέφη και μικρά παιδιά με υψηλά ποσοστά ζάχαρης ή με ε, μία σύνθεση που δεν συνίσταται όπως για παράδειγμα το αγελαδινό γάλα που δεν συνίσταται για τα βρέφη. Το ίδιο για του ισχυρισμού υγεία, όπω αναφέρθηκε η κατεξοδότηση κανονισμοί και εδώ ακολουθώ μια πιο διαρθρωμένη προσέγγιση. Όλοι οι ισχυρισμοί για τα παρασκευάσματα για βρέφη απαγορεύονται πλέον. Όσον αφορά τα παρασκευάσματα δεύτερη βρεφική ηλικία θα ληφθούν αποφάσει στο πλαίσιο του κανονισμού για του ισχυρισμού που καλύπτει συγκεκριμένα του ισχυρισμού που αφορούν την ανάπτυξη και την υγεία των βρεφών και των παιδιών. Και γνωρίζουμε όλοι ότι σύμφωνα με αυτόν τον κανονισμό μόνο οι ισχυρισμοί που βασίζονται σε αξιόπιστα ε, επιστημονικά στοιχεία επιτρέπονται ώστε να μην γίνεται παραπλάνηση των καταναλωτών. Και μην ξεχνάμε ότι έχει δικαίωμα εξέταση του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για όλα τα ζητήματα που ανακύπτουν για τα παρασκευάσματα αυτά στο πλαίσιο του κανονισμού περί ισχυρισμών. Οπότε θα υπάρξει ευκαιρία να συζητήσουμε περαιτέρω το ζήτημα αυτό στο μέλλον. Τώρα θα ήθελα να πω δύο λόγια για το DHA το οποίο αναφέρθηκε και την ε, η υποχρεωτική προσθήκη του DHA. Πιστεύω ότι εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι στην πρόταση ψηφίσματος η γνωμοδότηση της ΕΦΣΑ αναφέρεται μόνο μερικώς. Λείπει ένα κομμάτι της γνωμοδότησης της ΕΦΣΑ. Μάλιστα υπάρχει μια παράγραφος όπου αφού η ΕΦΣΑ εξηγεί όλες τις πιθανές ε, επιπτώσεις του DHA για τα παρασκευάσματα για βρέφη καταλήγει ότι φαίνεται φρόνιμο να παρέχεται προσχηματισμένο DHA σε ε, βρέφη δεύτερης ηλικίας όπως και στα βρέφη πρώτης ηλικίας παρότι τα ωφέλη αυτής της πρακτικής δεν μπορούν να ε, είναι βέβαια βάσει των δεδομένων που έχουμε τώρα και θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι η ΕΦΣΑ θα συμφωνήσει ε, με την παροχή κάποιων ε, ουσιών στα παιδιά μόνο εφόσον είναι ασφαλή. Αν λοιπόν η ΕΦΣΑ δεν είχε πιστεί ότι το DHA ε, ήταν εποφελές θα είχε συμφωνήσει με την προσθήκη αυτά. Κανένα επιστημονικό στοιχείο μάλιστα δεν αναφέρει, δεν υποστηρίζει το ενδεχόμενο κίνδυνο. Και τώρα δύο λόγια για τα φυτοφάρμακα. Εδώ θα ήθελα να τονίσω ότι ο κατεξοδότηση κανονισμός, κατεξοδότηση κανονισμοί έχουν ήδη ανοχή μηδενική. Είμαστε πολύ κοντά στη μηδενική ανοχή. Με το όριο το 0,01 μιλιγκράμμα ένα κιλό. Αυτό είναι ουσιαστικά το όριο ε, ποσοτικού προσδιορισμού. Βασίζεται στην αρχή της προφύλαξης. Επιπλέον, Έχουμε ήδη ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας των Τροφίμων να επικαιροποιήσει μια πιο ολοκληρωμένη αξιολόγηση του ζητήματος για επικαιροποίηση των κανόνων περί φυτοφαρμάκων βάσει επιστημονικών συμβουλών πλέον πρόσφατων. Ήδη δηλαδή το είχαμε κάνει αυτό τον Οκτώβριο 2014, αλλά δυστυχώς η ΕΦΣΑ τότε δεν είχε προλάβει να τηρήσει την προθεσμία ώστε να υιοθετηθεί η της πράξη. Επίσης, ε, τις ίδιες αυστηρές ε, διατάξεις ε, τις επεκτείναμε όσον αφορά τα φυτοφάρμακα για τα τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς. Τέλος, δύο λόγια για το επίπεδο ζάχαρης στα παρασκευάσματα για βρέφη. Πρέπει να πούμε ότι εδώ πράγματι αντιγράψαμε τους κανόνες που ίσχυαν αυτή τη στιγμή. Γνωρίζουμε ότι πρέπει να αναθεωρηθούν οι απαιτήσει σύνθεσης αυτών των προϊόντων. Ωστόσο, ήταν αδύνατο να ζητήσουμε από την ΕΦΣΑ να μας δώσει επιστημονική γνωμοδότηση επί του θέματος σε χρονικό πλαίσιο συμβατό με την προθεσμία της Κομισιόν για να εφηθήσει την κατεψιοδότηση πράξη του Ιούλιο του 2015. Όπως γνωρίζετε, η πόλη της ΕΦΣΑ είναι περιορισμένη και η ΕΦΣΑ εργάστηκε σκληρά τα τελευταία τρία χρόνια για πολλέ γνωμοδοτήσει που σχετίζονται με την υλοποίηση αυτού του κανονισμού, για παράδειγμα για τα προϊόντα ευρατίσματο, τα γαλάτα ανάπτυξη, τα αθλητικά τρόφιμα κτλ. Η Κομισιόν ήδη έχει δεσμευτεί δημόσια προ τα κράτη-μέλη και προ όλου του ενδιαφερομένου και αυτό μπορείτε να το δείτε στα πρακτικά των συναντήσεων. Να απαντά επίση και στα κοινοβουλευτικά ερωτήματα και μόλι ολοκληρωθεί η μεταφορά των κανόνων θα στείλουμε ένα αίτημα επιστημονική παροχή συμβουλών από την ΕΦΣΑ και θα προετοιμάσουμε αναθεώρηση των κανόνων. Τέλος, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι αν οι κατευθυντές κανονισμοί δεν υιοθετηθούν, αυτό θα σημαίνει ότι οι σημερινοί οι παλιοί κανόνες θα συνεχίσουν να ισχύουν. Κατά την άποψή μας, ε, μία ένσταση δεν πρόκειται να βελτιώσει την κατάσταση σε σχέση με το όσα έχουμε σήμερα και δεν θα κάνει τίποτα άλλο παρά να καθυστερήσει τη διαδικασία αναθεώρησης και της επιστημονικής επικαιροποίησης που τώρα βρίσκεται ήδη ε, πραγματοποιείται ήδη για τα φυτοφάρμακα και σύντομα θα γίνει και για τα επίπεδα ζάχαρης γιατί σε περίπτωση ένσταση, θα χρειαστεί να περιμένουμε την ψηφοφορία στην Ολομέλεια μετά στην Κομισιόν θα χρειαστεί να συζητήσουμε εσωτερικά για το τι συνέχεια θα δώσουμε σε αυτή την ένσταση. Αν κάποια από τα αιτήματα που αποτελούν κομμάτι αυτού του ψηφίσματος ακολουθηθούν και αλλάζουν ουσιαστικά τη σημερινή κατάσταση, σε αυτή την περίπτωση θα χρειαστεί επίσης να διενεργήσουμε και μια εκτίμηση αντικτύπου, το οποίο σημαίνει ότι η επικαιροποίηση των νέων κανόνων θα καθυστερήσει ακόμη περισσότερο και η Κομισιόν σίγουρα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να δεσμευτεί για κάποια προθεσμία για την υποβολή της νέας τη πράξη. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα επίση να πω ότι παραμένουμε στη διάθεσή σα για οποιασδήποτε ερωτήσει σε πιο τεχνικό επίπεδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Δεν πρέπει να το ξεχάσω. Δεν ξέρω κύριε Τέιλορ αν θέλετε να απαντήσετε, διότι ξέρετε έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ. Πολύ γρήγορα λοιπόν, ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Ενδιαφέροντα πάντως όλα όσα ακούσαμε. Ποτέ, ποτέ κανένας δεν με κατηγόρησε ότι είμαι μέλος της αστυνομίας θυλασμού. Κύριε Κροστέρ, θα μου ακούσατε στην αρχή που είπα ότι με τίποτα δεν είμαι κατά του βιβερό και ότι θέλω οι γονείς να αποφασίζουν πώς θα τέσουν το παιδί τους. Να είναι επιλογή για αυτούς. Ναι, είμαι πολιτικός και έγινα πολιτικός γιατί θέλω να καλυτερέψω τα πράγματα για τον κόσμο και για την εκλογική μου περιφέρεια. Αγωνίζομαι να μπορούν οι γονείς να έχουν ό,τι καλύτερο μπορούν για τα παιδιά τους. Το καλύτερο είναι ο θυλασμός, δεν το αμφισβητεί αυτό κανείς. Ο Πόι λέει 13% των ε, παιδιών στις 21 χώρες που μελέτησαν τρέφονται αποκλειστικά με θυλασμό. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι τα παρασκευάσματα για βρέφη, όταν αυτά χρησιμοποιούνται, να είναι όσο γίνεται καλύτερα. Και το να επιτρέπουμε τις διαφημίσεις για τα προϊόντα αυτά πρώτης και δεύτερης βρεφικής ηλικίας, είναι σαν να βάζουμε στο εμπόριο τα ίδια τα βρέφη. Πολλές φορές οι διαφημίσεις παρεξηγούνται και όπως είπαμε κινδυνεύουν τα παιδιά να υποφέρουν από παχυσαρκή αργότερα αν βασιζόμαστε στα λόμπη και στους ισχυρισμούς ε, των ε, κατασκευαστών αυτών των ε, προϊόντων. Εδώ πέρα πρόκειται μια ιδιαίτερα κερδοσκοπική αγορά. Να φροντίσουμε λοιπόν να δράσουμε προς το συμφέρον της υγείας των παιδιών και να απορρίψουμε την πρόταση αυτή κανονισμού. Πρόεδρος, Ευχαριστούμε. Η ψηφοφορία θα γίνει στις 14 Ιανουαρίου στην Επιτροπή μας και αν εγκριθεί τον Ιανουάριο θα ψηφίσουμε στην Ολομέλεια. Περνάμε τώρα στο τελευταίο θέμα που έχουμε για σήμερα στην ημερήσια διάταξη που είναι ανταλλαγή απόψεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με το έγκλημα κατά της άγριας πανίδας. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ευθύ αμέσω για την παρουσίασή της. Μη μακρηγορήσετε παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι. Το λαθρεμπόριο με προϊόντα της άγριας φύσης ε, και τα σχετικά εγκλήματα δεν είναι καινούργια φαινόμενα, ωστόσο η φύση του, η κλίμακα και οι συνέπειες τους έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Και δεν ε, μιλάμε μόνο για κάποια συμβολικής ε, σημασίας και ανάδειξης ήδη, ήδη δηλαδή που κινδυνεύουν με εξαφάνιση, αλλά και με εμπόδια στην ε, αϊφόρο οικονομική ανάπτυξη και βέβαια δίκτυα οργανωμένου εγκλήματος που σχετίζονται με τι δραστηριότητε αυτέ. Γι' αυτό ιδιαίτερω καλωσορίζουμε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που δείχνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο να καταδείξει αυτό το λαθρεμπόριο. Ιδιαίτερα υποστηρίζουμε το ψήφισμα του Ιανουαρίου 2014 και την σχετική επιστολή 81 και άνω βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς τον Επίτροπο Δέλα άμα τη του, άμα τη αναλήψη των καθηκόντων του. Είναι πολύ καλό λοιπόν στο ύψιστο πολιτικό επίπεδο να λαμβάνει τη δεύτερη σημασία το θέμα αυτό. Άλλωστε η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών τον, τον Ιούλιο του 2015 εξέδωσε αντίστοιχο ψήφισμα και βλέπουμε και δηλώσεις των ηγετών του G7 για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου προϊόντων της άρεας φύσης. Ιδιαίτερα λοιπόν θέλω με χαρά σήμερα να καταγράψω την επιτυχία της προόδου από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που μας επιτρέπει να υιοθετήσουμε ένα πρόγραμμα δράσης για την άγρια φύση πριν από την Παγκόσμια Μέρα Προστασίας της Φύσης που είναι η 3η Μαρτίου για το 2016 βεβαίως. έχουμε να κάνουμε μια πολυσχηδή προσέγγιση και μάχη για να, για να κερδίσουμε τον αγώνα αυτό. Συνεργαζόμαστε λοιπόν και με άλλες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, της Δικαιοσύνης και Εσωτερικών, ε, ΕΦΚΟ, Φορολογικών και αντίστοιχες γενικές διαθύνσεις. Επικεντρωνόμαστε σε τρεις ε, κύριες προτεραιότητες, την πρόληψη καταρχάς του λαθρεμπορίου και εδώ κοιτάμε τις ρίζες του κακού. Δεύτερον, την επιβολή της νομοθεσίας και την καταπολέμηση κάθε μορφής οργανωμένου εγκλήματος με πιο αποτελεσματικές κυρώσεις. Και επίσης ενισχύουμε τη συνεργασία μας με τους εταίρους μας το επίπεδο και με τις χώρες προελεύσεως και με τις χώρες όπου γίνεται η κατανάλωση ή η διαμετακόμιση των προϊόντων αυτών. Πολύ ευχαριστώ συνεργαστούμε μαζί σα. Ελπίζουμε να έχουμε και συμπεράσματα του Συμβουλίου και ελπίζουμε και θετική αντίδραση από πλευρά του Κοινοβουλίου. Κατά την προετοιμασία του προγράμματο δράσεω, παρακολουθούμε ταυτόχρονα και άλλε. Ε, δύο άλλες οδούς, με δύο παραδείγματα για να περιορίσω το χρόνο ομιλίας. Θα έχουμε μια μόνιμη επιτροπή που συνεδριάζει τον Ιανουάριο για να εξετάξει τα αντίστοιχα εθνικά προγράμματα δράσεως που πρέπει κάθε χώρα να καταθέσει εφόσον έχει θεωρηθεί ως χώρα που μπορεί να γεννά κάποιε ανησυχίε σχέση με το λαθρεμπόριο των ειδών αγρίας φύσης και βεβαίως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρακολουθήσει με αυστηρότητα την ε, απόλυτη υλοποίηση και βέβαια εάν υπάρχει πρόβλημα σε σχέση με αυτό με μια συγκεκριμένη χώρα κινδυνεύει και με αναστολή της συμμετοχής δεύτερον με συναδέλφους από τις ΗΠΑ προσπαθούμε να ενισχύσουμε περαιτέρω τη συνεργασία μας ιδιαίτερα ως προς τον προορισμό χωρών προτεραιότητας ώστε να αναλάβουμε με αυτές και τη διπλωματική δράση. Ξεκίνησε με ένα διάβημα στο Λάος Φερρυπίν πέρυσι. Κάτι που θα μπορούσαμε να επαναλάβουμε και πιο συχνά για να ακούγονται πιο ξεκάθαρα τα μηνύματά μας. Για να είμαι λοιπόν και ολοκληρώνοντας, το πρόγραμμα δράσης για την αγριαφύση έχει μπει σε τροχιά. Θα σας το παρουσιάσουμε στο πρώτο ε, τρίμηνο του 2016 και σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση, κύριε Γκέμπερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Κομισιόν ε, που ήρθε εδώ να μας παρουσιάσει την τρέξο κατάσταση. Όταν άρχισα να ασχολούμαι με αυτό το ζήτημα πριν από μερικά χρόνια εδώ στο Κοινοβούλιο, ήταν κάτι νέο. Τουλάχιστον έχουμε κάνει κάποια πρόοδο, τουλάχιστον στα χαρτιά πρέπει να πω. Έχουμε το ψήφισμα του Κοινοβουλίου, έχουμε μια ανακοίνωση, έγινε μια διαδικασία διαβούλευσης, μια τεράστια διάσκεψη πριν περίπου δύο χρόνια εδώ στις Βρυξέλλες. Έγιναν πολλά. Και τώρα έχουμε τον οδικό χάρτη που περιγράφει τρεις επιλογές δύο από αυτές χωρίς ε, νομοθεσία και η τρίτη με μια νέα νομοθετική πρόταση. Οι φήμες λένε ότι η Κομισιόν δεν θα διαλέξει την τρίτη επιλογή, δηλαδή την πιο νομοθετική επιλογή. Η ερώτησή μου λοιπόν αφορά ακριβώς αυτό. Μέχρι στιγμής οι περισσότερες ευρωπαϊκές πολιτικές έχουν βασιστεί σε μια σύσταση του 2007 και συχνά ε, όχι μόνο στον περιβαλλοντικό αλλά και σε άλλους τομείς παρατηρούμε ότι οι συστάσεις ε, δεν φέρνουν πραγματικά αποτελέσματα στην Ευρώπη. Τα κράτη-μέλη απλά τις αγνοούν. Οπότε πρέπει να κάνουμε πολλά περισσότερα. Και για να είμαι ειλικρινής, κοιτώντας τις ε, επιλογές 1 και 2 του δικού χάρτη, δεν κάνουν παρά λίγα παραπάνω από τη συστάση που έχουμε ήδη εδώ και μερικά χρόνια. Και παρατηρώντας κανείς το όλο ένα αυξανόμενο πρόβλημα του παρανόμου εμπορίου ειδών ε, της άγριας και χλωρίδας, ε, η κατάσταση είναι ενισχυτική. Μήπως θα έπρεπε να ε, σοβαρευτούμε λίγο, να, το, να τη δούμε λίγο πιο νομικά αυτή την εγκληματικότητα ως ένα σοβαρό έγκλημα όπως την εμπορία ανθρώπων, όπως τα ναρκωτικά. Με μια απλή σύσταση, τα κράτη-μέλη δεν θα κάνουν και πολλά. Ε, αρκεί να αγνοηθεί από ένα-δυο κράτη-μέλη και η Ευρώπη να παραμείνει ένα τρίπιο καλάθι όπως είναι αυτή τη στιγμή. Οπότε ε, παροτρύνω την Κομισιόν να, να ρίξει μια πιο ε, βαθιά ματιά στο πρόβλημα και να είναι λίγο πιο φιλόδοξη. Όπως πιστεύω ότι πρέπει να είναι. Ε, ξέρω ότι πολλά κράτη-μέλη θέλουν να κάνουν περισσότερα και ξέρω επίσης ότι πολλά κράτη-μέλη εξετάζουν την επικουρικότητα, τα κόστη κτλ. κτλ. Ε, κοιτώντας τη σελίδα 7 του οδικού χάρτη, ε, λέγεται την επιλογή 2, το κόστος αυτής της επιλογής θα ήταν περιορισμένο διότι δεν συνεπάγεται τη δημιουργία νέων υποχρεώσεων. Και αυτό μου δημιουργεί την εντύπωση ότι δεν θα φέρει και κανένα αποτέλεσμα. Όταν μιλάμε για περιορισμένο κόστος και μη δημιουργία νέων στόχων, νέων υποχρεώσεων ως βασικού στόχου, δεν πρόκειται λοιπόν ποτέ να ε, ανακόψουμε αυτό το κύμα της παρανομής εμπορίας ε, ειδών της αγριάς πανίδας. Ε, ξέρω ότι ε, πολλοί εύχομαι ε, ό,τι καλύτερο σε αυτή τη μάχη στην Κομισιόν ε, για τους επόμενους μήνες και στα κράτη-μέλη και θα ήθελα να μην ξεχνάτε ότι έχουν να γίνουν ακόμη πολλά. Ε, πρέπει να γίνουν πράγματα πιο επισταμένα γι' αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Εκ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε και την Επιτροπή βεβαίως την ευχαριστώ για, τις, για την παρουσίασή της. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι και άλλοι παράγοντες πέραν του οργανωμένου κλίματος επιδεινώνουν διαρκώς τη βιοπικιλότητά μας και πρέπει να έχουμε υπόψη ότι άπαξ και εξαφανιστεί ένα είδος δεν υπάρχει κανένα ποσό στον κόσμο που να μπορεί να το φέρει πίσω. Γίνεται πιο φτωχό ο κόσμο λοιπόν και οι μελλοντικέ γενναίε χάνουν ένα κομμάτι από τη φύση. Θα έπρεπε κανονικά όταν γεννιόμαστε και όταν πεθαίνουμε να αφήνουμε τον κόσμο όπως ακριβώς τον βρήκαμε. Άρα Πρέπει να είμαστε όλο και πιο φιλόδοξοι απέναντι στο οργανωμένο έγκλημα που κάνει αυτά τα εγκλήματα και να ορίζουμε όλο και πιο σαφείς στόχους. Και στους στόχους αυτούς θα πρέπει να μας απασχολήσει και το εάν ε, παραδείγματι υπάρχει δυνατότητα να απαγορευθεί η ε, η διατήρηση καλύτερα ζώων ως οικιακών εξωτικών που κινδυνεύουν με, απαγω... με εξαφάνιση. Πρέπει να υπάρχει αυτό. Πρέπει να υπάρξει επίσης η απαγόρευση των, ε, της διατήρησης τροφέων, ε, τροπέων από το θύραμα κάθε τύπου και κάθε είδους. Γιατί εάν τώρα δεν καταπολεμηθεί αυτή η διεθνής εγκληματικότητα και βέβαια το κυνήγι για να πάρει κανείς στο σπίτι του ένα τρόπεο, ε, κινδυνεύουν πολλά άλλα ήδη από εξαφάνιση. Αυτά και παρακαλώ να τα περιλάβετε στο έγγραφό σας. Ευχαριστώ κύριε Μακκίνες. Πρόεδρε ευχαριστώ και πολύ σύντομα δύο παρατηρήσεις. Βεβαίω το έγκλημα το σχετικό με την άγρια φύση είναι γενικώ σχετικό με το οργανωμένο έγκλημα. Και πρέπει να πιέσει η Επιτροπή περισσότερο ακόμη, αλλά πρέπει και τα κράτη-μέλη να συνεργαστούν μαζί μας για να φέρουμε αποτελέσματα και βέβαια ορισμένα κράτη ίσως χρειαστούν ειδικέ μονάδες στις αστυνομικές τους ε, αρχές προκειμένου να έχουν εξειδικευμένο προσωπικό για την καταπολέμηση αυτού του τύπου εγκλήματος και εμπορίου. Ευχαριστώ κυρία Μπέρνταρ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ και την Επιτροπή που μας έκανε τις προτάσεις αυτές. Είχαμε ιδρύσει μάλιστα από πέρσι μια διακομματική επιτροπή ευρωβουλευτών υπέρ της άγριας φύσης των οποίων κάποιοι άλλοι συνάδελφοι ναι, εδώ μέσα. Και θέλαμε ένα πρόγραμμα δράσης, διότι υπάρχει πολύ μεγάλο η εγκληματικότητα σχετική με την άγρια φύση, ανεξέλεγκτα δρούν αυτές οι οργανώσεις. Εμείς έχουμε κάνει συνεδριάσεις εδώ στην διακομματική αυτή επιτροπή ε, για το λαθρεμπόριο εις βάρος των ε, ειδών της άγρας φύσης, αλλά όχι μόνο αυτό και εμπόριο οικιακών ε, ζώων συντροφιάς καλύτερα. Βεβαίω υποστηρίζουμε από τις ε, προτάσεις που έχετε καταθέσει δύο στην τρίτη επιλογή, γιατί πιστεύουμε ότι αυτός είναι ο τρόπος να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το λαθρεμπόριο με είδη προερχόμενα από την άγρια φύση. Νομίζω ότι πάνω απ' όλα και περισσότερο από την πρώτη τη δεύτερη επιλογή ε, έχει η τρίτη τη δυνατότητα γιατί μπορεί να φέρει νομοθετήματα και χωρίς βέβαια να θέλουμε να νομοθετούμε για το καθετή η νομοθεσία νομίζω μπορεί να φέρει καλύτερα αποτελέσματα η νομοθεσία μπορεί να φέρει καλύτερα αποτελέσματα και εφαρμογή, επιβολή δηλαδή των κανόνων Δυστυχώς το λαθρεμπόριο δεν, ε, στα ίδια άγρια φύσης δεν αναγνωρίζεται ως προτεραιότητα για τα κράτη-μέλη. Αν και θα όφυλα να το πράξουν αυτό, γιατί είναι η τρίτη σε μέγεθος, σε όγκο οικονομικό παράνομη δραστηριότητα στον κόσμο, με τεράστια οικονομικά ποσά, με τεράστιο ε, όγκο με τεράστιο κέρδος ε, και δεν μιλάω μόνο για τα τρόπια από άγρια ζώα ή το ελεφαντοστούν αλλά και το εμπόριο σε σχέση με ζώα συντροφιά. Που μπορεί όταν πάει κανείς να τα αγοράσει στο σχετικό κατάστημα pet shop στη γειτονιά του να φαίνονται απόλυτα νόμιμα, αλλά πολλές φορές έχουν εξευρεθεί και αφαιρεθεί από την φύση. Έχουμε επίσης ε, διάφορα θέματα να συζητήσουμε αυτή τη νέα στρατηγική για την ε, συντήρηση της φύσης στην Αφρική, και άλλα, για την προστασία μάλλον της φύσης στην Αφρική και άλλα ζητήματα για τα ζώα και τα φυτά που φαίνεται να απασχολούν μια εμπορευματική δραστηριότητα με συνέπειες καταστροφικές. Και αυτό αφορά και την Ευρώπη. MEPs λοιπόν for Wildlife, αυτή η διακομματική ομάδα, θέλει και πιέζει την Επιτροπή και θα την πιέσει να προωθήσει την τρίτη επιλογή της το ταχύτερο δυνατό. Νομοθεσία δηλαδή με προτάσεις για την κάλυψη των κενών όπου υπάρχουν και ξέρουμε πολύ καλά ότι οι εθελοντικοί στόχοι δεν φέρνουν αποτελέσματα. Γιατί το έχουμε δει πολλές φορές αυτό. Χρειάζονται σαφείς ε, ενιαίοι ορισμοί από τις 28 χώρες. Χρειάζεται ένα σχέδιο βεβαίως, αλλά και η νομοθεσία που θα το στηρίξει ώστε να λαμβάνεται δράση κατά εκείνων οι οποίοι προκειμένου να αποκομίσουν κέρδος καταστρέφουν την άγρια φύση. Ευχαριστούμε. Κύριε Δορδάνο τώρα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Δύο παρατηρήσεις θέλω να κάνω σε σχέση με το χάρτη πορεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πρόγραμμα δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της ε, λαθρεμπορίας ζών. Όσον αφορά την νομική πτυχή τα προβλήματα της μεταφοράς του νόμου και της ομοιόμορφης εφαρμογής στις χώρες μέλη. Προτείνεται η αναθεώρηση της σύσταση της Επιτροπής του 2007 που αναφέρεται στους κανόνες εμπορία ζώων ή ακόμα ενίσχυση των κυρώσεων για το λαθρεμπόριο. Όμως, δεδομένο των προθεσμιών εφαρμογής των νέων κειμένων και τήρησης της αναλογικότητας, αυτό αποτελεί τροχοπέδι στη δράση μας. Έπειτα η πολιτική πτυχή έχει ενδιαφέροντος αλλά και γνώσεων και πραγματογνωμοσύνης για το θέμα, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί μια πλατφόρμα για το λαθρεμπόριο αυτό. Η οικονομική προσέγγιση λοιπόν κατά της διαφθοράς που προτείνεται τελικά παραδέχεται ότι τα ήδη υπάρχοντα κείμενα έχουν αποτύχει. Ευχαριστούμε πολύ και τώρα θα δώσουμε πάλι το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να απαντήσει. Ευχαριστώ πολύ για τις παρεμβάσεις σας. Πρώτον, θέλω να επιβεβαιώσω ότι πράγματι αυτό που θα κάνουμε είναι ότι θα εκδώσουμε ανακοίνωση με δράσεις. Το προσωπικό ετοιμάζει έγγραφο των υπηρεσιών μας με περισσότερες πληροφορίες για το εύρο στην κλίμακα των εγκλημάτων κατά της αγριάς πανίδας. Και μετά θα κάνουμε προτάσεις για νέα νομοθετικά κείμενα. Όμως, θέλω να υπογραμμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη ανακοινώσει στο θεματολόγιο της για την ασφάλεια ότι θα αναθεωρήσει ...στην τρέχουσα πολιτική και νομοθεσία όσον αφορά τα περιβαλλοντικά εγκλήματα το 2016. Περιλαμβάνεται εδώ και αναθεώρηση της οδηγίας για τα εγκλήματα κατά της άγριας πανίδας του 2009 που περιλαμβάνει το λαθρεμπόριο ζών και εξετάζει και το θέμα των κυρώσεων. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να μην μεν προκαταλάβουμε τα όσα θα αναφέρει, αλλά τη δράση που αναφέρεται. Πολύ σωστά τονίζεται τη σημασία που έχει η εφαρμογή. Και γι' αυτό πιστεύουμε ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε πιο στρατηγικά τη δράση μας. Πρέπει να βελτιώσουμε το συντονισμό μεταξύ των χωρών μελών και μερικές φορές μέσα στην ίδια χώρα μέλος. Πρέπει να υπάρχει περισσότερη συνεργασία με την Europol και την Eurojust που είναι δύο συντονιστικά σώματα για τις έρευνες που έχουν να κάνουν με διασυνοριακά ε, εγκλήματα και παραβιάσεις. Αναφερθήκατε στη γνώση και στην πραγματογνωμοσύνη που διαθέτουν οι χώρες μέλη. Όντως, αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Και βέβαια χρειάζεται περισσότερη συνειδητοποίηση και δυνατότητες διερεύνησης εγκλημάτων κατά της άγριας πανίδας. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και την εγκληματικότητα online και την νομοποίηση παράνομου χρήματος. Χρειάζονται συγκεκριμένες ιδέες προκειμένου να προχωρήσουμε γρήγορα για καλύτερη εφαρμογή με τα μέσα που έχουμε ήδη στη διάθεσή μας και με τη δική σας στήριξη. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πιστεύω ότι μπορούμε να κλείσουμε για σήμερα τη συνέντησή μας. Απλά να υπενθυμίσω στα μέλη και στο προσωπικό ότι το χριστουγεννιάτικο μας κοκτέιλ θα λάβει χώρα στο εστιατόριο του κτηρίου Γιάννη στον τρίτο όροφο. Ευχαριστώ.